Αγαπητοί συνάδελφοι, καλησπέρα σας και καλωσορίσατε ορίσατε στη συνεδρίαση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Καταρχάς έχουμε την έγκριση της σημερινής διάταξης, εγκρίνεται. Ευχαριστώ. Μια ανακοίνωση έχω του Πρόεδρου. Θυμίζουμε στα μέλη ότι εκπρόσωποι των Εθνικών Κοινοβουλίων θα έρθουν στην Επιτροπή μας αύριο το απόγευμα 9 Οκτωβρίου στις 2.30 με 4.30 πριν τις ψηφοφορίες για να συζητήσουμε τις διαρθωτικές μεταρρυθμίσεις και τα δημοσιονομικά που θα εφαρμοστούν στις διάφορες χώρες. Ε, και από ε, αύριο το πρωί θα αλλάξει και η διάταξη των εδράνων, δηλαδή να μην εκπλαγείτε αν έρθετε και δεν είναι η θέση σας εκεί που συνήθως κάθεστε. Είναι επειδή θα έχουμε εθνικούς βουλευτές. Ε, ανημέρω σχετικά με τις τρέχουσες διοργανικές διαπραγματεύσεις στις 2 Οκτωβρίου είχαμε τον τέταρτο ε, τριμερή διάλογο για την οδηγία για τις ε, κεφαλαϊκές ε, απαιτήσεις 5, τα διάφορα σχετικά θέματα, καταπολέμηση του ξεπλήματος και μεγάλη έκθεση μεταξύ άλλων. Έγινε ε, πρόοδος, επιτεύχθη μια συμφωνία και θέλω να ευχαριστήσω και τον κύριο Ερία γιατί ε, συζητήθηκε και μια διάλεξη που είχε κάνει για την καταπολέμηση του ξεπλήματος ε, βρώμικου χρήματος, ε, εσόδων από παράνομες δραστηριότητε, νομιμοποίηση. Και τελειώσαν οι ανακοινώσεις και προχωρούμε στην ημερησία διάταξη. Καλασορίζω τους τρεις φίλους προέδρους των τριών υποπτικών αρχών, Στίβεν Μαγιόρ, Ανδρέα Ερία και Γκαμπριέλ Μπερναρντίνου. Καλώς ορίσατε. Θα μας κάνετε μια παρουσίαση για τα πεπραγμένα και τις εμπειρίες σας στο περασμένο έτος, στο συντονισμό κυρίως και τη συνεργασία με τους νομοθέτες. Θέλουμε να ακούσουμε, ενδιαφερόμαστε για τις προτεραιότητες των οργανισμών σας για το επόμενο δωδεκάμινο. Ο κύριος Μαγιόρ θα μας μιλήσει και ε, ως ε, ε, πρόεδρος Μικτής Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών και ως δεύτερος αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου, όπως προβλέπεται από τον αντίστοιχο κανονισμό. Έχουν στείλει γραπτές δηλώσεις και οι τρεις πρόεδροι για τα πεπραγμένα των οργανισμών τους, των αρχών τους, το περασμένο έτος. Έχουν διανεμηθεί αυτά στα μέλη και υπάρχουν και στην ηλεκτρονική μας σελίδα θα κάνουν κάποιες αγωγικές παρατηρήσεις, ε, τοποθετήσεις. Ο κύριος Μαϊόρ θα έχει 10 λεπτά στη διάθεσή του γιατί ε, θα μας μιλήσει από πολλές ιδιότητες και μετά ο κύριος Ερία και ο κύριος Μπερναρντίνο ε, θα έχουν 5 λεπτά έκαστος. Και θα ακολουθήσει η κανονική διαδικασία ερώτα απαντήσεων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το έργο σας καταρχήν και καταρχάς και για την εξαιρετική εργαστή συνεργασία που έχουμε. Θα ήθελα επίσης να εκφράσω τη βαθιά μας προσήλωση και δέσμευση και στη δημοσιονομική διαδικασία αλλά και σε κάτι πιο σημαντικό που είναι η θεώρηση. Βέβαια και ο προπολογισμός είναι σημαντικό στοιχείο. Εκτιμώ πολύ επίση το έργο σα και στα πλαίσια ε, των συζητήσεων για το Brexit. Και προβλέπουμε και ελπίζουμε σε μια συμφωνία, ε, ώστε να πέσουν κάπω οι τόνοι. Είναι πολύ καλή πάντως η προετοιμασία στους οργανισμού σας. So, having said that, Τούτων ολολεχθέντων σας δίνω μέσω στο λόγο κύριε Μαγιόρ. Ευχαριστώ πολύ, Ρομπέρτο για τα φιλικά σου λόγια αυτά και τα θετικά σου σχόλια, για τη συνεργασία ε, με την Επιτροπή σας και από τις τρεις εποπτικές αρχές και οι τρεις πρόεδροι συνεργαζόμαστε πολύ καλά να σας δώσω πρώτα τη σύνοψη της Μικτής Επιτροπής και μετά θα περάσω στην ΕΣΜΑ, την Αρχή Κινητών Αξιών. ότι με πρόεδρε και μέλη του Κοινοβουλίου. Με χαρά σας μιλώ σήμερα εδώ υπό το ρόλο μου του Προέδρου της Μικτής Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών για το 2018. Θα αρχίσω με τα σημαντικότερα νομοθετικά θέματα διακλαδικά που ετέθηκαν σε ίσχυ φέτος. Ο κανονισμός PRIPS, από τότε που τέθηκε σε ισχύ, οι τρεις εποπτικές αρχές έχουν συνεργαστεί με τους ενδιαφερμένους έτσι ώστε γρήγορα να τεθεί σε ισχύ και ομαλά ο νέος κανονισμός. Προς το σκοπό αυτό έχουμε δημοσιεύσει ερωτήσεις και απαντήσεις για διάφορα θέματα έτσι ώστε να διευκρινίσουμε την εφαρμογή των κανόνων και να δώσουμε κοινέ πρακτικές εποπτείας αλλά και εφαρμογής ε, των ε, και του εγγράφου βασικών πληροφοριών, το KIT. Βεβαίως, ε, όταν είναι τόσο ευρία νέα νομοθεσία, ε, συνήθως ε, γνωρίζει κάποιες παιδικές ασθένειες. Αναγνωρίζουν υποπτικές αρχές τα θέματα με βάση τις εθνικές αρμόδιες αρχές και τους ενδιαφερόμενους που μας τα διαβίβασαν. Τα εξετάζουμε και προσπαθούμε να βρούμε κατάλληλες λύσεις. Για παράδειγμα, τον Ιούλιο καλέσαμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσει δημόσια καθοδήγηση για ποιο είδος προϊόντων και ιδιαίτερα ομολόγων καλύπτει αυτό αυτός ο κανονισμός στο πεδίο εφαρμογή τους. Επίσης αξιολογούμε ε, τα στοιχεία που μας δίνουν για τα διάφορα σενάρια επιδόσεων ε, και τις ε, αποδόσεις. Επειδή άργησε να εφαρμοστεί ο κανονισμός πριν σε ένα χρόνο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας ενημέρωσε ότι η αναθεώρηση θα αναβληθεί και αυτή χωρίς νομοθετικές αλλαγές από τον Ιανουάριο του 2020 οι ε, χρήστες σέκα ε, οι διαχειριστές θα πρέπει να ε, δίνουν βασικά έγγραφα πληροφοριών και τα usage και για τα prints. Αυτά εξηγήθηκαν από τις δικές μας εποπτικές αρχές προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα πρέπει να ληφθούν μέτρα και να γίνουν κινήσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να αποφύγουμε επικαλύψεις. Επίσης, η αναθεώρηση θα πρέπει να γίνει το συντομότερο σε ό,τι αφορά το έγγραφο βασικών πληροφοριών, έτσι ώστε οι συνομοθέτε να δούμε πώ χρειάζονται νομοθετικέ τροποποιήσει πριν το τέλο τη ε, τρέχουσα νομοθετική θητεία. Ε, άλλο σημαντικό στοιχείο για τη Μεκτή Επιτροπή το 2018 ήταν ε, η καταπολέμηση τη τρομοκρατία και του ξεπλήματο χρήματο. είδαμε πολλέ περιπτώσει όπου οι τράπεζες ε, δεν κατάφεραν να αποτρέψουν το οικονομικό ε, έγκλημα και πολλές φορές ήταν ε, τεράστιο αυτό το πρόβλημα. Το σημερινό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην αντίστοιχη νομοθεσία δηλαδή, μπορεί να μην αρκεί για την καταπολέμηση τρομοκρατίας και τη χρηματοδότησή της και το ξέπλυμα. Θα πρέπει αυτό να αναθεωρηθεί έτσι ώστε το ευρωπαϊκό σύστημα να μπορεί να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Βράχει πρόθεσμα, έκανε μια πρόταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το περασμένο μήνα και είναι καλά βήματα, πρώτα βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση για να συγκλίνουν οι αποπτικές προδιαγραφές και η εποπτεία όλων αυτών να γίνει πιο αποτελεσματική. Θεωρούμε ότι είναι σωστό η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή να παίξει σημαντικό ρόλο εδώ. Σε επίπεδο μεικτής επιτροπής ε, ασχολούμαστε με την ε, ε, εποπτεία της καταπολέμησης χρωματοδότησης τρομοκρατίας και του ξεπλήματος για να δούμε ποια είναι τα νέα στοιχεία, οι νέοι κίνδυνοι αναδιώνομοι και πώς μπορούμε με νέες κατευθυντήριες γραμμές να προχωρήσουμε και έχουμε μια συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για τα πρακτικά της ανταλλαγής προφοριών. Φέτος, η Μικτή Επιτροπή ε, συνέχισε το βασικό ρόλο της ελέγχου και εκτίμησης ε, διακλαδικών κινδύνων και ρίσκων. Σε βάθος έχουμε αναλύσει τις αναδυόμενες περιπτώσεις κινδύνου και καταφέραμε να εντοπίσουμε τους βασικούς κινδύνους ε, που αφορούν την εποπτεία. Έχουμε και μια αντίστοιχη έκθεση εξαμηνιαία. Και φέτος τονίσαμε και στις δύο εκθέσεις μας ε, τα προβλήματα και τις αβεβαιότητες που προκύπτουν από τον Brexit. Η Μεκτή Επιτροπή και πάλι εργάζεται πάρα πολύ ε, δραστήρια για την προστασία των Ευρωπαίων καταναλωτών και επενδυτών και για τον έλεγχο όλων αυτό. Η Μεκτή Επιτροπή μας ε, επέτρεψε σε μια ε, ημέρα, ημερίδα που κάναμε να έχουμε επαφές με τους ενδιαφερομένους. Ε, τονίσαμε ότι οι εποπτικές αρχές ενδιαφέρονται να υπάρχει διαφάνεια και ενημέρωση των καταναλωτών. Και θα εκδώσουμε την πρώτη επανάληψη μια σειρά εκθέσεων που θα βοηθήσουν τους καταναλωτές να λαμβάνουν αποφάσεις με τα λόγου και να συγκρίνουν αποτελεσματικά τα προϊόντα. Κυρίες και κύριοι, τώρα θα πρέπει εδώ να τελειώσω για τη Μεκτή Επιτροπή. Υπάρχουν θέματα όπως είναι το PRIPS, το Brexit, ε, το ξέπλυμα ε, του χρήματος και όλα αυτά θα συνεχίσουμε τα βρίσκουμε μπροστά μας και του χρόνου και τις επόμενες χρονιές. Και πάντα θα επικεντρωνόμαστε στην αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων. Έρχομαι τώρα ε, στη δήλωση που αφορά την ΕΣΜΑ το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου και θέλω να αφαιρθώ στο MIFID 2, ε, ε, στο CMU και τέλος στο Brexit. Αρχίζω με το MIFID 2. Ξεκινώντας με το Brexit, θα θυμάστε πολύ ότι τέτοιο καιρό πέρσι με ρωτούσατε για το εάν γινόταν σωστά η εφαρμογή και αν αναμέναμε κάποιες καθυστερήσεις. Σήμερα είμαι σε μια πολύ πιο καλή θέση για να απαντήσω σε αυτήν την ερώτηση, καθώς έχουμε την ημερομηνία έναρξης ε, που ήταν βεβαίως τον Ιανουάριο του 2018 και η οδηγία MIFID 2 πήγε πολύ πιο ομαλά από όσο φοβόντουσαν μερικοί, οπότε χαίρομαι που μπορώ να πω ότι υπάρχει γενικότερα πρόοδος. Πρώτα απ' όλα, για τα μέτρα εκείνα τα οποία αφορούν τα εργαλεία σύγκλησης, στόχο έχουν να διευκολύνουν την έγκαιρη και εναρμονισμένη εφαρμογή των κανόνων σε όλες ε, τις χώρες μέλη. Ένα σημαντικό κομμάτι του ερωτηματολογίου της MIFID 2 είναι αποτέλεσμα των ε, ερωτήσεων και ε, για διευκρινήσεις που έχουμε λάβει είτε από τα κράτη-μέλη είτε μέσω των αρμοδίων αρχών. Και αυτό ακριβώς αποδεικνύει την σημασία της ρυθμιστικής σύγκλησης για ολόκληρο το ρυθμιστικό πλαίσιο. Επιπλέον, η οδηγία MIFID 2 έχει δώσει νέα προοπτική στην χρήση των λεγόμενων γνωμοδοτήσεων της ΕΣΜΑ. Τους τελευταίους 12 μήνες η ΕΣΜΑ εξέδωσε γύρω στις 400 γνωμοδοτήσεις προς τις αρμόδιες αρχές ε, και όσον αφορά τα waiver ε, διαφάνειας και <clears throat> για άλλα ζητήματα και έχουμε όλες αυτές τις νομοδοτήσεις για τον πολυτεχνικό τομέα των δευτερογενών αγορών και θεωρούμε ακριβώς ε, ότι μπορούμε να εκδίδουμε αυτές τις γνωμοδοτήσεις και για ζητήματα outsourcing. Τώρα για να έρθω στα δεδομένα και τις ανάλογες λύσεις πληροφορικής εδώ πέρα Χαίρομαι για το ότι όλε οι αρμόδιε αρχέ αποφάσισαν να αναθέσουν κάποια παραδοτέα στο ευρωπαϊκό επίπεδο και να συνεργαστούν στενά με το προσωπικό τη ΕΣΜΑ για να, συλλέξουν, να οικοδομήσουν έξι νέα συστήματα δεδομένων και να συλλέξουν πληροφορίε για χιλιάδε συναλλαγέ ανά την Ευρωπαϊκή Ένωση. όπω ίσω ξέρετε είχαμε κάποιε αρχικέ καθυστερήσει όμω, δεδομένη της κλίμακα των απαιτούμενων προσπαθειών θεωρώ ότι έχουμε κάνει μια καλή αρχή τέλο η εφαρμογή του πακέτου MIFID-MIFIR σημαίνει πως είχαμε κάποια προβλήματα στην εισαγωγή του νέου πακέτου για την ΕΣΜΑ. Αυτό ήταν μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη για τους ε, μικροεπενδυτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση που αντιμετώπισαν διάφορα προβλήματα στις διαφορές των συμβάσεων μεταξύ κρατών μελών. Με τις νέες μας αρμοδιότητες την άνοιξη οθετήσαμε κάποια μέτρα που απαγόρευαν τις διαδικές επιλογές ε, και την, ε, και την πώληση των CFTs και άλλα βελτιώθηκε άμεσα η προστασία των επενδυτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να στραφώ τώρα στην ε, διαδικασία του σημειού που έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ στις εντολές του επίπεδου 2 όσον αφορά τους κανονισμούς τυκλοποίησης και στις δύο περιπτώσεις οι συνομοθέτες φρόντισαν να υπάρξει μια αρκετά μεγάλη περίοδος εφαρμογής κατά το οποίο βοήθησε τον σχεδιασμό και την εκτέλεση. Επιπλέον η ΕΣΜΑ εξακολουθεί να στηρίζει το έργο αυτό μέσω των διαφόρων δραστηριοτήτων ρυθμιστικής σύγκλησης, κάτι το οποίο περιλάμβανε εξετάσεις από ομοτήμους και ένα διατομεακό σχέδιο το οποίο ανέφερα και προηγουμένως. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να διατηρηθεί αυτή η όρμη καθώς Έχουμε μια όλο και μεγαλύτερη σύγκληση η οποία απαιτεί και την συμμετοχή των λιανικών επενδυτών. Στο πλαίσιο αυτό εκτιμώ την ε, πρόταση της ε, ΕΣΜΕ η οποία θα πρέπει να υιοθετηθεί σε αυτήν την ε, θητεία. Θα πρέπει λοιπόν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να προχωρήσουν αμέσως στην υιοθέτησή τη Αντιλαμβάνομαι βεβαίω ότι οι νομοθετικέ αυτές προτάσεις είναι φιλόδοξες και η αντίθεση από κάποιους ε, είναι αναπάντεχα ισχυρή. Το βλέπω ως αντίφαση, δηλαδή να υποστορίζουμε την Ένωση των Κεφάλαια Αγορών αφενός και από την άλλη να είμαστε κατά των προτάσεων που περιλαμβάνει και κάποια βασικά στοιχεία σύγκλησης ε, και μετακίνησης κάποιων αρμοδιοτήτων εποπτεία στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Τώρα θα αναφερθώ στο Brexit. Μετά τις τέσσερις συγνωμοδοτήσεις του 2017 για τις δραστηριότητες με τον κατάσταση στις 27 χώρες ε, συνεχίσαμε να βλέπουμε αυτό το ζήτημα με τις αρμόδιες αρχές στο πλαίσιο του συντονιστικού δικτύου εποπτικών αρχών και επιπλέον ως η εποπτική αρχή των αποθετηρίων συνεχίσαμε να κάνουμε ένα σχεδιασμό εκτάκτου ανάγκης παρακολουθούμε προσεκτικά την εκτέλεση των ε, σχεδίων αυτών ε, έτσι ώστε να πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις 27 χώρα στην περίπτωση που το Μάρτιο του 2019 δεν έχουμε κάποια συμφωνία. Επειδή πλησιάζει σύντομα αυτή η προθεσμία συνεχίζουμε να εστιάσουμε στις ε, διάφορες κατηγορίες ρίσκου στην περίπτωση που έχουμε ένα Brexit χωρίς συμφωνία. Θα ήθελα λοιπόν να σας ευχαριστήσω για την συνεχιζόμενη στήριξή σας και παραμένω στην διάθεσή σας για ερωτήσεις ε, σήμερα το απόγευμα, αλλά και όποτε εσείς το θέλετε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πληρέστατη παρουσίαση. Ανδρέα Βία, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ο Ρομπέρτο, μακρά η διαδικασία για αποκατάσταση των συζυγίων των Ευρωπαϊκών Τραπεζών. Πετύχαμε πρόοδο πέρσι σταθεροποιήθηκαν περίπου στο 14,5% τα δέοντα ποσοστά στο δεύτερο εξάμεινο του 2017 και αυτά τα υψηλότερα επίπεδα σύγκληση υποστηρίζουν την ανάπτυξη σε πολλού τομεί και για διάφορα αξιόγραφα που αντιμετωπίζουν κινδύνου. Υπάρχουν σε πολιτικών δράσεων. Συμφωνήθηκαν στο Συμβούλιο για τα κόκκινα δάνεια. Επιταχύναμε με τα μέτρα όσον αφορά την εκαθάριση των συζυγίων των τραπεζών. Κατά 250 δις είχαμε μείωση των κόκκινων δανείων τελευταία χρόνια και έτσι είμαστε στο αναγκαίο ποσοστό 3,6%. Θα πρέπει οι πρωτικέ αρχέ να ασκήσουν πιέσει για να τηρηθεί και να επιταχυνθεί η ιδέουσα προσαρμογή, εκμεταλλευόμενη τα, θετική η μακροοικονομική πρόβλεψη. Η ολοκλήρωση τη μειώσεω των κινδύνων και το σχετικό πακέτο θα οδηγήσει στην ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων μετά την κρίση και περιμένουμε διάφορε εντολέ που θα δοθούν στην αρμόδια αρχή. Σα έστειλα κάποια σημεία όσον αφορά την ταχεία εφαρμογή των κατατέλειων μέτρων το κατάλληλο πλαίσιο για εποπτικές αρχές που θα υποβάλουν και τις εκθέσεις. Υποστηρίζουμε και την πρόταση σχετική του Κοινοβουλίου και κάποιες ανησυχίες εκφράζουμε σχετικά αφορά τον ορισμό των διαφόρων στοιχείων. Υπάρχει μια ανάγκη να εστιάσουμε τις προσπάθειές μας από νομοθεσία πρωτογενή σε εποπτικές πρακτικές για να καταπολεμήσουμε τον κατακαιρματισμό στις τραπεζικές αγορές της Ευρωπαϊκής Ενώσης και να προωθήσουμε το διαμερισμό του κινδύνου στον ειδικό τομέα. Ετοιμάζουμε ένα έγγραφο για τα ρυθμιστικά εμπόδια όσον αφορά τη συνεργειακή σταθεροποίηση, όσον αφορά τα, τα προβλήματα του παρελθόντος και την αποκατάσταση των τραπεζικών εργών, έχουμε δύο προκλήσεις για την ενιαία αγορά και την Τραπεζική Ένωση υπαρξιακής φύσεως. Και θα αποτύχει η Ευρωπαϊκή Ένωση αν η επόμενη κρίση τελικά μας βρει να πολεμούμε τα δύο παλαιά μέτωπα. Του επόμενου μήνε μέγιστη προτεραιότητα για μα, θα είναι να βρούμε ανταπόκριση στην πρώτη της Ευρωπαϊκής στην εφαρμογή του τελικού πακέτου τη Βασιλεία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήδη ξεκινήσαμε συλλογή στοιχείων. Έχουμε βρει δειγματολόγια τραπεζών Θέλουμε να δούμε τα νέα διεθνή πρότυπα τι αντίκτυπο θα έχουν και προτείνουμε αναλογικό τρόπο για να εφαρμόσουμε τα πρότυπα στο νομικό μα πλαίσιο. Παρατηρώ ότι κάποιε προτάσει για το πακέτο εκδιώσεω του κινδύνου συνεπάγονται εμπροστοβαρή στοιχεία τη νέα συμφωνία ασυλία, προδικάζοντα την ανάλυση μα. Η έκθεσή μα πρέπει να είναι έτοιμη μέχρι τον Ιούνιο του 2019. Θα είναι σημαντικό να περιμένουμε πρώτα και τα αποτελέσματα, ώστε η απόφαση να ληφθεί εμπεριστατωμένα για να πετύχουμε τα πλήρη ωφέλη των μέτρων αποφασιστική δράση απαιτείται. Θέλουμε περιχειρησικό σύστημα εξυγίανση, σταθερή πρόοδο, συμμόρφωση με τι απαιτήσει MRL, συμφωνία για κρίσιμες λειτουργίε και ένα πιο εναρμονισμένο πλαίσιο για τις κοινοφελείς υπηρεσίες και διευθυντήσει για την ρευστοποίηση των τραπεζών. Αυτό μαζί με την πρόοδο όσον αφορά το σχήμα ασφαλή των καταθέσεων είναι βασικά για να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη μεταξύ αρχών που είναι κάτι πολύ σημαντικό για την λειτουργία μια ολοκληρωμένη τραπεζική αγορά οι σοβαρέ παραβιάσει ε, τη νομοθεσία για την καταπολέμηση ξεπλήματο χρήματο και την καταπολέμηση τη νομοκρατία χρειάζονται μια απάντηση σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Και πέρα από τι εργασίε τη Κοινή Επιτροπή που αναφέρθηκαν, οι εποπτικέ αρχέ ξεκίνησαν ένα σχέδιο πλήρε για να θεωρήσουν την αποτελεσματικότητα των εποπτικών αρχών για θέματα καταπολέμηση ξεπλήματο χρήματο. Και θα γίνει μια συνάντηση των αρμοδίων και θα εξετάσουν τα θέματα και διάφορα διαθέσιμα εργαλεία. Στόχο να εντοπίσουμε βέλτιστε πρακτικέ και να δώσουμε τροφοδότη αρμόδιε αρχέ, ούτω ώστε να ενισχύσουμε τι εποπτικέ προσεγγίσει. Αλλά για πραγματικά να συμβάλλουμε σε αποτελεσματικότερη καταπολέμηση του φαινομένου του ξεπλήματο χρήματο επίπεδο Ευρωπαϊκή Ενώση, χρειαζόμαστε περισσότερου πόρου και σαφήνεια όσον αφορά τι εξουσίε που θα έχουν οι, οι ευρωπαϊκέ αρχέ. Οι τραπεζικέ αρχέ. Λοιπόν, πρέπει να επεξεργαστούμε διάφορα μέτρα και ολοκληρώνουμε τι εργασίε για τα πρότυπα που μα ανέθεσε η νομοθεσία και προσπαθούμε να εξετάσουμε τι γίνεται με τη σύγκληση την εποπτική στα, στο νέο πλαίσιο. Και το θέμα νέων υπηρεσιών, όσον αφορά τι πληρωμέ, ε, είναι κάτι που αλλάζει την τραπεζική αγορά. Ξεκινήσαμε μια γενική συζήτηση για το θέμα αυτό, για το FinTech και ξεκινήσαμε μια, έναν κατάρτιση οδικού χάρτη και συλλογή γνώσεων. Αφού εξετάσαμε κινδύνους και ευκαιρίες από fintech και προβλήματα για τις ε, τράπεζες και τα σχετικά μοντέλα, θα εξετάσουμε τι γίνονται τα καθεστώτα διοδότησης, προσέγγισης, τα ρυθμιστικά μέτρα και τα κέντρα καινοτομίας. Θα ήθελα επίση να πω ότι αυξάνεται η χρήση ε, των εργαλείων δημοσιολόγηση και παβίση χρόνου στον τομέα καταπολεμήσεω ξεπλήματο χρήματο. Πολύ θετικά τα αποτελέσματα. Πιστεύω όμω ότι η εργαλειοθήκη μα για αναθεώρηση και αλλαγή των εποπτικών πρακτικών των εθνικών αρχών δεν είναι κάτι που είναι παρκές. Εξέταση ομοτήμων πολύ σπάνια αμφισβητεί τι πρακτικέ, η παραβίαση ε, του, νο, της νομοθεσίας δεν είναι σωστή προσέγγιση. Ανεξάρτητα ανεξάρτητοι έλεγχοι θα μπορούσαν να ενισχύσουν την εποπτική σύγκληση, κυρίως αν μπουν σε ένα σύστημα διακυβέρνηση πιο ουδέτερο. Με απογοήτευση βλέπω ότι οι προτάσει Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι σχετικέ, δεν την χάνουν ευρεία υποστήριξεω. Το Brexit είναι και θα παραμείνει για λίγο ύψιστη προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή. Θέλουμε να επιταχυθεί η προετοιμασία για περίπτωση μη συμφωνία και είναι σημαντικό να ξεκινήσουμε διαπραγματεύσει με του συναδέλφου του Ηνωμένου Βασιλείου γρήγορα διευθετήσει για υποπτική συνεργασία μετά το Brexit. Διότι σύντομα ίσω δοκιμαστούν αυτέ οι δυνατότητε αν δεν υπάρξει συμφωνία. Το Brexit ασκεί πολύ πιέσει στο φορέα μα και στο προσωπικό για προετοιμασία τη μετεκατάσταση στο Παρίσι. Καλά πάει η προετοιμασία, αλλά καθυστερήσει για την ολοκλήρωση τη νομοθεσία σχετική οδηγεί σε αναβολή όσον αφορά την υλοποίηση συμβάσεων. Όνο όταν τον Οκτώβριο θα υπάρξει συμφωνία μεταξύ των νομοθετών θα εξασφαλίσουμε μετακίνηση ε, στο Παρίσι τέλος Απριλίου του 2019. Πρέπει να πούμε ότι αυτές οι αβεβαιότητες επηρεάζουν πολύ το προσωπικό μας. Πρέπει να κάνουν προετοιμασίες για μια δύσκολη μετακόμιση. Πρέπει να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι με τις ε, οικογένειές τους. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, Ανδρέα. Ελπίζουμε θέμα της μετακόμισης να τελειώσει επιτέλους αυτός ο τριμερής διάλογος ε, χωρίς τέλος. Ε, υπάρχει το παράδειξο γιατί βεβαίως ε, υποτίθεται ότι πρέπει να είναι στην διαδικασία της συναπόφασης αλλά το Συμβούλιο δεν ήθελε να το δεχτεί γιατί είπε ότι είναι απόφαση του Συμβουλίου. Και έτσι είπαμε εντάξει τι να σας πω. Είναι λίγο παράδοξο λοιπόν. και ελπίζω τώρα να υπάρχει μια συμφωνία σε ένα κείμενο το οποίο θα οριστικοποιηθεί για να προετοιμάσει το έδαφος για μια αναθεώρηση της κοινή δήλωσης και να μην έχουμε τα ίδια προβλήματα στο μέλλον. Και βεβαίω ε, στόχο έχω να διασφαλίσουμε ότι αυτό θα γίνει το συντομότερο δυνατόν. Αλλά όπως ξέρετε είναι ένα φάκελο που αφορά πολλέ επιτροπές, οπότε δεν είναι 100% δική μα υπόθεση. Τούτου λεχθέντος ε, και με συγχωρείτε για αυτή την παρατήρηση, αλλά έπρεπε να γίνει. Λοιπόν, Γκάμπριελ, είναι η σειρά σα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και τους βουλευτές ε, της Επιτροπής σας. Πέρσι η αρχή μας ε, συνέχισε να εργάζεται σκληρά για να υπάρξει μια σωστή υποπτία του κλάδου των ασφαλιών και των συντάξεων ε, σε ολόκληρη την Ευρώπη. Έχουμε ένα ενιαίο βιβλίο κανόνων και στο πλαίσιο αυτό προτείναμε στην Κομισιόν περαιτέρω απλοποιήσεις και αναλογικά μέτρα για να μειωθεί το βάρος των μικρομεσαίων ασφαλιστικών εταιριών και να μην υπάρχουν περιορισμοί όσον αφορά τις επενδύσεις σε ακάλυπτα ομόλογα και μετοχές οι οποίες δεν είναι εισηγμένες. Τώρα προσπαθούμε ακριβώς να δούμε πώς θα περιλάβουμε τις ε, περιπτώσεις ε, της επένδυσης ε, στην βιώσιμη οικονομία. Στα εποπτικά ζητήματα προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση που θα προκύψει από ένα Brexit χωρίς συμφωνία. Έχουμε εκδώσει τέσσερις γνωμοδοτήσεις. Επίσης υπάρχει μια πλατφόρμα διασυνοριακής συνεργασίας για να υπάρχει μια καλύτερη συνεργασία μεταξύ των αρχών της χώρας προέλευσης και προορισμού της κάθε εταιρεία. Έχουμε συντονίσει 13 πλατφόρμες που περιλαμβάνουν τις εθνικές εποπτικές αρχές από πολλά κράτη-μέλη και έχουν αναλυφθεί διάφορες εποπτικές δράσεις. Τα επιχειρηματικά μοντέλα αυτών των εταιριών συνήθως στηρίζονται στην ανάπτυξη εκτός της οικίας αγοράς όπου ο κίνδυνο θα υλοποιηθεί μέσω μακροπρόθεσμα. Βρήκαμε κάποιες ελλείψεις στις τεχνικές διατάξεις, ασάφειες στις, ε, αξιώσεις και διάφορα προβλήματα όσον αφορά στις ε, αξιώσεις που αφορούν περίπλοκα προϊόντα αλλά και ιατρικέα λάθη. Μπορεί λοιπόν να περιπλακεί η κατάσταση και στις ε, οικίες αγορές και να υπάρχει μια δυσπιστία όσον αφορά τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Αυτό όμως δείχνει και τους περιορισμούς του υφιστάμενου πλαισίου. Γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό να χρησιμοποιήσουμε την αναθεώρηση του κανονισμού της ΕΙΟΠΑ για να έχουμε μια ενισχυμένη έντολη για τη ρυθμιστική σύγκληση. Θα αναφέρω λοιπόν τέσσερα σημεία. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να έχουμε την εντολή να κάνουμε ανεξάρτητες αξιολογήσεις των εθνικών ε, αρχών ε, και πρακτικών αξιολόγησης. Δεύτερον, όσον αφορά τις ε, διασυνοριακές συναλλαγές θα πρέπει να μας ενημερώνουν οι εθνικές αρχές για τις διασυνοριακές δραστηριότητες θα πρέπει να αναλάβουμε τη διατήρηση μιας βάσης δεδομένων για να υπάρχει μια διαφάνεια για τα διασυνοριακά προϊόντα και να έχουμε μια σαφή εντολή για να φτιάξουμε πλατφόρμες συνεργασίας και να δίνουμε κατευθυντήριε γραμμές στι εθνικές εποπτικέ αρχές. Οι πλατφόρμες θα πρέπει να χρησιμοποιούν ως ένα εργαλείο προληπτικό και όχι αντιμετώπισης κρίσεων. Τρίτον, θα πρέπει να έχουμε την δυνατότητα να κάνουμε ανώνυμες αγορές σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τέταρτον, για να υπάρχει η διαφάνεια στα stress test θα πρέπει να έχουμε την δυνατότητα να δημοσιεύουμε μεμονωμένα αποτελέσματα όπως γίνεται ήδη στον τραπεζικό τομέα. Καταλήγοντας λοιπόν θα ήθελα να αναφερθώ στις ε, τελευταίες εξελίξεις στην Ένωση Κεφαλαιαγορών και στο Πανευρωπαϊκό Συνταξιοδοτικό Προϊόν το λεγόμενο ΠΕΠ. Το ΠΕΠ αυτό θα είναι επιτυχία μόνο εάν το εμπιστευτούν οι Ευρωπαίοι πολίτες. Οι Ευρωπαίοι πολίτες χρειάζονται σαφείς πληροφορίες και να υπάρχει μια διασφάλιση ποιότητας και διαφάνειας. Ως Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή η ΕΙΟΠΑ μπορεί να διασφαλίσει αυτή την ε, ποιότητα και ομοιομορφία σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και οπωσδήποτε θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε να διασφαλίσουμε υψηλά επίπεδα προστασίας των καταναλωτών και σταθερότητα των αγορών. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Γκάμπριελ. Την Πέμπτη θα γίνει ο πρώτος τριμερής ε, διάλογος. Το Κοινοβούλιο ζήτησε να παίξει αυτό το ρόλο η ΑΕΟΠΑ και θα πολεμήσουμε για αποδοχή του κειμένου μας από το Συμβούλιο. Θα σπρώξουμε και τα άλλα θέματα βέβαια. Ήρθε η ώρα να πάμε στους ομιλητές. Για το ΕΛΚ, ο Μάρκους Φέρμπερα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα μιλήσω στη μητρική μου γλώσσα, τη γερμανική. Δεν θα πω τίποτα για το μύφιτ. Χαίρομαι και εγώ που πάνε καλά τα πράγματα. Έχω μια ερώτηση προς τον κύριο Ερία ε, της Ευρωπαϊκής Αρχής Τράπεζων. Τους τελευταίους μήνες είδαμε παραβιάσεις ε, του ξεπλήματος ε, χρήματος και της καταπολέμησης χρηματοδότησης της ε, τρομοκρατίας. Δεν έχετε αγγλικά διερμηνία Καλά, τα δικά μου αγγλικά δεν κάνουν όμω, Έχω και την ερώτηση στα γερμανικά γραμμένη και τη διαβάζω. Α, τώρα διατίθενται και τα αγγλικά μάλιστα. Μήπως και γαλλικά μπορώ να τα πω αλλιώ. But for our Irish colleagues, we should safeguard English. Όχι, για τους Ολλανδούς ε, συναδέλφους θα κρατήσουμε τα αγγλικά παρά το Brexit. Λοιπόν, τι έλεγα, ε, ε, ξέπλυμα χρήματος ε, και καταπολέμηση χρηματοδότησης τρομοκρατίας. Από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν λάβαμε μια πρόταση νομοθετική καινούρια που προβλέπει ότι η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών θα έχει νέες αρμοδιότητες. Αλλά είναι πολλές οι περιπτώσεις ξεπλήματος χρήματος. Και τι γίνεται με τις εθνικές εποπτικές αρχές. Κάνουν αρκετά. Ένα κατάφορο παράδειγμα είναι αυτό που έκανε η Μαλτεζική η ε, τράπεζα με την τράπεζα Πιλάτος που ξέπλανε και χρήματα εκτός από τα χέρια της. Ε, και ε, υπήρχαν διάφορες ατασταλίες και σε παρόχους υπηρεσιών και οικονομικό έγκλημα. Τίθεται λοιπόν το ερώτημα αν αρμόδιες υποπτικές αρχές ασχολήθηκαν με αυτό το θέμα, με τη Μαλτέζικη περίπτωση, ε, εκφράσατε σημαντικές επιφυλάξεις για τον τρόπο που λειτουργεί η εποπτεία των τραπεζών στη Μάλτα και παρόλα αυτά αποφασίσατε να μην αρχίσετε ε, μια διαδικασία προσφυγής επί παραλήψη, όπως προβλέπετε στο άρθρο 17 του βασικού κανονισμού λειτουργία της EBA δεδομένου και του ρόλου που θα έχετε στο μέλλον ως ε, υπαριθμόν ένα ε, ε, αρμόδιος για την καταπολέμηση αυτού του φαινομένου, γιατί δεν κινητοποίησατε το άρθρο 17 και στις άλλες αρχές υπάρχει περιθώριο ελιγμών για την καταπολέμηση του ξεπλήματος. Η ΟΠΑ και η ΕΣΜΑ θα πρέπει να έχουν σχετικές αρμοδιότητες, να αποκτήσουν δηλαδή αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Μου επιτρέπει να διαλύσω οι εσδήποτε παρεξηγήσεις. Είχαμε παρα... έρευνα η παραβίαση του δικαστικού του νόμου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Πιλάτος και αποφασίσαμε αυτή την παραβίαση και έγινε από την αρμόδια μονάδα η έρευνα. Έχει ληφθεί μια απόφαση στην περίπτωση της Μάλτας και εφαρμόζεται η απόφαση. Στέλνουμε και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την απάντηση των αρχών της Μάλτας για το θέμα του ελέγχου και θα δούμε κατά πόσο η απόκριση των Μαλτέζικων αρχών αρκεί ή θέλουμε να επιβληθούμε στις εθνικές αρχές. Δεν επιδιώκουμε παράβαση όσον αφορά την FSA της Άλματ. Διότι ο κανονισμός για τι ευθύνε του φορέα FSA δεν καθορίζεται επαρκώς στο ε, κείμενο με αναμφισβήτητο τρόπο που να πούμε ότι οι δυναμίες που εντυπώσαμε ε, αποτελούν παραβίαση του νόμου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Η διατύπωση οδηγίας του CRD4 δεν είναι σαφής και η ενσωμάτωση της οδηγίας στην νομοθεσία της Μάλτας να επιτρέπει να ακολουθήσουμε την αυτή την οδό. Στέλνοντας επιστολή στην FSA της Μάλτας, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στους Ευρωβουλευτές, εντοπίσαμε κάποια βήματα που πρέπει να λάβει η αρχή FSA της Μάλτας για να καλύψει τα κενά που εντοπίσαμε εμείς στην έρευνά μας. Θα δοθεί λοιπόν κάποια συνέχεια. Uh, uh, και κάποια σχόλια. Όπως είπα και στην αρχή υποστηρίζαμε ότι υπάρχει συγκέντρωση των διαφόρων φορέων και τι είδαμε ότι η EBA έχει αποκτήσει τη μέγιστη τεχνογνωσία και θέλουμε να αποφύγουμε κατακαιρματισμό των πόρων. Και τι γίνεται στην πράξη. Στις περισσότερες περιπτώσεις όταν υπάρχουν θέματα εξεπλήματος χρήματος στα αξιόγραφα γίνεται αυτό μέσω των τραπεζικών συστημήτων. Μιλάμε για διανομή χρηματοστικών προϊόντων και διανομή πόρων και αυτά γίνονται μέσω των δικτύων των τραπεζών για να διανεμηθούν αυτά τα προϊόντα. Υποστηρίζουμε κεντρική αντιμετώπιση του προβλήματος. Κάτι άλλο που μάθαμε. Οι αρχές, οι εποπτικές έχουν ελάχιστες δυνατότητες να δράσουν εκτιμώντας αν λειτουργούν σωστά εθνικές υποπτικές ε, πρακτικές. Όταν υπάρχουν προβλήματα να πάμε επί τόπου, ε, υπάρχουν, βλέπετε, όρια όσον αφορά τη χρηματοδότηση. Δύσκολο να πηγαίνουμε πάντα επί τόπου, να βλέπουμε τι γίνεται σε εθνικό επίπεδο. Τι έγινε εδώ. Στην περίπτωση του προβλήματο ξεπλήματο χρήματο, ίσω να υπάρχει και σε άλλα μέρη. Αλλά δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε σαν ευρωπαϊκέ εποπτικέ αρχέ. Επακριβώ. Ο Γκάμπριελ, πολύ σύντομα. Συμφωνώ με αυτά που είπε ο Στίβεν για τις εξουσίες. Καλό να υπάρχει κεντρική αντιμετώπιση. Κάτι άλλο για το ξέπλυμα χρήματος. Πρόβλημα συντονισμού υπάρχει και συνεργασίας μεταξύ των μονάδων συλλογή ε, πληροφοριών για οικονομικά θέματα και των εποπτικών αρχών. Σε περιπτώσεις διαμεσολάβησης είδαμε ότι υπάρχουν κάποια στοιχεία που εμφανίζονται για ξέπλυμα χρήματος, αλλά δύσκολο να κυκλοφορήσουν οι πληροφορίες μεταξύ των αρμοδίων εθνικών αρχών και των ποπτικών αρχών. Και αυτό δημιουργεί προβλήματα όσον αφορά την εφαρμογή των κανόνων. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το καλύψει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Συγγνώμη, συγγνώμη που δευτερολογώ. Για να σε ενημερώσω. Βλέπουμε τι έγινε με την περίπτωση της Μάλτας και το Πιλάτος. Κάναμε έρευνες. Επίσης και στη Λετωνία και την Τάπεζα ε, στην ε, Δανία. Όπως είπα και στην αρχή, εξετάζουμε το τι γίνεται στην εποπτεία στον αυτό το ξέπλυμα χρήματος όταν κάτι μελήξει. Στο τέλος του έτους θα έχουμε δύο κατευθυντήρες γραμμές και μία έκθεση και δύο άνθρωποι τα επεξεργάζονται αυτά. Θα αξιολογήσουμε το έργο μας. Νομίζω ότι πολλά πετύχαμε σε αυτούς τους τομείς και είμαι αρκετά ε, υπερήφανος για τα πεπραγμένα μας. Ευχαριστώ πολύ. Αν θυμάμαι σωστά, στην επιστολή σας είπατε ότι δεν ασχολούμαστε τόσο με το FCA λόγω της νομοθεσίας προτείνατε και βελτίωση του CRD για να είναι πιο ξεκάθαρες οι καταστάσεις. Θα το λάβουμε υπόψη και στον τριμερή διάλογο. Πολ Τάγκ, ευχαριστώ. Θέλω και εγώ να αναφερθώ στη σταθερότητα της χρηματοδότησης, κάτι που αναφέρατε. Έχουμε το σχέδιο δράσος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πολύ ευπρόσδεκτο από το Ευρωκοινοβούλιο. Είναι μια αλλαγή που τη χρειαζόμασταν από παλιά. Και έχει μείνει πίσω ο χρηματοπιστωτικό τομέα όσον αφορά τη βιωσιμότητα, εν τη ενία του ε, όρου. Εξετάζουμε τη βαθμολόγηση, ταξινόμηση ε, και τους διάφορους στόχους. Εξέφρασε σε έκθεση πρωτοβουλίας ότι ο ρόλο των εποπτικών αρχών είναι σημαντικότατο. Χρειαζόμαστε δεσμεύσει για αλλαγέ. προ βιώσιμο χρηματοπιστωτικό τομέα. Χρειαζόμαστε όμω επίση και ευελιξία στην υλοποίηση των μέτρων. Είναι θέμα υποχρεώσεων και Αυτό Αυτός συνδυασμό χρειάζεται. Οι εποπτικοί φορεί παίζουν σημαντικότατο ρόλο. Χρειάζεται και προώθηση των βέλτιστων πρακτικών. Πώς βλέπετε το ρόλο των τριών εποπτικών αρχών Πώς μπορείτε να συμβάλλετε και οι εποπτικές αρχές, οι ευρωπαϊκές, τι χρειάζονται για να παίξουν σωστά το ρόλο τους, το ρόλο που θέλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να διευκρινίσουμε την εντολή των εποπτικών αρχών και των εθνικών εποπτικών αρχών, να εξετάζονται διάφοροι κίνδυνοι και διάφοροι, παρα... παράγοντες, να έχουμε καλύτερη βιωσιμότητα των αγορών. Σε ένα σχέδιο εκθέσεως στις εντολές αναφέρεται ήδη η βιωσιμότητα, δίπλα σταθερότητα και αποτελεσματικότητα του χρηματοστικού συστήματος. Και οι οίκοι αξιολόγησης δεν συμπεριλαμβάνουν τη βιωσιμότητα και τους κινδύνους με τον ίδιο τρόπο στη μεθοδολογία όπως οι τράπεζες χρειαζόμαστε ελέγχους αντοχής τραπεζών και το ίδιο για τα συνταξιωτικά ταμεία ενδεχομένω. Αυτή είναι η γενική ερώτηση. Πώς βλέπετε το ρόλο σας και τι χρειάζεστε για να διαδραματίσετε αυτό το ρόλο. Ευχαριστώ πολύ που το θέσατε αυτό. Κοίταξε, από πλευρά ΕΣΜΑ, δύο είναι τα βασικά στοιχεία για τη βιωσιμότητα. Πρώτον, να εξασφαλίσουμε ότι στην παροχή πληροφοριών από τους εκδότες της εισηγμένες εταιρείε λαμβάνεται παρκώς υπόψη ο κίνδυνος, ο μακροπρόθεσμος κίνδυνος, η κίνδυνη από πλευράς βιωσιμότητας και κυρίως ο περιβαλλοντικός κίνδυνος. Να εξασφαλίζουμε ότι η βαθμολόγηση, η αξιολόγηση αντικατοπτρίζει σωστά τους μακροπρόθεσμους κινδύνους που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα. Κάτι άλλο. Η η ενημέρωση, εκθέσει για τα χρηματοστατικά, να, οι εκδότες να ενημερώνουν επαρκώς του επενδυτέ όσον αφορά του κινδύνου βιωσιμότητα. Από την άλλη πλευρά, αυξάνεται η ζήτηση από την κοινότητα των επενδυτών, λιανικών επενδυτών, θεσμικών επενδυτών, που θέλουν να επενδύσουν σκόπιμα σε βιώσιμε επενδύσει. Και γι' αυτό είναι σημαντική η ταξινόμηση, διότι τελικά θέλει να δώσει την ευκαιρία στου επενδυτέ που θέλουν πραγματικά να επενδύσουν σε βιώσιμε επενδύσει αυτοί να μπορούν να το κάνουν αυτό αξιόπιστα. Το σχέδιο δράσεως μας επηρεάζει ποικιλοτρόπως. Θα δούμε πώς η βιωσιμότητα και τα στοιχεία αυτής να συμπεριληφθούν σε χρηματοδοτικές συμβουλές που δίνουμε. Ένας πελάτης θέλει να επενδύσει σε βιώσιμη επένδυση. Πώς αυτό επηρεάζει τις συμβουλές που του δίνουμε και το στόχο που θα θέσουμε στην αγορά. Και άλλο θέμα, θέματα αν ή και αξιολόγηση λαμβάνουν επαρκώ υπόψη του μακροπρόθεσμου κινδύνου οι οποίοι σχετίζονται με τη βιωσιμότητα. Τελικό σχόλιο. Το ενδιαφέρον είναι ότι ο δημόσιο τομέα έχει μείνει πίσω και ο ιδιωτικό τομέα ηγείται. Προωθεί το ζήτημα και χρειάζεται ένα αξιόπιστο τρόπο βιώσιμε επενδύσει να διαχωριστούν από τι επενδύσει που δεν είναι βιώσιμε. Πολύ γρήγορα Υποστηρίζω το θέμα της αξινόμησης. Είναι βασικό στον τομέα μας. Ο ρόλος πρασίνων διοντολογικών κοινωνικών παραγόντων στην εποπτική αξιολόγηση και στις δοκιμές αντοχής είναι εργαλεία που εποπτικές αρχές μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να οθήσουν τις τράπεζες να λαμβάνουν περισσότερο τις πτυχές αυτές ε, υπόψη τους. Καλώς. Κοιτάξτε, η βιωσιμότητα, η βιωσιμότητα είναι αρκετά σημαντική. Αυτό ήθελα να πω. Κοιτάξτε το χρηματοσυντικό τομέα. Οι ασφαλίσεις και οι συντάξεις έχουν διαφορετικό επιχειρηματικό μοντέλο και η βιωσιμότητα λαμβάνεται περισσότερο στις συντάξεις υπόψη και στις ασφαλίσεις. Είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε ότι στις ασφαλίσεις δεν είναι μόνο το θέμα των στοιχείων ενεργητικού, αλλά και των ευθυνών. Η αλλαγή του κλίματος όσον αφορά τη στήριξη των ασφαλιστών, την αντασφάλιση των ασφαλιστών, την εγγύηση των ασφαλιστών, είναι καλό κίνητρο να κινηθούν προς οικονομία χαμηλού άνθρακα. Και η ασφάλιση μπορεί να δώσει τα κατάλληλα κίνητρα τόσο ώστε να αλλάξει η οικονομία. Πώς τα βλέπουμε τα πράγματα στην ΑΙΟΠΑ. Είναι γενική οριζόντια προσέγγιση. Δεν υπάρχει μια και λύση. Πρέπει να δούμε τι γίνεται από πλευρά των κεφαλαίων, αλλά τι γίνεται με την κυβέρνηση, διαχείριση των κινδύνων και από πλευρά διαφάνεια. Ε, είπατε, το είπε αυτό, Πολ, και το εξετάζουμε. Θέλουμε να συμπεριλάβουμε για τη δοκιμή αντοχή το 2019 του τομέα των συντάξεων και ένα στοιχείο που αφορά την βιωσιμότητα και το ίχνος άνθρακα. Ευχαριστώ. Ashley Fox. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και να ευχαριστήσω και τους τρεις ε, πρόεδρους. Είμαι εισηγητής ε, στην κανονισμό για την ε, ευρωπαϊκή μαζική χρηματοδότηση και βεβαίως τα είχαμε συζητήσει αυτά και στις συνεδριάσεις των σκιωδών εισηγητών. Θα απευθυνθώ τώρα στον πρόεδρο της ΕΣΜΑ. Εμείς είχαμε προτείνει πως η ΕΣΜΑ θα πρέπει να εποπτεύει τις πλατφόρμες είπε αυτό το καστός, αλλά η ομάδα μου είναι πολύ επιφυλακτική και γνωρίζω από ιδιωτικές συζητήσεις πως και η ΕΣΜΑ ανησυχεί για την ανάληψη αυτού του ρόλου και από πλευράς δυνατοτήτων αλλά και από πλευράς αποτελεσματικής διοίκησης ε, καθώς θεωρούμε πως οι εθνικές εποπτικές αρχές είναι σε καλύτερη θέση υποπτίας αυτού του προϊόντος και άλλα ανησυχώ και για το τι θα σημαίνει αυτό στην πράξη. Ο κανονισμός αυτός εξαρτάται από το να λειτουργούν οι πλατφόρμες με μία άδεια PST, η ε, οποία υποπτεύεται σε εθνικό επίπεδο. Κύριε Πρόεδρε, θεωρείτε πως η ΕΣΜΑ θα είναι σε θέση να έχει μια σαφή άποψη των ρυθμιστικών πρακτικών, πόσο μάλλον της πείρας και της ικανότητας να ε, χειριστεί αυτό το καθεστώς ενθαρρυνθήκα από την δήλωσή σας για το πώς εφαρμόσατε τα εργαλεία αυτά στην MIFID και θα ήθελα να σας ρωτήσω σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι οι ανάλογες τέτοιες αρμοδιότητες θα τέριαζαν στον κανονισμό του crowdfunding για να υπάρξει ομοιόμορφη εφαρμογή σε όλα τα κράτη-μέλη. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα βεβαίως Χαίρομαστε για το ότι η Κομισιόν μας εκτιμά και θέλει να μας δώσει επιπλέον ρυθμιστικές αρμοδιότητες. Αυτό το οποίο είπα εγώ είναι πως ε, το λογικότερο είναι να μας δοθούν νέες αρμοδιότητες που είναι πιο κοντά στην αγορά χονδρικής ε, στα αποθετήρια, παραδείγματο τα κτλ. Αυτό είναι λογικό να γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ενώ αφετέρου τομείς όπου υπάρχουν πολλές επαφές με τους καταναλωτές σε διάφορες γλώσσες όπου χρειάζεται κανείς να αντιλαμβάνεται την τοπική κατάσταση ε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνουν ε, ως άμεση εποπτεία από το ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πιο λογικό να γίνει στο εθνικό επίπεδο αλλά να υπάρχει η κατάλληλη ρυθμιστική σύγκληση κατά το οποίο αναφέραμε όλοι στις δηλώσεις μας. Ε, συγκεκριμένα λοιπόν για το θέμα του crowdfunding, νομίζω ότι ήδη το 2014 είχαμε δημοσίευσει μια γνωμοδότηση όπου λέγαμε ότι καλό θα ήταν να υπάρχει μια νομοθεσία ειδικά για αυτό το ζήτημα ε, το οποίο έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Προσωπικά εγώ κοιτώντας και τον ρόλο που θα έχουμε θα έλεγα πως οι μικρότερες επενδύσεις ε, στο ευρωπαϊκό επίπεδο αυτή τη στιγμή αυξάνονται σε μέγεθος, θα επανέρχονται στο εθνικό επίπεδο και άλλα ο ρόλος της ΕΣΜΑ θα αφορούσε τις μικρότερες επενδύσεις και όχι τόσο πολύ τις μεγαλύτερες. Και επιπλέον η ΕΣΜΑ θα ανταγωνιζόταν με τις εθνικές αρμόδιες αρχές ε, γιατί η πλατφόρμα αυτή θα είχε την επιλογή αν θα το έκανε σε εθνικό ή σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και νομίζω πως αυτός ο σχεδιασμός μπορεί να βελτιωθεί. Νομίζω πως θα είναι πιο λογικό να γίνει ακριβώς μια επιλογή των μεγαλύτερων εκείνων περιπτώσεων που είναι πιο λογικό να γίνουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ οι μικρότερε βεβαίω θα είναι πιο λογικό να γίνουν σε τοπικό επίπεδο κιόλα. Σα ευχαριστώ. Θα κάνουμε αυτό το οποίο προτείνετε λοιπόν. But you didn't ask about ICO. Δεν ρωτήσατε το ICO, γιατί αυτή είναι η πιο δύσκολη ερώτηση. <laughs> No, because if you want to improve a... Όχι, για να βελτιωνόμαστε, ανάλογα με τις ε, προτάσεις και τις υποδείξεις, να βελτιωνόμαστε και εμείς. Ωραία. Ο Βολφ Κλίντς. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να το θέμα το ξεπλήματος και εγώ δεν θέλω να το κουράσω πάρα πολύ, αλλά αρκεί πραγματικά να έχει τη βασική ευθύνη γι' αυτό η EBA, η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή. Αν, αν μειώσουμε το ξέπλυμα ε, στο τραπεζικό τομέα θα το μετατοπίσουμε. Ε, πολύ υπάρχει στη χώρα μου στην κτηματαγορά, στο λαθρεμπόριο ε, όπλων, ναρκωτικών, στην πορνεία, πάρα πολύ ισχυρά. Δηλαδή αν έχουμε μια ευρωπαϊκή τραπεζική εποπτεία που είναι αρμόδια για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και να την περιορίσει, τότε τα πλυντήρια θα βρούνε άλλους δρόμους και άλλους τρόπους για να ξεπλένουν χρήματα και ακόμα και στο χρηματοπιστωτικό τομέα θα πάνε στις παρατράπεζες ή στις σκιώδεις τράπεζες που δεν ελέγχονται. Ε, ε, χρειαστεί λοιπόν να την ε, προχωρήσουμε λίγο παρακάτω αυτή τη σκέψη. Ξέρετε ότι δεν μου αρέσει να δημιουργούνται νέοι οργανισμοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και νέε αρχέ, γιατί έχουμε προβλήματα με του πολίτε που σου λέει και άλλη γραφειοκρατία και άλλο οργανισμό φτιάχνουν. Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση, μήπω χρειαζόμαστε μία αρχή ξεχωριστή, αυτόνομη, που δεν θα έχει μόνο την εποπτεία, αλλά μπορεί να επιβάλλει και κυρώσει, χωρί να πείπτει ράβδο. Δεν πρόκειται να λειτουργήσει όλο αυτό το θέμα. Αυτό το δεύτερο. Στίβεν Μαγιόρ, σωστά αναφέρθηκε στο ε, θέμα ανάμεσα στο Users Kit και τα PRIPS, ε, δηλαδή ε, το έγγραφο βασικών πληροφοριών και τα PRIPS. μέχρι τις αρχές του επόμενου έτους δεν νομίζω να προβλέπουμε ε, να, μπορεί να λυθεί το πρόβλημα, ούτε μέχρι τα τέλη του έτους. Ε, έχουμε το Μάιο ευρωεκλογέ από το Μάρτιο-Απρίλιο το Κοινοβούλιο θα κλείσει, μετά θα πρέπει να στηθεί το νέο Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πάει λέγοντας. Και προβληματίζομαι και διερωτώ με μήπως θα μπορούσαμε να πούμε ότι θα παραμείνει το έγγραφο βασικών πληροφοριών, το usage kit δηλαδή και τα αντίστοιχα δεν λήγουν το τέλος του 19 ή το 2020 και αν βελτιωθεί το kit του PRIPS και γίνει μια σκληρή ε, αξιολόγηση ε, να συγχωνευτούν τα δύο όποτε έρθει αυτή η ώρα μετά από ένα-δύο χρόνια. Και το τρίτο και τελευταίο αφορά ε, τις επιστολές αδράνειας, no action letters. Υπάρχει ήδη αυτό στις Ηνωμένε Πολιτείες, στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι στιγμής όχι. Και διήστανται πάρα πολύ απόψεις αλλά θα μπορούσα να φανταστώ ότι θα είχε νόημα και εδώ να εισαγάγουμε αυτό το ε, μέσο και το εργαλείο. Τελειώνω, τελειώνω. Ε, εάν διαπιστώνουμε. την πρότασή μου να βάλω μια τελεία, ούτε αυτό δεν με αφήνεται. Λοιπόν, όταν βλέπουμε ότι δεν μεταφέρεται ε, μια νομοθεσία και δεν εφαρμόζεται, να υπάρχουν και αντίστοιχες προτάσεις και συνέπειες. Απάντησε. Κοιτάξτε, όσον αφορά το ρόλο της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής, υπήρχε μια ομάδα υπό το συντονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εκπροσωπούνται και τις Επιτροπικές Αρχές. Συνεπέρανε ότι μέσω μακροπρόθεσμα Λοιπόν, ειδικό φορέα, ένα ευρωπαϊκό φορέα για την καταπολέμηση του χρήματο μαζί με τον κανονισμό ίσω θα χρειαζόταν για καλύτερο εναρμονισμένη εφαρμογή. Ήδη ολοκληρώθηκαν οι σχετικέ συζητήσει και η ομάδα συνεπέρανε ότι για την ώρα είναι δύσκολο να φτάσουμε σε αυτό το στόχο τόσο μακριά όσον αφορά την κεντρική αντιμετώπιση των ευθυνών και ίσως θα είχαμε κάποιο ρόλο να εξασφαλίσουμε σωστό συντονισμό όσον αφορά ανταπόκριση στο θέμα αυτό. Και ο ρόλο της Ευρωπαϊκής Τραπεζική αρχή δεν θα περιοριστεί στις τράπεζες. Υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής ε, περιεσίας Τραπεζών να δημιουργήσουμε, ε, να έχουμε κοινή ε, απάντηση όσον αφορά τα προβλήματα με το ξέπλυμα βρώμικου χρήματο. Πολύ γρήγορα για το usage kit. Θέλουμε να επεκτείνουμε την εξαίρεση για usage στα πλαίσια του PRIPS. Αλλά αυτό θα συνέχιζε να εφαρμόζει αθέμητους κανόνες για τα ασφαλιστικά προϊόντα. Γι' αυτό οι τρεις αρχές θέλουν να κινηθούμε τάχιστα. Προφανώς θα σεβαστούμε τη λήξη της θητείας σας και ότι θέλετε εγκαίρως να ολοκληρωθεί το νομοθετικό σας έργο. Εργαζόμαστε σκληρά για να ολοκληρωθεί το έργο το πρώτο τρίμηνο του χρόνου, λαμβάνοντας υπόψη το ότι κατανοούμε ότι θα υπάρξει δυνατότητα, ευκαιρία που θα είναι όμως, θα έχει μικρή διάρκεια. Στο πρώτο τρίμηνο του επόμενου έτους η καλύτερη επιλογή είναι γρήγορη αξιολόγηση. Οι εκθέσεις είναι έτοιμε στο πρώτο τρίμηνο του επομένου χρόνου για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μπορεί αυτή να αποφασίσει ακολούθως για ενδεχομένε νομοθετικέ τοπολογίε. Για το θέμα αυτό, την επιστολή για μη δράση, πρέπει να το εξετάσουμε Πρόσφατα υπήρχε υποχρέωση εκαθάριση σε τριξωτικά ταμεία και το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο είχαν αποφασίσει ότι θα έπρεπε να αναβληθεί υποχρέωση εκαθάρισης ή περίοδος εξαίρεσης. Και τελικά σε μια δήλωση είπαμε ότι δεν είναι εποπτική προτεραιότητα αυτή. Βέβαια αυτό δεν γίνει και τη μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου στους εμπλεκομένους Οποιαδήποτε βοήθεια επ' αυτού θα ήταν κάτι που θα εκτιμούσαμε αφάνταστα. Ευχαριστώ πολύ. Σβέν Γκίγκολντ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και χαίρομαι που σας ε, ξαναβλέπουμε. Έχω να αφαιρθώ στο θέμα του ξεπλήματος χρήματος ξανά. Πρέπει να διακρίνουμε δύο πράγματα. Το ένα είναι το τι κάνουμε μακροπρόθεσμα και το τι χρειαζόμαστε τώρα για να επιτύχουμε κάποια πρόοδο και δεν πρέπει το καλύτερο να είναι εχθρός του καλού. Οπότε τώρα είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε ό,τι μπορούμε αυτή τη στιγμή για να εφαρμόσουμε κάποια πράγματα και από την άλλη να μην κλείσουμε τη... ενδεχόμενο μιας μακροπρόθεσμης λύσης. Γι' αυτό ακριβώς λοιπόν θα ήθελα να ρωτήσω την ΕΣΜΑ και την ΑΙΟΠΑ να μας πούν πόσους πόρους έχουν αφιερώσει αυτήν την στιγμή στην καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος. Ποιο και πόσο προσωπικό εργάζεται πάνω σε αυτό το θέμα και τι σκοπεύετε να κάνετε στις αρχές που διευθύνετε. Κατόπιν, Γκαμπριέλ, για την ΕΙΟΠΑ. Είχαμε ήδη κάποιες ε, συζητήσεις ε, το θέμα της ε, για το θέμα των αργυραμιβών λοιπόν έχετε λάβει κάποια έχετε λάβει κάποια θέμα για κάποιες πρωτοβουλίες για το θέμα του ορισμού του στον τομέα των ασφαλιών. Πρέπει να το δούμε. Αξίζει αυτός ο καταναλωτές. Και τέλος, προς την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή, μου προξενεί κάποια έκπληξη το ότι παρά την τοκοκληφία στον ε, τομέα του συναλλάγματος ε, η αρχή σας είναι κατά του να υπάρχει μια δυνατότητα για την αρχή σας να περιοριστούν τα υπερβολικά τέλη για την μετατροπή των νομισμάτων σε ευρώ στην κοινή αγορά. Και πάλι δεν αντιλαμβάνομαι γιατί είστε κατά. Πρέπει να αναλάβουμε δράση από κοινού νομίζω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, για το θέμα του ξεπλήματος ε, χρήματος... Ε, Βεβαίω πρέπει να έχουμε κάποιες προτεραιότητες στην κατανομή των πόρων. Εστιάζουμε στο θέμα της ρυθμιστικής σύγκλησης, οπότε μπορώ να είμαι σύντομος. Έχουμε δώσει ελάχιστου πόρους θα έλεγα βασικά συμμετέχουμε στην μεικτή επιτροπή και βεβαίως ε, το θέμα αφορά και τις ασφαλίσεις και τις συντάξεις και υπάρχουν διαφορετικά στοιχεία που μας δείχνουν ότι κάτι τέτοιο μπορεί να είναι δυνατό. Γι' αυτό ακριβώς ε, θεωρώ ότι περισσότεροι πόροι σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι η καλύτερη λύση τελικά. Ε, θα το κάνετε τώρα ή όχι. Ε, κοιτάξτε, δεν έχουμε αυτή τη στιγμή τους πόρους ε, για να αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα αυτά, γιατί θα πρέπει να αφαιρέσουμε τους πόρους από άλλα ζητήματα, όπως τις διασυνοριακές συναλλαγές, που είναι πιο σημαντικά, όπως είπα. Για τα άλλα ζητήματα που αναφέρατε, πράγματι αυτά είναι κάποια προϊόντα τα οποία στοχεύουμε και βεβαίως ε, έχουμε κάνει κάποια δουλειά όσον αφορά την ασφάλιση προστασίας πληρωμών. Είναι ένα ιδιαίτερο κλάδος όπου ο ρόλος των προμηθειών επηρεάζει πάρα πολύ το αποτέλεσμα και ξεκινήσαμε και εξετάζουμε αυτή τη στιγμή σε ολόκληρη την Ευρώπη την ταξιδιωτική ασφάλεια γιατί έχουμε κάποιες επιφυλάξεις ε, όσον αφορά την προστιθέμενη αξία για τους ε, καταναλωτές. Και ακριβώ ε, εξετάζουμε το πώς θα μπορούσαμε να δούμε τον κίνδυνο για τους λιανικούς καταναλωτές, ένα από τα οποία βεβαίως αφορά και τις προμήθειες ε, οι οποίες χρεώνονται και τώρα βρισκόμαστε στην δεύτερη φάση όπου ακριβώς ε, λαμβάνουμε υπόψη ε, και στην πρίψ την κατάσταση αυτή και έχουμε μπει σε πολύ πιο βαθιά νερά με τις εθνικές αρχές για να αντιληφθούμε το πώς γίνεται και έχουμε ξεκινήσει και τις ε, επισκέψεις. Ε, κοιτάμε συγκεκριμένα προϊόντα πια. Αντιμετωπίζουμε διάφορες ε, καταστάσεις και οπωσδήποτε αυτό θα μας απασχολεί στα επόμενα χρόνια. Σύντομα τώρα, δεν γνωρίζω τον αριθμό των ανθρωπορών ε, θα είναι οπωσδήποτε κάτι παρόμοιο με αυτό του Γκάμπριελ. Να σας πω επίσης πως ε, η δική μας εμπειρία είναι περιορισμένη γιατί κατά κανόνα αυτό δεν αντίθεται στην ρυθμιστική αρχή των αξιογράφων, αλλά στην αρχή των τραπεζών ή σε κάποιον άλλον ο οποίο ασχολείται με το ξέπλυμα χρήματο. Οπότε υπάρχει και θέμα αποτελεσματικότητας. αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει ξέπλυμα χρήματος αλλά βεβαίως ε, η είσοδος θα έλεγα γίνεται μέσω του τραπεζικού συστήματος και γι' αυτό ακριβώς εμείς λέμε ότι θα πρέπει να έχουμε αυτή τη στιγμή έναν συμβουλευτικό ρόλο αλλά έχει νόημα νομίζω να τα λάβει αυτά η τραπεζική αρχή. Θα κάνετε κάτι περισσότερο. Ε, κοιτάξτε, πέρσι ήδη στο πλαίσιο της ε, κοινή επιτροπής έχουμε αποφασίσει να αφιερώσουμε περισσότερους πόρους στο θέμα. Για τις υπηρεσίες σύγκλησης των νομισμάτων, το έχουμε κοιτάξει αυτό με εκπροσώπους των καταναλωτών στην ομάδα των ενδιαφερομένων, των stakeholders. Εγώ δεν νομίζω να διαφωνεί η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή με το RTS. Αν το ζητήσει και το επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία θα το κάνουμε. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αλλά δεν είμαι βέβαιος ότι τα ανώτατα όρια στις τιμές είναι ο σωστός τρόπος να προχωρήσουμε. Ότι υπάρχει θέμα που πρέπει να λυθεί, υπάρχει. Πρέπει να ξαναδούμε ε, κάποια μέσα και εργαλεία και να λάβουμε δράση στο τομέα αυτό. Ευχαριστώ. Δεν έχω μιλητέ από την ΚΟΥ, η FTD και η ΕΝΕΦ, λέει ο Πρόεδρος. Όλα. Λαμασούχ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στα αγγλικά ο κύριος Λαμασούχ. Θα συνεχίσω από την ερώτηση που έκανε ο συνάδελφος Κλίντς. Την περασμένη εβδομάδα στέλατε μια επιστολή ε, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το έγγραφο βασικών προφοριών PRIPS ε, και τα λοιπά. Για το 19 θα επανέλθετε για να κάνετε αλλαγές στο εγγράφο βασικών ε, πληροφοριών πριν εφαρμοστεί στα προϊόντα ως ΕΚΑ, usage. Μέχρι τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει απαντήσει τι συνέχεια θα δώσει. Πότε πιστεύετε ότι θα μπορέσουν να επιβληθούν ως ευρωπαϊκή νομοθεσία αυτές οι αλλαγές. Πόσο χρόνο χρειάζονται οι φορείς των αγορών για να ε, προσαρμοστούν. Γιατί όλα αυτά θα πρέπει να είναι έτοιμα μέχρι τα τέλη του επομένου έτους, που μου φαίνεται πάρα πολύ μικρό διάστημα. Ευχαριστώ. Ε, κύριε Λαμασού, να απαντήσω εγώ, λέει ο κύριος Μπερναρντίνο. Όπως είπε ο Στίβεν Μαγιόρ, πιστεύουμε ότι μπορούμε αυτές τις προσαρμογές να τις έχουμε έτοιμες σχετικά γρήγορα. Κάποιες μικροαλλαγές δεν είναι εκ αναθεώρηση του ΠΡΙΠΣ. Ή κάποιες μικροαλλαγές και προσαρμογές ως προς τις επιδόσεις ας πούμε. Αλλά για να είμαι πολύ ειλικρινής μαζί σας, πρέπει να πω ότι γίνεται μέγας λόγος για το έγγραφο βασικό πληροφοριών ΠΡΙΠΣ και ότι δεν είναι και τόσο αποτελεσματικό. Εμείς έχουμε τις αφιβολίες μας, δεν έχουμε στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι κάποια από αυτά που αναφέρονται ήταν εις βάρος των καταναλωτών και τα λοιπά, ότι τους βλάπτουν. Δεν έχουμε τέτοια στοιχεία. Το κόστος των συναλλαγών που πολύ συχνά αναφέρεται είναι μάλλον ένα θέμα στρεβλής εφαρμογής, κακής εφαρμογής και όχι μεθοδολογίας. Τι κάνουμε λοιπόν ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει κάποιες μικροβελτιώσεις που μπορούμε να πούμε από την εμπειρία μας ότι χρειάζονται και βελτιώνουν την κατάσταση και στις αρχές του 19 θα κάνουμε προτάσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να τις υποβάλει σε εσά και να ολοκληρωθούν όλα αυτά εγκαίρως έτσι ώστε να υπάρχει και χρόνος για την εφαρμογή. Και θέλω να υποστηρίξω αυτό που είπε ο Στίβεν Μαγιόρ. Αυτό που έχει σημασία και εδώ είναι να είναι παντού ήδη οι κανόνες του παιχνιδιού ε, ως προς την ενημέρωση των καταναλωτών και των ε, επενδυτικών ε, ταμείων και των ασφαλίσεων. Με τον κίνδυνο της επαναλήψεως να πω και εγώ ότι παρατηρούμε ότι υπάρχουν θέματα εφαρμογής όσον αφορά το PRIPS. Κάτι που αναφέρα και εγώ στην αρχή είναι το θέμα του πεδίου εφαρμογή. Κάποια προϊόντα είναι εντό πεδίου εφαρμογή και καλύτερο θα ήταν να μην είναι και υπάρχει και νομικό επιχείρημα υπέρ στενότερου πεδίου εφαρμογή, κυρίω όσον αφορά το θέμα διάφορων ομολόγων και διάφορα κενά που υπάρχουν σε κάποια κράτη-μέρη. Δεν εκδίδονται πλέον κάποια ομόλογα προ όφελο των λιανικών επενδυτών και αυτό αντιβαίνει την προοπτική τη ενώσεω τη ενιαία αγορά κεφαλαγορών, τη ενιαία κεφαλαγορά. Είδαμε και θέματα επιδόσεων και μέσω ερωτηματολογίου το αντιμετωπίσαμε η μεγαλύτερη ανησυχία για τις τρεις αρχές είναι οι επιδόσεις. Κάτι που θα αντικατοπιστεί και στην επιστολή. Πρέπει να είναι στο επίκεντρο των, της στοχευμένης αξιολόγησης για το κόστος συναλλαγών. Δεν έχουμε πιστεί ακόμα ότι είναι θεμελιώδες πρόβλημα. Ξέρουμε ότι είναι περίπλοκη η μεθοδολογία. Απ' την άλλη αντικατοπτήσει το γεγονός ότι κάθε φορά που αγοράζεις και πουλάς χάνεται κάποια οικονομική αξία και αυτό πρέπει να αντικατοπτήσει τις επιδόσεις των προϊόντων αυτών που πολλούνται σε πακέτα. Σε περιπτώσεις όπου ο τομέας ανησύχησε, περί κόστου συναλλαγής ζητήσαμε στοιχεία και η αξιολόγησή μας γίνεται βάση στοιχείων και αφορά περισσότερο λανθασμένη εφαρμογή της μεθοδολογίας από ότι τη μεθοδολογία αυτή καθεαυτή. Γι' αυτό κανείς μπορεί να επιχειρηματολογήσει υπέρ στοχευμένης αναθεωρήσεως που θα επί των επιδόσεων. Προφανώς είμαστε σε επαφή και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτή θα πρέπει να τοποθετηθεί και να πει κατά πόσο αυτό είναι κάτι είναι εφικτό. Χρειάζεται κουβέντα πριν εκφράσουμε την εκτίμησή μας για τη δέουσα λύση. Το καταλαβαίνουμε βέβαια ότι τα χρονικά περιθώρια είναι πολύ στενά. Καλώς. Δεν έχετε σχόλια. Νίνα Γκίλ, ευχαριστώ. Ε, ήδη το συζητήσαμε αυτό. Ο ΙΕ εξέδωσε ανησυχητική έκθεση. Είπε ότι πρέπει να δράσουμε επιγόντως για το κλίμα. Κάτι που είπε ο Πολ για το χρηματοστικό τομέα που έχει βασικό ρόλο να παίξει στον αφορά το θέμα αυτό εξετάζουμε το θέμα της προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για φιώσιμη χρηματοδότηση. Και την δέουσα μεταρρύθμιση. Είναι μετριοπαθής οι προτάσεις. Ξέρω, άκουσα, μ' αρέσει η άποψή σας. Κάπως απαντήσατε. Είπατε τι παραπάνω μπορείτε να κάνετε. Θα μπορούσατε να ηγηθείτε ως εποπτική φορείς. Στίβεν, είπες ότι ο δημόσιος τομέας υστερεί και ότι ο ιδιωτικός τομέας προηγείται τι κάνουμε βάσει των εκθέσεων για να εξασφαλίσουμε στο ότι ο δημόσιο τομέας θα μείνει πίσω. Γκάμπριελ, είπες ότι θα αναλάβει δοκιμές αντοχή για τον τομέα των ασφαλίσεων. Θα ήταν δυνατόν, μήπω, για το υψηλό βαθμό εκθέσεως επενδύσεων ε, των συνταξιωτικών ε, ταμείων στους βιώσιμους τομείς ή στην πυρηνική ενέργεια μιλήσατε για αρνητικές συνέπειες ε, της μη πράσινή οικονομίας στις τράπεζες. Μπορεί να κάνω το ίδιο εδώ. ΕΣΜΑ, Brexit. Ετοιμάζεται κάποιο μνημόνιο συνεννόησης για εποπτική συνεργασία με το Ηνωμένο Βασίλειο. Το ξεκαθαρίζετε κάπως. Πού βρισκόσαστε. Πότε θα ολοκληρωθούν οι προσπάθειες. Υπάρχουν πολλές ανησυχίες στον κανονισμό για τα επενδυτικά ταμεία. Στείλατε επιστολή πρόσφατα στον αντιπρόεδρο Τρομπόφσκης και είπατε ότι θέλετε αναθεώρηση του ΜΥΦΙΔ από ό,τι κατάλαβα. Γιατί πράγμα ανησυχώ ότι κάποια από αυτά δεν εφαρμόζονται καν σωστά και πάμε προς αναθεώρηση ε, ε, κάποιου ανέτοιμου μέτρου. Αυτό θα έχει συνέπειες ε, μετά, ε, για την ενιαία αγορά, την νομισματική μετά το Brexit. Λοιπόν, τι γίνεται, είμαστε για την ένωση κεφαλογορών. Και κάτι άλλο για την καταπολέμηση του ξεπλήματος χρήματος. Διάφοροι συνάδελφοι τα ανέφεραν αυτό. Καλωσορίζουμε τη δράση που κάνατε ε, κατά της DUSK και της ING. Ίσως θέλετε περισσότερες εξουσίες που δεν σας δίνουν τα κράτη-μέλη. Το είδαμε σαν αναθεώρηση. Άρα πώς μπορούμε να λύσουμε το συγκεκριμένο πρόβλημα. So uh, σύντομα, ο κύριος Μαγιόρ, για την βιωσιμότητα και την εμφορία, τώρα θυμήθηκα την ερώτηση ότι χρειάζεστε. Ε, πόρους, τι να χρειαζόμαστε. Ε, μάλλον έχετε κουραστεί να τα ακούτε αυτά από τις αρχές. Δυστυχώς, χρειαζόμαστε πόρους. Έτσι έχουν τα πράγματα για να κάνουμε τη δουλειά μας για το πώς θα ενταχθεί και η βιωσιμότητα και στην παροχή συμβουλών, benchmarks, ορόσημα, όλα αυτά χρειάζονται πόρους. Κατά την άποψή μου, το πρόγραμμα δράσης είναι σωστό και χαιρόμαστε με τις ε, δράσεις που έχουν ανατεθεί στην Ευρωπαϊκή Αρχή ΕΣΜΑ και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κίνδυνου. Για το θέμα ε, του Μνημονίου Συνεννόησης. Περί τίνος πρόκειται. Αν γίνει άτακτο Brexit, χωρίς συμφωνία θα έχουμε ένα μνημόνιο συνεργασίας και συνεννόησης ε, όπως με πάρα πολλές ε, τρίτες χώρες. Έχουμε κάποια μνημόνια που μας επιτρέπουν να λειτουργούμε για την προστασία των επενδυτών και την ασφάλεια. Ας πούμε, όταν θέλετε να κάνετε μια έρευνα για κατάχρηση αγοράς και ένας από τους εμπόρους ή τους, τους traders είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, χρειάζεται αυτό το μνημόνιο για ανταλλαγή πληροφοριών που χρειάζονται όταν κάποιος ε, ε, μπλεκόμενος φορέας είναι εκτός της Ένωσης. Τέτοιου είδους μνημόνια συνεννόηση χρειαζόμαστε και μέχρι το Μάρτιο ε, του 19 πρέπει να υπάρχει με το Ηνωμένο Βασίλειο. Τώρα που βρισκόμαστε η Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές ε, των 27 που έχουν συμφωνίες με το Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και με την ΕΣΜΑ και λόγω των δικών μας αρμοδιοτήτων είπαμε ότι θα προσπαθήσουμε να έρθουμε με μια κοινή θέση για τα μνημόνια συνεννόησης. Έχουμε φτάσει σε αυτό το στάδιο ήδη και λαμβάνοντας υπόψη και τις ευρύτερε διαπραγματεύσεις και το χρονοδιάγραμμα, αργότερα θα απευθυνθούμε στους συναδέλφους του Ηνωμένου Βασιλείου για να βεβαιωθούμε πάντα ότι είμαστε ε, ε, πρόθεσμοι πριν τα τέλη Μαρτίου. Γιατί θα πρέπει όλα αυτά να τα γνωρίζουν οι ενδιαφερομένοι εγκαίρως πάρα πολύ. Για το MIFID και το MIFIR και τη σχετική επιστολή είναι λίγο άσχετο αυτό το θέμα σε κάποιο βαθμό. Τι βλέπουμε. Η ευρωπαϊκή νομοθεσία προφανώς δεν ήταν πάντα σχεδιασμένη ε, με το να έχουμε εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης πολύ κοντά μας μια πολύ μεγάλη ε, αγορά με μεγάλη ρευστότητα. Πώς <laughs> λοιπόν θα προετοιμαστούν οι MIFID και MIFIR ε, σε αυτή τη νέα κατάσταση ότι πολύ κοντά μας θα έχουμε την αγορά αυτή με πολλά, πολύ υψηλή ρευστότητα. Αυτό θα το δουν και 27. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάνει σχετικά προτάσεις ε, στο ΕΜΙΡ, ας πούμε, που το αντικατέστησε από το ΕΜΙΡ 2 και στο ΕΣΜΑ, αντίστοιχα και στο Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να δούμε το ΜΥΦΙΤ και το ΜΥΦΙΡ αν είναι το κατάλληλο πλαίσιο για το νέο περιβάλλον. Όμω δεν θέλουμε να σταματήσουν να κλείσουν οι συναλλαγέ με τρίτε χώρε, απλώ να έχουμε ε, ίσου κανόνε παιχνιδιού ανάμεσα ε, σε επενδυτικές ε, εταιρείε ε, και στις αγορές εντός και εκτός τη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί τι γίνεται τώρα, στις περισσότερες περιπτώσεις η οδηγία και ο κανονισμός μη MIFIR έχουν το πρόβλημα ότι το εθνικό επίπεδο δεν είναι αρμονισμένο με το ευρωπαϊκό και πολλά κράτη-μέλη επιτρέπουν ε, πρόσβαση από εμπόρους ή ε, επενδυτικές εταιρείες ε, που επενδύουν σε υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έρχονται από το εξωτερικό. Ο κύριος Μπερναρντίνο για τα δύο τελευταία για το μνημόνιο συνεννόησης με τις αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου. Το ίδιο κάνουμε και εμείς με την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή. Συνεργαζόμαστε με τις εποπτικές αρχές των 27 κρατών μελών έτσι ώστε να μπορούμε και από την ΕΙΟΠΑ να έχουμε μια συνεννόηση σε περίπτωση που δεν επέλθει συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο για το Brexit. Πολύ σημαντικό αυτό. Για το θέμα της δράσης και της αλλαγές που γίνονται σε σχέση με τη βιωσιμότητα και την αηφορία. Συμφωνώ. Αυτό μπορεί να γίνει και χωρίς ταξινόμηση. Βέβαια, η ταξινόμηση θα μας διευκόλυνε σε πολλές περιπτώσεις για τα stress test ή διάφορες αναλύσεις. Ε, αλλά προσπαθούμε και χρησιμοποιώντας και τη δημόσια πληροφόρηση ε, για τα στοιχεία ενεργητικού σε διάφορους τομείς της οικονομίας να αναλύσουμε ε, ποια είναι η έκθεση πούμε, ασφαλιστικών εταιριών για να κατανοήσουμε πού βρίσκονται. Γιατί αυτό μπορεί να είναι ρίσκο κίνδυνο στο ίδιο του το χαρτοφυλάκιο και πρέπει να αρχίσουν να το διαχειρίζονται. Πάντω έχουν αρχίσει να το σχεδιάσουν, να το προγραμματίζουν και να έχουν τις επενδυτικές τους ε, δομές και στα πλαίσια της ε, ε, οδηγίας για την ε, φερεγγιότητα. Δύο. Και δεν είναι μόνο τα στοιχεία ενεργητικού και του παθητικού. Θα πρέπει να υπάρξει μια μετάβαση σταδιακή, γιατί αυτό είναι ένα από τα ρίσκα. Όταν κάποιος αναβάνει μια δράση κάποια στιγμή, να μην έχουμε ένα κόσμο 0-1, όπου θα έχουμε ένα μεγάλο αριθμό στοιχείων ενεργητικού που θα έχουν αποτύχει. Δηλαδή θα πρέπει ο κύκλος αυτός να είναι ενάρετος έτσι ώστε οι συντάξει και οι ασφάλειες ε, να έχουν τις απαραίτητε ε, επενδύσεις, τα κίνητρα για να επενδύουν οι εταιρείε σε μια ε, μεταβατική οικονομία στη μετάβαση προς την απαγκίστρωση από το διοξίδιο του άνθρακα. Γι' αυτό θα ε, κάνουμε και τις δοκιμές αντοχής στα στρες test του χρόνου για τις ασφάλειες και τις, ε, ε, τα συνταξιωτικά ταμεία. για το θέμα αυτό δεν είναι ότι η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή θέλει περισσότερες αρμοδιότητες γιατί στέκονται τα κράτη. Αλλά έχουμε πρόβλημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχουμε μία ενιαία αγορά και βεβαίως η εποπτεία μπορεί να είναι τόσο ισχυρή όσο ο ασθενέστερος κρίκος. Οπότε βλέπουμε ε, χρήματα, προϊόν εγκλήματος να μετακινούνται από εδώ και από εκεί και δεν υπάρχει απαραίτητο συντονισμός. Κάποιες τράπεζες που κατά βάση ε, έχουν κλείσει ε, κατόπιν παρεμβάσεων των Αμερικανικών αρχών. Έχουμε λοιπόν ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα. Το θέμα είναι πώς θα το λύσουμε. Το έγγραφο και η πρόταση της Κομισιόν προτείνουν κάτι και εμείς είμαστε έτοιμοι βεβαίω. να δώσουμε κάποια στήριξη στην πρώτη φάση γιατί δεν υπάρχουν άλλα εργαλεία διαθέσιμα. Και έχουμε αναπτύξει κάποια πείρα σε αυτόν τον τομέα. Για τον Brexit να προσθέσω επίσης πως η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή έχει εγκρίνει αυτό το οποίο λέμε κάποια μνημόνια πλαίσια με τις αρχές ε, του Ηνωμένου Βασιλείου και είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε με τους Βρετανούς ε, συναδέλφους ε, καθώς θα περάσουν σε αυτή την φάση διαπραγματεύσεις. Ελπίζουμε σύντομα βεβαίως γιατί ο χρόνος ε, τελειώνει. Σας ευχαριστώ και επί τη ευκαιρία να ευχαριστήσω και την ΕΣΜΑ για την επιστολή για τις επενδυτικές εταιρείε. Και Μάρκους, να απευθύνομαι στον εισηγητή Ευχαριστούμε, Στίβεν. Λοιπόν, θα τα δούμε αυτά στον τριμερή διάλογο και θα δούμε πώς θα ενσωματωθούν. Υπάρχουν πολύ καλές προτάσεις. Αν Σαντέρ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τους Προέδρους για την ανταλλαγή αυτή απόψεων που έχουμε. Δύο ερωτήσεις έχω να σας κάνω. Σήμερα βλέπουμε να αναπτύσσονται και να χρησιμοποιούνται τα κρυπτονομίσματα, όλο και περισσότερο. πρέπει να πλαισιώσουμε αυτή την εξέλιξη, γιατί βλέπουμε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και παγκοσμίω σήμερα, να υπάρχουν λίγα πλαίσια για τη ρύθμιση αυτό. Στις εργασίες μας για το crowdfunding εξετάζουμε κάποιες προτάσεις που στόχο έχουν να ε, υιοθετηθούν κάποιες διατάξεις έτσι ώστε οι πλατφόρμες αυτές crowdfunding να ε, εκδίδουν ICO ή ε, κάποια coins, νομίσματα. Στην Ευρώπη, αν θέλουμε λοιπόν να προχωρήσουμε σε αυτή τη δραστηριότητα, χρειαζόμαστε κάποιες ασφαλιστικές δικλείδες για να προστατευόμαστε από τον κίνδυνο. Αλλά και το πλαίσιο να είναι αρκετά ευέλικτο, έτσι ώστε να μην ε, παρεμποδίζεται η καινοτομία. Πώς τα βλέπετε εσείς όλα αυτά. Πιστεύετε ότι τα κρυπτονομίσματα και τα κρυπτοενεργητικά είναι κάτι ε, ελπιδοφόρο για το μέλλον. Θα πρέπει να το αναπτύξουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να το ρυθμίσουμε, αν το ρυθμίσουμε με βάση ποια στοιχεία. Ε, διατηρώντας πάντα αυτή την ισορροπία ανάμεσα στην ασφάλεια και την ανάπτυξη της αγοράς ε, στην Ευρώπη. Επίσης, θεωρείτε ότι ένα νομοθετικό πλαίσιο crowdfunding είναι σκόπιμο. Και ένα δεύτερο ερώτημα. Είναι κάτι στο οποίο αναφερθήκατε εσείς ε, επιμακρών προηγουμένως και αφορά το θέμα της βιώσιμης χρηματοδότησης. Και σας ερωτώ για συγκεκριμένους δείκτες, τους πράσινους δείκτες λεγόμενους, οικολογικούς. Πώς τα βλέπετε όλα αυτά και πώς πιστεύετε και με τους δείκτες αυτές δεν θα πρέπει να ευνοούνται οι επιχειρήσεις ε, περισσότερο εκείνες που κάνουν ιδιαίτερες προσπάθειες για τη μετάβαση σε μια βιώσιμη οικονομία. Δηλαδή πώς θα αναγνωρίσουμε και κάποιες άλλες επιχειρήσεις που μπορεί να μην είναι τόσο επιμελείς αλλά κάνουν πολύ μεγάλες προσπάθειες. Δηλαδή επιβραβεύονται συγκεκριμένοι μόνο. Και πιστεύετε ότι θα πρέπει οι δείκτες αυτοί να έχουν να κάνουν μόνο με το θετικό ισοζύγιο δεξιδίου του άνθρακα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις δύο ρωτήσεις για τα ICOs και τη βιωσιμότητα. Τι μπορούμε να πούμε τώρα όσον αφορά το ότι με τις αρχικές προσφορές σε νομίσματα θα πρέπει να δείτε ε, σαν ρυθμιστικός φορέας πώς αυτά εντάσσονται στο ρυθμιστικό πλαίσιο των ισχύων και πρέπει να εξασφαλίσει κανείς ότι από τη μια πλευρά ότι οι ισχύοντες κανόνες δεν πνίγουν την καινοτομία, απ' την άλλη οι καινοτομίε θα πρέπει να ανταγωνίζονται σε θεμητό ε, πεδίο ε, με, με ισχύουσες τεχνολογίες ε, και με τους υφιστάμενους νόμους περί συλλογής κεφαλαίων. Τι κάνουμε λοιπόν για αυτά τα νέα μέσα που βγαίνουν να αξιολογήσουμε το πώς είναι θεμητή όρη του ανταγωνισμού μεταξύ των εισερχόμενων χρηματοπιστωτικών καινοτομιών και των υφισταμένων τεχνολογιών. Τι κάνουμε. Σε αυτή τη φάση αξιολογούμε ποια νέα προσφορά χρηματοπιστωτική εντάσσεται στο χρηματοπιστωτικό πλαίσιο. Μερικές από τις νέες προσφορές νομισμάτων σε χρηματοπιστωτικά προϊόντα και με τον κλασικό ορισμό αφορά τη συλλογή κεφαλαίων με προπτική ε, κέρδους και δυνατότητα μεταφοράς δικαιωμάτων μαζί με τι εθνικέ εποπτικέ αρχέ, εξετάζουμε κάθε περίπτωση ξεχωριστά με κάθε προσφορά σε αυτών των νομισμάτων εξετάζουμε είναι χρηματοστικό μέσο ή όχι και από τη στιγμή που θεωρείται χρηματοστικό μέσο εντάσσεται σε ένα ρυθμιστικό πλαίσιο. Αν υπάρχει μια πλατφόρμα που εμπορεύεται σε αυτά τα νομίσματα και αυτά ρυθμίζονται μέσω της ρυθμιζόμενης πλατφόρμας. Ακολουθεί το ερώτημα τι κάνουμε αυτές τις νέες προσφορές νομισμάτων που είναι εκτός του ρυθμιστικού πλαισίου. Κάνουμε την αξιολόγηση σαν Συμβούλιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε να εκφράσουμε άποψη. Δεν θέλω να πω κάτι τώρα. Υπάρχει διάκριση μεταξύ των χρηματοστικών μέσων και αυτών που δεν είναι χρηματοστικά. Είναι πολύ σημαντική αυτή η διάκριση. Και μέχρι τέλος του έτους θα βγάλουμε πόρισμα. Πρέπει να έχουμε επίγνωση ότι μέχρι τώρα αυτές οι νέες προσφορές νομισμάτων είχαν πρόβλημα να αποδείξουν τη βιωσιμότητά τους και τι συμπληρωματικά ωφέλη δίνουν σε σχέση με άλλους τρόπους συλλογής κεφαλαίου. Αν υπάρχει κάποιο πρόσθετο όφελος, ίσως θα έπρεπε να μας προβληματίζει, είναι ότι είναι ανώνυμα αυτά τα νομίσματα και αυτό το θέτουμε και στο θέμα του ξεπλήματος χρήματος, το συζητήσαμε πριν που και αυτό ίσω να είναι κάτι που πρέπει να συζητήσουμε και στην προσφορά αυτών των νέων μέσων, αυτών των νέων νομισμάτων. Δύσκολο μακροπρόθεσμα να δούμε αν θα πετύχουν κάποια από αυτά, αλλά αυτό δεν αφορά το ρυθμιστικό φορέα. Εμεί θέλουμε να δώσουμε το ρυθμιστικό πλαίσιο, ε, ούτω ώστε οι καινοτομίε να λειτουργήσουν και να ισχύουν τα ίδια πρότυπα και προδιαγραφέ και όροι, όπω και με τα παλιά μέσα. Και συμμετέχονται στην αγορά πρέπει να αποφασίσουν κατά πόσο τα νέα αυτά μέσα, τα νέα νομίσματα έχουν κάποια αξία. Τελευταίο, Α, για τη βαθμολόγηση, την Είναι σημαντικό εκεί. Να δούμε ότι θα υπάρξουν διάφορα στήματα βαθμολόγησης. Βάσει δικτών που θα σχετίζονται με τη βιωσιμότητα όσον αφορά τις υποβόσκουσες επενδύσεις. Τώρα, ο ρυθμιστικός φορέας τι μπορεί να κάνει. Να εξασφαλίζει ότι είναι οι δείκτες ε, αξιόπιστοι. Οι επενδυτέ μπορούν να βασιστούν σε αυτού. Εμεί, αριθμιστικοί φορεί, δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μόνο ένα σύστημα ή μόνο δύο. Αυτό το αποφασίζουν οι προτιμήσει των επενδυτών. Οι ρυθμιστικοί φορεί εξετάζουν την αξιοπιστία του και τι πληροφορίε δίνουν περί των επενδύσεων. Ε, πρέπει αυτοί οι δείκτε να είναι σωστοί και να μπορούν να βασίζονται οι επενδυτέ από αυτόν. Να υπάρχει αξιοπιστία. Για τα κρυπτο στοιχεία ενεργητικού. Το επενδύσαμε αυτό το θέμα το 2013 με έκθεση και γνωμοδότηση το 2014. γραφήσαμε πρόταση. Αφορούσε το ρυθμιστικό μέλλον. Επί τριών πυλών βασιστήκαν. Πρώτος, νομοθετικές αλλαγές. Ούτω ώστε ο τομέα των κρυπτονομισμάτων κυρίως να μπουν στην εντολή της οδηγίας περί πολεμή του ξεπλήματο χρήματο. Και αυτό το καλύψαμε. Συμπεριλαμβάνεται στο NMLD 5 μετά προειδοποίηση προς τον καταναλωτή. Να ξέρουν οι καταναλωτές με άλλα λόγια ότι υπάρχει έλλειψη προστασίας αν επενδύσουν σε αυτά τα κρυπτονομίσματα και τα κρυπτοστοιχεία ενεργητικού. Μετά ήθελαμε να διαχωρίσουμε τον επίσημο ρυθμιζόμενο τομέα από τον τομέα των κρυπτοστοιχείων ενεργητικού, ούτως ώστε οι τράπεζες να μην διανέμουν κρατούν και επενδύουν ε, μέσω αυτών των κρύπτο στοιχείων ενεργητικού. Αυτή η στρατηγική πιστεύω ότι είναι στέρη. Πρέπει να παραδεχτώ όμως ότι δεν λειτουργεί ως αναμενόταν. Πιο συγκεκριμένα, η προειδοποίηση για τους καταναλωτές δεν φαίνεται να εισακούγεται επαρκώ. Δεν είναι αρκετά αποτελεσματική όσον αφορά την ευαισθητοποίηση των καταναλωτών για το γεγονό ότι υπάρχει έλλειψη δικτύου ασφαλεία όσον αφορά αυτού του είδου επενδύσει. Και βλέπουμε ότι σε κάποια κράτη-μέλη οι προτάσεις για την προστασία των καταναλωτών της λιανικής μέσω σχετικής νομοθεσίας ε, είναι κάτι που προχωράει. Άρα κάτι γίνεται στην ενιαία αγορά. Και ο διαχωρισμός, η πρόταση διαχωρισμού δεν εφαρμόζεται. Είδαμε ότι σε κάποια κράτη-μέλη οι αρχές αδειοδότησαν συναλλαγές σε κρυπτονομίσματα σαν ιδρύματα πληρωμών. Μπορεί φορέας που ε, πολύ ε, νόμιμα συστήματα πληρωμών και κρύπτο στοιχεία ενεργητικού να πλησιάσει τον πελάτη. Πρέπει να το εξετάσουμε αυτό το θέμα και να αναθεωρηθεί η προτινόμενη προσέγγιση. Δεν έχει οριμάσει στο μυαλό μου το θέμα για να μπορέσω να προτείνω κάτι. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας ρωτήσω για την καταπολέμηση του ξεπλήματος χρήματος. Τα εξής τρία. Πρώτον, για τη γενική αναγνώριση ότι οι πόροι δεν επαρκούν. Θέλω να θυμίσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε το Σεπτέμβριο μια σειρά μέτρων για ενίσχυση των πόρων ιδιαίτερα ακριβώς για να υπάρξει καλύτερος συντονισμός ε, στο έργο των ε, αρχών σας. Φαντάζομαι ότι θα τα έχετε μάθει αυτά που εξήγηλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αρκών αυτά ε, μήπως το Κοινοβούλιο θα πρέπει να προβληματιστεί σοβαρά για κάποια πρωτοβουλία να ενισχύσει το οργανόγραμμα που έχει ε, προβλέψει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ε, συντονίζονται οι διάφορες υπηρεσίες σας στην καταπολέμηση του ξεπλήματος. Δεύτερη ερώτηση. Κάτι που αναγνώρισε και είναι πολύ σημαντικό ο κύριος Ενρία, που είναι ο ρόλος των Ηνωμένων Πολιτειών εν προκειμένου. Είναι προφανές ότι υπάρχει μια κουλτούρα καταπολέμησης του ξεπλήματος ε, που είναι πολύ πρόσφατη, λίγα χρόνια, ας είμαστε ειλικρινείς, ξεκίνησε αυτό, για να καταπολεμηθεί το οργανωμένο έγκλημα, το διεθνές, σε πολλές δραστηριότητες, αλλά κυρίως στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Ερωτώ λοιπόν, εμείς βρισκόμαστε σε άμεση συνεργασία στενή και συντονισμό με τις βορειοαμερικανικές αρχές, διότι όλοι γνωρίζουμε ότι επηρεάζουν τα παγκόσμια οικονομικά και μάλιστα με τεράστιο τρόπο, πολύ μεγαλύτερο από τις δικές μας αρχές. Έχουμε πολύ συγκεκριμένες εμπειρίες με τράπεζες που χρειάστηκε να κλείσουν, όπως και εσείς αναφέρατε προηγουμένως, ακριβώς γιατί έτσι αποφάσισαν οι ΗΠΑ σε μεγάλο βαθμό. Και θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω και το εξή. τρίτη ερώτηση. Η πρακτική των ευρωπαϊκών τραπεζών που άρχισαν να εργάζονται πολύ σοβαρά κατά την άποψή μου στο συγκεκριμένο. Γιατί όλες οι τράπεζες τώρα έχουν πολύ ισχυρά τμήματα για να αναλύουν ε, την προέλευση των χρημάτων. Υπάρχει συντονισμός ε, ε, καλών υβέλτιστων πρακτικών και συνεργασία για να φτιάξουμε ένα εγχειρίδιο, ένα κώδικα συμπεριφορά και διοντολογία. Και μια τελευταία ερώτηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπέζων ε, ε, ε, έρευνα για τις δραστηριότητες της Bank στη Λετωνία. Το ψάξατε και πού καταλήξατε. Και πώς βρέθηκαν όλα αυτά τα λεφτά, τεράστια ποσά, από πού έρχονται. Προφανώς για ξέπλυμα ήρθανε, αλλά από πού. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η πρόταση της ε, Κομισιόν ε, περιέχει 10 επιπλέον ειδικού ε, για το ξέπλυμα χρήματο και με ρωτάτε τώρα εάν επαρκούν. Ε, θεωρούμε ότι είναι το ελάχιστο από πλευρά πόρων για να κάνουμε κάτι, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι 12 άτομα για το ξέπλυμα χρήματο σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν είναι κάτι το εξωφρενικό. Όσον αφορά την συνεργασία με τη ΣΥΠΑ, βεβαίως υπάρχουν πίνακες, ε, ε, υπάρχουν και φορείς, ε, όπως χάρη η σχετική task force, όπου συνεργάζονται οι εποπτικές αρχές. Όμως, παρόλα αυτά, η συνεργασία δεν είναι αυτή που θα μπορούσε να είναι. Θεωρούμε ότι σε κάποιες από τις περιπτώσεις που είδαμε πρόσφατα οι ευρωπαϊκές αρχές ε, δεν ε, είδαν τα όσα έπρεπε να γίνουν. Γι' αυτό καλωσορίζω και την πρόταση της ε, Κομισιόν που σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή θα έπαιζε και ένα ρόλο επαφής με τρίτες χώρες για αισθήματα ξεπλήματος χρήματος. Για την περίπτωση της Λετωνίας λάβαμε ένα αίτημα από την Κομισιόν να ερευνήσουμε ζητήσαμε πληροφορίες από τις αρμόδιες αρχές. Τις λάβαμε την προηγούμενη εβδομάδα και τώρα τις αξιολογούμε. Ευχαριστώ. Thank you. Σας ευχαριστώ. Δεν βλέπω ούτε τον κύριο Φόξ ούτε την κυρία Μπέρες, οπότε θα περάσουμε στο Catch the Eye. Μάλλον έχω και ένα πολύ συγκεκριμένο ερώτημα. Μια που έχουμε την ευκαιρία εδώ να έχουμε και τον Ashley Fox με τον οποίον θα συζητήσουμε και αύριο για την ε, χρηματοδότηση της ανάπτυξης. Λοιπόν, για την αρχική προσφορά σε νομίσματα. Κάτι το οποίο βεβαίως σχετίζεται με αυτό το οποίο συζητούσε ο Ανδρέα πριν. Εγώ έχω μια πιο επιφυλακτική θα έλεγα προσέγγιση, οπότε θα ήθελα να ρωτήσω και τον Στίβεν και τον Ανδρέα ε, για την πρόταση αυτή περί κάποιων τροπολογιών για να περιληφθεί και η αρχική προσφορά σε νομίσματα στο πλαίσιο του κανονισμού. Uh, ε, πρώτα απ' όλα, η προσωπική μου άποψη δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρξει κάποιο συνδυασμό ε, του crowdfunding. Ε, μπορούμε να τα δούμε ξεχωριστά τα δύο ζητήματα και για το ζήτημα των αρχικών προσφορών σε νομίσματα. Πρέπει να γνωρίζουμε πως κάποια από αυτά είναι μέσα χρηματοδότησης ενώ άλλα όχι και εκεί πέρα ακριβώς εστιάζουμε με τις εθνικές ε, ρυθμιστικές αρχές. Όταν είναι ένα μέσο χρηματοδότησης δεν θέλουμε να έχει κάποιο προνομιακό καθεστώς αλλά ούτε και ένα χειρότερο καθεστώς. Θα πρέπει να υπάρχουν ίσοι όροι ανταγωνισμού με τα υφιστάμενα μέσα χρηματοδότησης. Δεν υπάρχει κάποιος λόγος ε, ούτε είναι πιο επωφελή για την ε, κοινωνία ή την οικονομία από τα παραδοσιακά χρηματοδοτικά μέσα. Αυτή είναι η βασική προσέγγιση της ΕΣΜΑ για το crowdfunding. Ήδη έχω κάνει κάποια σχόλια για το ποιο θα είναι ο καλύτερος τρόπος εποπτείας είτε σε ευρωπαϊκό είτε σε εθνικό επίπεδο. Γενικότερα θα έλεγα ότι υπάρχει μια σαφής συζήτηση για το εάν θα πρέπει να αρχίσουν να ρυθμίζονται αυτές οι δραστηριότητες ή εάν θα υπάρξει κάποιος διαχωρισμός. Μέχρι τώρα ήμουν σε αυτούς που έλεγαν εντάξει ας αφήσουμε αυτόν τον κλάδο να είναι να αναπτυχθεί η καινοτομία αρκεί να υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες για τους ε, καταναλωτές ε, και να υπάρχει ένας σαφής τρόπος να αποφεύγεται η διάδοση στον τομέα που ρυθμίζεται. Αλλά όπως είπαμε, θεωρώ ότι αυτό δεν λειτουργεί όπως αναμέναμε και στον τομέα επίσης του crowdfunding ε, ακούμε συνεχώς για τράπεζες ή ε, πελάτες ε, των οποίων δεν τους θεωρούν επαρκώς αξιόπιστους αλλά παρέχουν κάποια υποδομή πληρωμών σε αυτούς οπότε η διασύνδεση είναι αρκετά έντονη και γύρονται κάποια ζητήματα προστασίας των καταναλωτών. Και για να είμαι ειλικρινής, δεν το παρακολουθώ το θέμα πολύ στενά, αλλά πρέπει να ξαναδούμε αυτήν την ε, διαφορετική προσέγγιση. Καθώς νομίζω έχει ξεπεραστεί από τις εξελίξεις ε, στην αγορά και τις πρωτοβουλίες που έχουν λάβει κάποιες αρχές. Πρέπει λοιπόν να δούμε κλάδους ε, στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Ναι, ε, σας ευχαριστώ. Αύριο εξετάζουμε τις τροπολογίες, δεν ψηφίζουμε, ναι, κανένα λάθος. Οπότε έχουμε λίγο χρόνο ακόμα. Περβάνω Περές. Ευχαριστώ πολύ. Ζητώ συγγνώμη τους τρεις προέδρους ε, ήμουν παρούσα σε όλη τη ε, διάρκεια ε, των παρουσιώσεων σας, αλλά εξ αποστάσεως πήρα όλα όσα είπατε. Είχα μια άλλη υποχρέωση. Για το ξέπλυμα. Χαίρεστε όλοι με την πρόταση, για την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και η EBA τώρα είναι πιο καλά εξοπλισμένη. Έχω μια ερώτηση και προς τους τρεις σας. Δεν βλέπετε εδώ κανένα πολιτικό κίνδυνο Δηλαδή να υπάρξει πολιτική συμφωνία για το ξέπλυμα, αλλά όχι για το πώς θα εφορμαστούν ε, στην πράξη οι νέες ρυθμίσεις. Δηλαδή, αν προχωρήσουμε στην πολιτική συμφωνία, αλλά αν δεν έχουμε τίποτα για τη σύγκληση, για τα στρέστες, για τη διακυβέρνηση και για τους επιτόπιους ελέγχους, τι να την κάνουμε την πολιτική συμφωνία. Θα είναι διακοσμητική αυτή η μεταρρύθμιση. Δεύτερη ερώτηση το πεδίο εφαρμογή των ε, τεστ αντοχής, των stress test. Και εκεί πρόκειται ε, να χρησιμοποιηθεί αρχή της αναλογικότητας και να εφαρμοστεί, δηλαδή ε, να ελεγχθούν μόνο οι σημαντικές εταιρείε, τα ιδρύματα ή το σύνολο. Και μάλιστα όλα αυτά να δημοσιευθούν. Εν πάση περιπτώσει, πώς θέλετε να βλέπετε να δημοσιεύονται τα αποτελέσματα. Και τέλος, για το Brexit. Πώς να το πω. Είδαμε με το θέμα των επενδυτικών εταιριών ότι μπορεί να υπάρξει ένας κίνδυνος έτσι, ε, τσαπατσουλιάς, κάποιας ε, πλημελούς και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βρεθεί μεταξύ ε, σφύρας και άκμονος. Όταν φτιάξαμε το MIFID δεν σκεφτήκαμε ότι το 80% της αγοράς θα βρισκόταν σε τρίτο ε, κράτος και το σύστημα των κλάδων ε, ε, θα έδινε ένα διαβατήριο, ας πούμε, χωρίς να υπάρχει σύγκληση. Μήπως θα πρέπει λίγο με την ησυχία μας να το σκεφτούμε και να ξαναγράψουμε την περίφημη τρία 3 που περιμένουμε. Αυτή είναι μια ερώτηση για τον Στίβεν Μαγιόρ. Διάβασα με πολύ μεγάλη προσοχή την επιστολή σας και τη σχολιάσαμε ε, επί μακρόν επίσης και σχολιάστηκε ευρύτερα. Μας λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, α, χαλάσατε το μοντέλο που προτείναμε εμείς, που ήταν ένα αμυγές ε, μοντέλο ισοδυνάμων και τώρα πηγαίνετε σε κλαδικές ρυθμίσεις. Γι' αυτό σας λέω ότι είμαστε στριμωγμένοι. Και δεν είναι τέλεια αυτή η ρύθμιση που έχει βρεθεί. Μήπως λοιπόν χρειάζεται να καθίσουμε λίγο να το σκεφτούμε, να αναλύσουμε την κατάσταση και με την ησυχία μας να προχωρήσουμε σε γερή νομοθεσία παρά ε, τώρα με τρόπο επιπόλαιο να φτιάξουμε κάτι. Δεν λέω ότι είναι επιπόλαιοι οι νομοθέτες, αλλά καλύτερα να έχουμε μια MIFID 3 έτσι πιο γερή, πιο στιβαρή παρά κάποιες επιδιορθώσεις. Okay, uh, on email you ask... Για το email ε, ρώτησες αν υπάρχει κάποιος κίνδυνος να κινηθούμε προς ευρωπαϊκές διευθετήσεις χωρίς ε, να έχουμε πιο μακροπρόθεσμε ρυθμίσει. Υπάρχει σύμφωνα με ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διαμαρτυρήθηκε σοβαρά όσον αφορά τα προβλήματα, όσον αφορά την επιβολή των διαφόρων κανόνων και να υπάρχει ένας όγκος ε, ρυθμίσεων στον τομέα αυτό. Εδώ θα υπάρχουν τομεί όπου θα υπάρχει μια ανάγκη να ακολουθηθούν διαφορετικέ εφαρμογές των κανόνων τα διάφορα κράτη-μέλη, πραγματικά πρόβλημα. Αλλά το θέμα για μένα είναι ότι αυτοί οι πολιτικοί κίνδυνοι θα πρέπει να αναλυθούν κάποιο να του αναλάβει. Διότι πρέπει να έχουμε πιο ολοκληρωμένη ε, ευρωπαϊκή απάντηση, εν πάση περιπτώσει. Και αυτή τη στιγμή πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την ισχύουσα νομοθεσία σε αναφάση δοκιμέ αντοχή, τα stress test. Να διευκρινίσω κάτι. Η δική μα δοκιμή έχει σαν στόχο 48 ε, τράπεζες φέτος, διασυνοριακούς φορείς, τους μεγαλύτερους επίσης οργανισμούς. Και θέλουμε αναλογική δοκιμή αντοχών που είναι κάτι χρήσιμο και για άλλα είδη φορέων. Η δημοσίευση των αποτελεσμάτων. Είμαστε πολύ θετικοί. Χρειάζεται να δημοσιεύονται αποτελέσματα. Η αγορά εκτιμά πολύ την αποκάλυψη των στοιχείων, όμως μετά τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων φέτος θα προσπαθήσουμε να εκφράσουμε κάποιες απόψεις και σκέψεις. Τι κάνουμε τώρα, δημοσιεύουμε τα απορίσματα, αλλά το τελικό πτωτικό αποτέλεσμα είναι διαθέσιμο στο τέλος της διαδικασίας αξιολογήσεως μερικούς μήνες μετά. Άρα υπάρχει χρονική υστέρηση και πρέπει να βρούμε άλλο τρόπο να συνοδεύουμε τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων με τα εποπτικά αποτελέσματα της επενδυτικής επιχειρήσης. από την πλευρά μου προτείναμε ένα πλαίσιο εναρμόνισης της προληπτικής αντιμετώπισης των επενδυτικών εταιριών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό ήταν αποτέλεσμα μακρού προβληματισμού. Θεωρούμε ότι το προτινόμενο πλαίσιο είναι στέρεο και θα βελτιώσει την κατάσταση που τώρα είναι κατακαιρματισμένη σε κράτη-μέλη. Σίγουρα θα υποστηρίξουμε μία πρόοδο προς αυτή την κατεύθυνση. Λοιπόν, εν πρώτης, το θέμα του IML. Βέβαια, αυτό έχει ύψη την προτεραιότητα συζητήσεις. Ναι, το ξέπλυμα του χρήματος και είναι και το πιο γενικό θέμα που έχουμε. Είναι το θέμα της επιβολής των μέτρων. Έχουμε πολλούς κανονισμούς σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Αλλά την ενδεδειγμένη φροντίδα για τη σωστή εποπτεία και εφαρμογή είναι κάτι το οποίο είναι προφανώς όσον αφορά την καταπολέμηση του του χρήματος αλλά είναι και κάτι που αποτελεί πραγματικότητα όλο και περισσότερο. Συμφωνώ μαζί σας. Καλό να ρυθμίσουμε το πρόβλημα του ξεπλήματο χρήματος. Υπάρχει γενικότερο θέμα το οποίο χρήζει αντιμετωπίσεω. Να εξασφαλίσουμε καλύτερη εποπτεία και το ρόλο των ευρωπαϊκών ε, αρχών που θα κινούνται μέσω εποπτικής συγκλήσεω. Πρέπει να προχωρήσουμε σε αυτό. Για να είμαστε ειλικρινεί, όπως το είπαν και οι συνάδελφοι. Είναι και θέμα πόρων. Κάθε φορά που σε ευρωπαϊκό επίπεδο δίνονται εντολές και ανατίθενται εξουσίες και καθήκοντα σε ευρωπαϊκούς φορείς, αν διατίθενται οι κατάλληλοι πόρια αυταπατώμεθα. Κοιτάξτε το θέμα της βιωσιμότητας που αναφέρθηκε επανειλημμένα ήδη. Μακροσκελής κατάλογος καθηκόντων, σχεδίων δράσεως κλπ. Αλλά πόροι τίποτα μέχρι τώρα. Άρα εμείς τι να κάνουμε. Άρα υπάρχει ένα γενικό θέμα σοβαρότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο και προσοχής που πρέπει να δοθεί όσον αφορά την εποπτεία και εφαρμογή. Όσον αφορά τις δοκιμές αντοχής, εν συντομία, είναι σημαντικό να υπάρχει ευελιξία για τον καθορισμό της βάσης των δοκιμών αντοχής. Βλέποντα τον ασφαλιστικό τομέα, Φερρυπίν, άλλαξαν οι κίνδυνοι με την πάρα των ετών και το είδο των δοκιμών αντοχή πρέπει να προσαρμοστεί δεόντω. Παραδείγματο χάρη, πριν από δύο χρόνια, βασικό θέμα ήταν τα χαμηλά επιτόκια. Και είναι με ειλικρινή, δεν ήταν τόσο μεγάλο πρόβλημα για του μεγάλου ομίλου στην Ελλάδα. Περισσότερο για μεσαίου μεγέθου και μικροτέρου μεγέθου επιχειρήσει, που αν κατέρεαν συλλογικά μπορούσαν να τεθεί θέμα σταθερότητα. Έπρεπε να ξεπεράσουμε του μεγαλύτερου ομίλου. Φέτο κάνουμε με 42 μεγαλύτερου ασφαλιστικού ομίλου στην Ευρώπη τι δοκιμέ αντοχή στον ασφαλιστικό τομέα. Επικεντρωνόμεθα επί του ενδεχομένου τη αυξήση των αποδόσεων, φυσικών καταστροφών κλπ. Ε, πρέπει να έχουμε ευελιξία. Η δημοσίευση είναι πάρα πολύ σημαντική, χρειάζεται μεγαλύτερη διαφάνεια. Ευτυχώ στον τομέα των συντάξεων, μάλλον δυστυχώ στον τομέα των ασφαλίσεων ε, δεν έχουμε την εντολή που έχουν συνάδελφοι τη Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή να ζητήσουν δημοσίευση. Στου συμμετέχοντε στι στις δοκιμέ αντοχών, ζητούμε από αυτού να δημοσιεύσουν τα δικά του αποτελέσματα. Δεν μπορούμε να το επιβάλλουμε, δεν έχουμε την εξουσία. Θα ήταν θεμελιώδη αναθεώρηση που θα γίνει να έχουμε αυτή την εξουσία που ήδη έχουν οι συνάδελφοι του τραπεζικού τομέα. Λοιπόν, εν συντομία, όσον αφορά τα θέματα των επενδυτικών εταιριών και του MIFID και MIFIR. Είχαμε απευθύνει μια επιστολή στον αντιπρόεδρο Ντομπρόφσκης ε, για το θέμα του MIFID 2, MIFIR και για την πλευρά των επενδυτικών εταιριών και καταλήξαμε στο εξής. Έτσι όπως λειτουργεί ο κανονισμός μέχρι στιγμής δεν έχει λάβει υπόψη το ότι υπάρχει μια αγορά με μεγάλη ρευστότητα δίπλα και πρέπει να έχουμε ίσους όρους ανταγωνισμού και βεβαίως οι επαφές με αυτή τη μεγάλη αγορά να γίνονται με τις ίδιες ε, προδιαγραφές όπως παραδείγματος χάρη επενδυτικές εταιρείε. αν δείτε άλλα νομοθετήματα, αυτό ρυθμίζεται σωστά, αν δείτε το Ινοσέκα, τον ΕΜΙΡ και τα λοιπά, έχουμε προβλέψει τις ε, τρίτες χώρες, αλλά όχι σε αυτόν τον ε, κλάδο. Και το πρόβλημα εδώ πέρα είναι ότι τα περισσότερα στοιχεία για τις τρίτες χώρες καθορίζονται στο εθνικό επίπεδο και αυτό σημαίνει ότι έχουμε πολλές ε, διαφορές και κινδύνους όσον αφορά τους ίσους όρους ανταγωνισμού. Βεβαίως δεν είναι δική μου δουλειά να αποφασίσω το τι θα κάνουν οι συνομοθέτες. Ε, δικαίως λέτε ότι ε, δεν υπάρχει μια εύκολη λύση. Ε, πρέπει να ρυθμιστούν διάφορα ζητήματα πριν το πετύχουμε. Σας ευχαριστώ κυρία Γουλφ. Ο κύριος Γουλφ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριοι για τα σχόλιά σας. Έχω ένα λεπτό μόνο, οπότε θα ξεπεράσω τα πρακτικά και θα επικεντρωθώ στο πέμπτο σημείο που αναφέρεται, αυτό του Brexit. Τον Μάρτιο η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο κατέληξαν σε μια συμφωνία και αυτή η συμφωνία έλεγε ότι οι κανόνες της Ένωσης ε, και για τα χρηματοπιστωτικά θα συνεχίσουν να ισχύουν μέχρι την 31 του 2020. Σύμφωνα με το σχέδιο Checkers ε, της Βρετανικής κυβέρνησης επιβεβαιώνεται ότι ισχύει αυτή η συμφωνία και ότι θα συνεχίσουν να έχουν το διαβατήριο οι Βρετανικές εταιρείε μέχρι την 31 του 2020 και θα πρέπει να συνεχίσουν να συμμορφώνονται με τους κανονισμούς ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Νομίζω είναι σαφές αυτό. Δεύτερον, τώρα έχει ξεκαθαρίσει ότι ο κύριος Μπαρνιέ και ο πρόεδρος Τούσκ έχουν πει ότι μια συμφωνία Καναδάς συν συν συν ε, προσφέρεται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εξακολουθείτε να επιβεβαιώνετε ότι θα ισχύει η προθεσμία της 31ης 12 του 2020 ή δεν έχει ξεκαθαρίσει αυτό μέχρι στιγμής και Τέλος, θεωρώ πως οι αγορές και οι επιχειρήσεις ε, θα είναι πολύ ευγνώμονες για την ψύχρεμη αντιμετώπιση σας της, ε, του πώς θα διεξάγονται οι συναλλαγές ε, κατόπιν γιατί βεβαίως είχα εργαστεί πάνω από 15 χρόνια στο City πάνω στον τομέα αυτόν. Το γεγονός λοιπόν ότι προετοιμάζεται ένα μνημόνιο για την περίπτωση που δεν υπάρξει συμφωνία για το Brexit. Ε, σημαίνει ότι μπορούμε να πούμε ότι εάν έχουμε Brexit χωρίς συμφωνία θα ε, καταλήξουμε κάπου σχετικά γρήγορα για να ηρεμήσουν και οι αγορές. Σας ευχαριστώ. Κοιτάξτε, να ξεκινήσω από το τελευταίο. Το μνημόνιο όπως έχουμε με πολλές ε, τρίτες χώρες, τα συζητήσαμε και στην ε, ακρόαση και όπως είπαν ε, και οι συναδελφοί Γκάμπριελ και Ανδρέα, έχουν τις ίδιες απόψεις που θα πρέπει να έχουμε μέχρι το Μάρτιο και έχουμε ήδη καθορίσει εσωτερικά και την θέση μας ως 27 της Ένωσης. Βεβαίω κάποια στιγμή θα έρθουμε σε επαφή με τους συναδέλφους ε, του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά ε, όπως είπε και ο Ανδρέα πρέπει να είμαστε αρκετά αυστηροί, γιατί εάν δεν υπάρξει αυτό το μνημόνιο και πρέπει να το γνωρίζουν ε, αυτό οι συμμετέχοντες στη αγορά, είναι θέμα του αν θα υπάρχει εγκαίρος. Τώρα δεν είμαι εγώ κατάλληλο για να κρίνω το θέμα της νομιμότητας των διαφόρων προτάσεων, οπότε δεν θα σχολιάσω. Αυτό το οποίο λέω πρακτικά είναι ότι αν υπάρξει κάποια μεταβατική συμφωνία, αυτό ε, σημαίνει ότι θα υπάρχουν κάποιες ε, προβλέψει σχετικά. Αλλά δεν θα πω τίποτα περισσότερο, ούτε θα προβλέψω το τι θα γίνει στις πολιτικές διαπραγματεύσεις. Ο Πρόεδρος, έτσι κι αλλιώς οι όροι που ισχύουν για τη μεταβατική περίοδο είναι σαφέστατοι, το κείμενο είναι δημόσιο, υπάρχει συμφωνία ε, ε, Βασιλείου Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν υπάρχει τίποτα. Και ελπίζουμε να έχει και θετική έκβαση η τελική φάση των διαπραγματεύσεων για να ρυθμιστούν όλα και η μεταβατική περίοδος και η επόμενη. Εναπόκειται τώρα στην κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου να ε, λύσει τα ε, κρεμή ζητήματα με τρόπο θετικό και σύμφωνα με τις αρχές μας. Ωραία. Μπορούμε να ολοκληρώσουμε λοιπόν αυτό το σημείο της ημέρης της διάταξης και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Στίβεν Μαγιόρ, τον Ανδρέα ε, Ενρία και τον Γκάμπριελ Αρτίνο. Ήταν πάρα πολύ ζωντανή, ενδιαφέρουσα όσο και χρήσιμη η συζήτηση αυτή. Ε, συνεχίζεται βεβαίω η συνεργασία μας μαζί σα. Βρήκαμε κάποια σημεία που χρειάζονται δουλειά. Ο διάλογος επίσης συνεχίζεται και είναι ουσιώδης. Ευχαριστούμε πολύ και περνούμε στο επόμενο θέμα όπου θα προεδρεύσει ο Πέτερ Σίμων, αντιπρόεδρος μας, και προηγουμένως πρέπει να σας πω ότι η ψηφοφορία για τις οικονομικές πολιτικές της Ευρωζώνης αναβάλλεται. Είχε προβλεφθεί για αύριο το θέμα αυτό. Αναβάλλεται η αυριανή ψηφοφορία. Σας ευχαριστώ. Äh, äh, Αγαπητοί συνάδελφοι, ο κύριος Σίμων, είμαστε στο σημείο 7 και 8, δύο εκθέσεις μαζί θα συζητήσουμε, διασυνοριακή κατανομή των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, είναι το θέμα 7 και το 8, διευκολύνοντας τη διασυνοριακή κατανομή των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων. Και στις δύο εκθέσεις είναι συγκεκριτή ο κύριος Βολφ Κλίντς, στον οποίο δίνω αμέσω το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Και τα δύο νομοθετικά ε, κείμενα θα σχολιάσω από κοινού. Είναι οδηγία και κανονισμός. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε μια πρόταση για ε, διευκόλυνση, προώθηση και εμβάθυνση της ε, κεφάλαια αγορά για να διευκολυνθούν οι διασυνοριακέ κατανομέ των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων. Προ το σκοπό αυτό έχουμε δύο οδηγίε για το IFM και ο ΣΕΚΑ ε, που πρέπει να αλλάξουν και δύο κανονισμοί. Το Συμβούλιο στη θέση του για το θέμα αυτό έχει ήδη καταφέρει ευρεία συμφωνία και έχει κάνει προτάσεις, τροποποίησεις που σε μεγάλο βαθμό με βρίσκουν σύμφωνο για να επιταχυθούν οι διαπραγματεύσει στο τριμερή διάλογο, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο μέχρι να τελειώσει η θητεία. Εκεί όπου συμφωνώ με το Συμβούλιο και μπορώ να δεχτώ τη θέση του, δεν έχω κάνει νέε τροπολογίες και έχω συμφωνήσει με τη θέση του Συμβουλίου. Παράδειγμα, όταν τα κράτη-μέλη στο μέλλον δεν, απαιτούν, δεν επιτρέπεται να απαιτούν ε, φυσική παρουσία ε, μιας επενδυτικής εταιρείας στην επικράτειά τους, έχω ευθύσει την πρόταση του Συμβουλίου. Υπάρχουν τρεις τομείς όπου δεν μπορώ να συμφωνήσω ακριβώς ούτε με το Συμβούλιο ούτε με την Επιτροπή, είμαι κάπου στη μέση και θα ήθελα σύντομα να σας τα παρουσιάσω. Ο πρώτος τομέας αφορά το λεγόμενο pre-marketing, δηλαδή πριν την ε, αγορά. Ποια, ε, ε, ποιος είναι ο ορισμός και πώς διαμορφώνεται το pre-marketing. Έχω κάνει την εξή πρόταση. Κατά την άποψή μου, τα επενδυτικά ταμεία μπορούν να κάνουν αυτές τις δραστηριότητες απρόσκοπτα στο βαθμό που αφορά εναλλακτικές μορφές συλλογικών επενδυτικών ταμείων που δεν έχουν ακόμα άδεια ε, ή ε, έδρα στην ε, λόγο χώρα. Στα αγγλικά αυτό λέγεται established. Την έκθεση την έχω γράψει και στα αγγλικά. Και η αγγλική μετάφραση για μένα είναι το, το πρωτότυπο κείμενο, το αρχικό κείμενο που ισχύει έτσι και το, ο, ο γιατί έχω διαπιστώσει ότι στη γερμανική μετάφραση μετά υπάρχουν ε, κάποιες ασάφειες. Γι' αυτό αναφέρομαι στο αγγλικό κείμενο. Τα γραφειοκρατικά εμπόδια ε, θα πρέπει να αρθούν ε, πάντα πριν την κυκλοφορία στην αγορά, έτσι ώστε εκείνοι που προσφέρουν τις υπηρεσίες να ε, βολιδοσκοπήσουν το ενδιαφέρον των επενδυτών χωρίς βαριές διαδικασίες και να υπάρχει μια διαδικασία ανταλλαγής έτσι, πληροφοριών ping-pong πριν εγκατασταθούν ή πάρουν άδεια επίσημα. Βεβαίως, συμφωνώ με την Κομισιόν και το Συμβούλιο ότι το pre-marketing δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για να ε, παρακάμπτονται οι κανόνες κυκλοφορίας στην αγορά. Και εδώ έχω υιοθετήσει την ε, διατύπωση του Συμβουλίου που γίνεται, ε, κάνει λόγο για περίοδο 18 μηνών όπου να είναι δυνατόν να κυκλοφορεί το προϊόν ε, στην αγορά εφόσον τηρούνται οι όροι που ορίζουν τις δραστηριότητες pre-marketing. Όλες αυτές θα πρέπει βεβαίως ε, εσωτερικά να ρυθμίζονται και μετά από αίτημα των εποπτικών αρχών να διατίθενται και να, και να διαβιβάζονται. Ε, το δεύτερο αφορά την λήξη των προσφορών των επενδυτικών ταμείων που κυκλοφορούν στην αγορά και απόσυρσή τους αν θέλει κάποιο να διακόψει τη δραστηριότητά του σε ένα κρατο μέλος. Προσπάθησαν το Συμβούλιο και η Επιτροπή να βάλουν αυθαίρετες ε, ε, ρυθμίσει με ποσοστά ε, από ποιο μέγεθος και μετά μια εταιρεία ή ο επενδυτής να μην επιτρέπεται πια ή αν θέλει να αποσυρθεί με διάφορα ποσοστά του συνολικού επενδυτικού όγκου του Ταμείου εάν δεν είναι μεγάλη δράση ε, σε μια χώρα να μπορεί να ε, αποσύρεται. Σας λέω, αυτά είναι αφαίρετα και πολύ δύσκολο να ελεγχθούν ως προτάσεις. Γι' αυτό επέλεξα ένα διαφορετικό δρόμο. Λέω, τα επενδυτικά ταμεία δεν θα πρέπει να επιβάλλεται να έχουν μια ε, δραστηριότητα εμπορική αν δεν τους συμφέρει πλέον. Βεβαίως θα πρέπει να προστατεύονται οι επενδυτές και τα συμφέροντά τους, ακόμα και αν η εταιρεία που προσφέρει την επένδυση αυτή ε, διακόπτει τη λειτουργία της. Άρα τα επενδυτικά ταμεία ανεξαρτήτως ε, μεγέθους να μπορούν να διακόπτουν την προσφορά τους, αλλά όπως προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει ε, κάθε επενδυτής να έχει τη δυνατότητα να εξαγοράζει το προϊόν. Αν θέλει να παραμείνει Ε, ο, ε, ο καταναλωτής παύλα επενδυτής θα πρέπει να συνεχίσουν οι εταιρείε αυτές να παρέχουν πληροφορίες, να τις δημοσιεύουν και να κάνουν ό,τι προβλέπεται. Το τρίτο αφορά τα τέλη. Έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά, προεργασία ε, το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για περισσότερη διαφάνεια. Εγώ προτείνω κάποιες αλλαγέ, έτσι ώστε τα τέλη να είναι απαιτητά μόνο εάν είναι απαραίτητε και θεμητές οι εποπτικές δράσεις. Και αυτά τα θεμητά τέλη θα πρέπει να ανταποκρίνονται ε, στο πραγματικό κόστος εποπτείας που προκύπτει από τις ε, δραστηριότητες αυτές. Και κάτι άλλο που συζητήσαμε και με τους προέδρους των τριών εποπτικών αρχών, ε, να πω δύο λόγια για το PRIPS. Μας είπαν ότι στη διασυνοριακή κατανομή των οργανισμών αυτών, των επενδυτικών, θα πρέπει να δούμε και το PRIPS Kids και ε, τα ταμεία των χρηματαγορών. Μα κοιτάξτε, δεν είναι δικό μας αντικείμενο αυτό για το έγγραφο βασικών πληροφοριών των PRIPS. Ε, δεν είναι δουλειά της συγκεκριμένη έκθεσης να το συζητήσουμε με τους κοιόδης ηγητές και να έρθουμε σε επαφή με το Συμβούλιο και την Επιτροπή. Αν καταλήξουμε όλοι Ε, ότι θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με το, με το ε, έγγραφο βασικών πληροφοριών των ΟΣΕΚΑ ή των ΠΡΙΠΣ και αν θα πρέπει οπωσδήποτε αυτή τη στιγμή να αντικατασταθεί το ένα από το άλλο γιατί δεν είναι ικανοποιητικό. Εν πάση περιπτώσει, αν συμφωνήσουμε ε, ότι είναι σκόπιμο να ασχοληθούμε και στη συγκεκριμένη έκθεση με αυτό, Καλώς. Απλώς εγώ δεν θέλω να καθυστερήσουμε εξ αυτού του λόγου και μετά να στριμωχθούμε και να μην ολοκληρώσουμε το θέμα ε, με σωστό τριμερή διάλογο ε, πριν το τέλος της παρούσης θητείας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, Βόλφ, για το ΕΛΚ, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να συγχαρώ τον συνάδελφό μας για το έργο του που ήταν έξοχο και για μας αποτελεί μια καλή βάση εργασιών με κάποια συμπληρώματα ή ενδεχομένως τροπολογίες. Να αναφέρω κάποια στοιχεία. Δεν είμαστε αντίθετοι εκ των προτέρων. Το pre-marketing, πριν διατεθούν στο εμπόριο τα προϊόντα, να διευρυθεί όσον αφορά τα εφιστάμενα ταμεία, αν το επιθυμούν, αν θέλουν να δώσουν πληροφορίες όσον αφορά τις προθέσεις που έχουν, να ανοιχτούν και σε άλλες χώρες. Στόχος αυτού του κειμένου είναι να αναπτυχθούν οι διασυνοριακές επενδύσεις. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε για να τις ενθαρρύνουμε αυτές. Θα πρέπει ό,τι μπορούμε να κάνουμε ληφθεί υπόψη. Συμφωνούμε να περιοριστεί η πρώτερη διάθεση στους εμπορευμένους, τους θεσμικούς επενδυτές και όχι στους χρήστες usage και του λιανικού εμπορίου, retail όσον αφορά το θέμα της κοινοποίηση. Τη διακοπή της κοινοποίηση αναφέρει πολύ περίπλοκο σύστημα ο εισηγητής που χρειάζομαι κάποιο χρόνο για να μπορέσω να κατανοήσω. Χρειάζεται να επικοινωνήσω μαζί του. Εκ των προτέρων δεν είμαι αντίθετο. Θα θέλαμε όμως να καταλάβουμε καλύτερα. Οι αρχές βάσει των οποίων μπορεί κανείς να παραιτηθεί από την υποχρέωση να δημιουργήσει φυσικό ε, φορέα σε κάποιο, στο φιλοξενούν ε, κράτος μέλος φαίνεται ελκυστικό όρος υπό την προϋπόθεση να δούμε ποιες είναι οι συνέπειες οι φορολογικές εξετάζοντας άλλα θέματα, άλλα χαρτοφυλάκια κάτι που θα συζητήσουμε εδώ και με την έκθεση στο CCTB ε, λάβαμε υπόψη ότι ο βασικός λόγος για τον οποίο κάποιες πολυεθνικές τρίτων χωρών δεν μπορούσαν να φορολογηθούν και να πληρώσουν φόρο στα κέρδη των επιχειρήσεων μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ενώσης είναι διότι δεν είχαν φυσική παρουσία. Φυσική εγκατάσταση, φυσική έδρα. Δεν πρέπει να διευκολύνουμε λοιπόν ε, φορο, τέτοια φοροδιαφυγή μέσω τέτοιων διατάξεων που είναι προφανώς και μία απλούστευση. Όπως και η θέλω να πω που ναι μεν δεν είναι θέμα του κειμένου που συζητούμε αλλά μήπως σε αυτή την ευκαιρία μπορούμε να ρυθμίσουμε και ένα άλλο πρόβλημα. Τον PRIPS kit που συζητήσαμε επί μακρόν με τους ε, εκπροσώπους των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών. Μήπως μπορούμε μέσα αυτού του κειμένου να καλύψουμε και αυτή την περίπτωση. Σας ευχαριστώ. Αλέν για τους σοσιαλδημοκράτες η Μαρή Ντελβό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, θα ήθελα να πω ότι καλοδεχούμενες οι προτάσεις της Κομισιόν για να διευκολύνουν την διασυνοριακή διανομή των ταμείων και να έχουν περισσότερες επιλογές οι επενδυτές. Ναι, και ελπίζουμε έτσι να μειωθούν οι διαφορές μεταξύ κράτων μελών όπου κάποια αυτή τη στιγμή έχουν πολύ ανεπτυγμένες αγορές ενώ άλλα κράτη-μέλη έχουν ελάχιστα τέτοια ταμεία διαθέσιμα. Και να ευχαριστήσω και τον Βολφ Κλίντς, ε, τον εισηγητή αντιλαμβάνομαι ότι έχει δεχτεί πολλές αλλαγές που προτείνει η Κομισιόν. Πρώτον, επειδή συμφωνεί και δεύτερον, επειδή θέλει να προχωρήσει γρήγορα το θέμα αυτό και στηρίζω ακριβώς αυτή τη διαδικασία. Για τα διάφορα ζητήματα λοιπόν πρέπει να ομολογήσω ότι δεν έχω ακόμα κατασταλάξει. Για την προεμπορία βεβαίως είναι δύσκολο να καθοριστεί η έννοια και δεν ξέρω εάν χρειαζόμαστε όλους τους όρους που προτείνει η Κομισιόν, εάν πρέπει να διαγράψουμε κάποιους. Αυτό το ομοίο μου φαίνεται σαφές είναι ότι πρέπει να περιοριστεί ε, χρονικά. Νομίζω 18 μήνες είναι μια βολική περίοδος. Για την ε, ειδοποίηση αυτή πρέπει να βρεθεί μια ισορροπία, γιατί ειλικρινά, εάν το κάνουμε πολύ δύσκολο να βγει κανείς από μια αγορά, ε, θα αποθαρρυνθούν ε, οι διαχειριστές και να μπουν σε μια αγορά. Τότε αν θέλουμε μια ζωντανή αγορά, ε, τότε δεν θα πρέπει να γίνει πολύ δύσκολη η ειδοποίηση, αλλά βεβαίως πρέπει να υπάρχει προστασία των επενδυτών και επαρκής πληροφορίες. Και έχω και μία ερώτηση. Ποιο είναι το νόημα της ειδοποίησης αν ε, ο διαχειριστής ε, θα συνεχίσει να πληρώνει τέλεια ακόμα και όταν έχει ειδοποίηση. Ε, για μένα είναι περίπλοκο αυτό το ζήτημα. Γιατί βεβαίως θα πρέπει να υπάρχει και η απαραίτητη παρακολούθηση. Και βεβαίω υπάρχει και η πρόταση της Κομισιόν να δημιουργηθεί ακριβώ αυτό το ενεργό εργαλείο για την ΕΣΜΑ και στα διάφορα ένα link προς τα διάφορα site για τα TRIPS, ε, όπως είπε και ο εισηγητής, ε, καλό είναι να ζητήσει μια λύση για την παράταση των εξαιρέσεων από το ΣΕΚΑ. Θα το παρακολουθήσουμε ενδιαφέρον και τέλος αφορά ακριβώς ε, το θέμα αυτό της άγρας πελατών και θα πρέπει ακριβώς να δούμε τι θα γίνει με αυτό. Πρέπει λοιπόν να δούμε αυτά τα ζητήματα για να προχωρήσει το ζήτημα. Ευχαριστούμε Μαρή. Άσλη για το ECR. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρόεδρε, ο κ. Κεμάλος και ό,τι ζήτησε να τον συγχωρήσετε και να διαβάσω και αυτή τη δήλωση εκ μέρους του. Το ECR συμφωνεί με την πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ξεχρονιστεί το USITS και το AIFMD. Είναι εκπληκτικό που διαβάζουμε ότι μόνο 37% του USITS και περίπου 3% του AIF είναι καταχωρημένα προς πώληση σε πάνω από τρία κράτη-μέλη. Είναι σαφέ ότι περισσότερα πρέπει να γίνουν για να ενθαρρυνθεί η διασυνοριακή διάθεση των προϊόντων usage και AIF το ECR υποστηρίζει νέα μέτρα για τη μείωση του κόστους των διαχειριστών των ταμείων να μπορούν να κινηθούν διασυνοριακά και να αυξηθεί η διασυνοριακή διάθεση ε, των ε, διαφόρων επενδυτικών ταμείων. Να αυξηθεί ο ανταγωνισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κάτι που βοηθήσει του επενδυτές να έχουν μεγαλύτερη επιλογή και καλύτερη αξία θα έχουν στα χέρια τους. Όμως πιστεύουμε ότι χρειάζεται καμία καλύτερη ισορροπία μπορεί να επιτευχθεί με μεγαλύτερα μέτρα διαφύλαξης ώστε οι λιανοπολιτές, οι τωρινοί που βασίζονται σε εσωτερικό ε, διαμεσολαβητή να, να μπορέσουν να συνεχίσουν να το κάνουν αυτό κατά τη διάρκεια τη επενδύση και θα πρέπει να υπάρχουν και άλλε δυνατότητε στου διαχειριστέ που έχουν σταματήσει να θέτουν ένα προϊόν σε ένα κράτο μέλο, θα θέλουν να συνεχίσουν να εξυπηρετούν από μακριά του επενδυτέ του αφού έχουν πάψει τι δραστηριότητε. Η γενική προσέγγιση του Συμβουλίου κάνει τεχνικέ αλλαγέ που πρέπει να υποστηρίξουμε. Όπω και ο εισηγητή, και εμεί θέλουμε αυτέ οι προτάσει να συμφωνηθούν πριν το τέλος της ε, νομοθετικής θητείας. Μια τυποποίηση της διαδικασίας κοινοποίησης είναι κάτι που απαιτείται. Αυτό διαφαίνεται και σε άλλα θέματα της ε, ενιαίας κεφαλαγοράς που επεξεργαζόμαστε. Ε, Επίκαιρε πληροφορίες, σύγχρονες πληροφορίες στο διαδίκτυο είναι κάτι που είναι σημαντικό για τις αρμόδιες αρχές και για τους επενδυτές. Βασική διάταξη είναι να απαγορεύσουμε τα κράτη-μέλη να απαιτούν φυσική έδρα στην επικράτειά τους για αυτά τα ταμεία ε, που θέλουν να διαθέσουν προϊόντα στην αγορά. Συμφωνούμε με τον εισηγητή και το Συμβούλιο για να υποστηρίξουμε αυτή την προσέγγιση. Τώρα, όσον αφορά την διάθεση εκ των προτέρων, το pre-marketing στην αγορά, συμφωνούμε με πτυχέ τη πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πτυχέ τη Γενική Προσεγγίση του Συμβουλίου και συμφωνούμε και με το σχέδιο κειμένου του εισηγητού. Θα προσπαθήσουμε ε, να υποβάλουμε τι σχετικέ τροπολογίε για να συγκεράσουμε προσεγγίσει για την πάυση δραστηριοτήτων συμφωνούμε με τι αλλαγέ που προτείνονται, αλλά δεν πιστεύουμε ότι τα NCA θα πρέπει να συνεχίζουν να εισπράττουν τέλη από τη στιγμή που έχει σταματήσει η δραστηριοποίησή του στην αγορά. Τέλο, θα θέλουμε να προσέξουμε ε, και τι προθεσμίε εφαρμογή να έχουμε μια διαδικασία λογική όσον αφορά την υλοποίηση. Πρόεδρε, ο ΣΑΙΤ προσβλέπει σε συνεργασία με τον εισηγητή και τους άλλους κοιόδης τους ε, επόμενους μήνες και σας ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Ο πρόεδρος Ασλή. Ο Σβέν Γκίγκολτ από πλευρά των Πρασίνων. Στα αγγλικά θα είμαι πάρα πολύ σύντομος πρόεδρε και σας ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Πρώτον, θα ευχαριστήσω πολύ τον Βόλφ Κλίντς για το σχέδιο έκθεσή του. Συμφωνούμε με τη διαδικαστική πρόταση. Δηλαδή να υιοθετήσουμε κάποια από τα στοιχεία στα οποία έχει καταλήξει το Συμβούλιο για να ε, υπάρχουν κάποιες πιθανότητες να ολοκληρώσουμε αυτό το θέμα ε, το συντομότερο. Δεν έχω μελετήσει ε, το φάκελο με μεγάλες λεπτομέρειες όπως και εσύ Μάντι. Ο πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή. Α, δεν μεταφράστηκε αυτό που είπατε πρόεδρε. Λοιπόν, Καλά, δεν είπα και τίποτα κακό. Λοιπόν, η πρώτη μας εντύπωση όμως ποια είναι, διαβάζοντας έτσι ακροθυγώς την έκθεσή σας, ότι κινείστε προς μία κατεύθυνση ουσιαστικά, δηλαδή αποδυνάμωση των προτάσεων για την προστασία των επενδυτών, ε, προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αποδυναμώνεται από τη μια χωρίς να ενισχύεται ε, από την άλλη, εμεί πάντα είμαστε πρόθυμοι να συζητήσουμε ό,τι θέλετε, αλλά το Κοινοβούλιο είναι πάντα υπέρ τη ισχυρή προστασία των επενδυτών. Έχουμε συμφωνήσει και σε προηγούμενα θέματα, ακριβώ για να προχωρήσουμε τελικά στην Ένωση Κεφαλαίου Αγορών. Αν δεν έχουμε ισχυρέ διατάξει σε όλα τα κρατημέλη για την προστασία των επενδυτών, δεν πρόκειται να ε, ε, προχωρήσουμε σε μια ολοκλήρωση τη αγορά που θέλουμε όλοι να δούμε για να αυξηθεί ο ανταγωνισμός ε, και ε, ε, επιλογή των επενδυτών και των καταναλωτών. Στις δικές σας προτάσεις λοιπόν δεν είδα να υπερασπίζεστε στεναρά την ενδυνάμωση και της προστασίας των επενδυτών. Προσανατολίζεστε πιο πολύ στην πλευρά της προσφοράς και όχι της ζήτησης. Άρα θα φροντίσουμε να επαναφέρουμε την ισορροπία στην προσέγγιση του Κοινοβουλίου Πάντως, όπως πάντα και στο παρελθόν, έτσι και τώρα προσβλέπουμε στην καλή συνεργασία και με εσάς κύριε Σιγητά και με όλους τους υπολείπους εδώ, συναδέλφους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ Σβέν. Ε, πρέπει να πω ότι δεν ήταν και εδώ πέρα ο άλφος από τους πράσινους. Ε, να σας πενθυμίσω. Για, για την Κούετς, όχι τους πράσινους. Α, ναι, ναι, σωστό. Τώρα δεν έχουμε εμεί σχέση με το Ιρλανδικό κίνημα ανεξαρτησίας, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, έτσι. Ναι. Λοιπόν, Περβάνς Μπερές. Ναι. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν είναι παρούσα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να πάρει το λόγο όσον αφορά το θέμα των PRIPS διότι σαν εισηγήτρια για το θέμα αυτό έχω πλήρη επίγνωση ότι έχουμε μια επικαιρότητα που δημιουργείται για το θέμα αυτό και θα ήθελα να μην ε, διασκορπιστούμε στις προσπάθειές μας να έχουμε μια συντονισμένη προσέγγιση για την εντόπιση του προβλήματος. Δεν χρειαζόμαστε κατακαιρματισμό της νομοθεσίας, δεν θέλουμε να την κάνουμε εύθραυστη. Το επιχείρημα που ακούμε είναι να λένε ότι η εφαρμογή του PRIPS ε, ήταν καθυστερημένοι, οπότε με καθυστερήσουμε έτσι περαιτέρω. Εντάξει, θεμητό αυτό, αλλά κατανοώ και την αντίθεση του usage να συμφιλιώσει ε, τα διάφορα στοιχεία. Από πλευράς νομοθέτου δεν θέλουμε μία και μοναδική γενική λύση, αλλά θέλουμε τα κατάλληλα εργαλεία που επιτρέπουν μια συγκρισιμότητα των χρηματοπιστωτικών προϊόντων που προσφέρονται στον καταναλωτή στη λογική αυτών που ήθελε να κάνει το Κοινοβούλιο. Κατόπιν πρωτοβουλία Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρέπει αυτό να το εξετάσουμε προσεκτικά και να μην το εκμεταλλευόμαστε. Κινούμενοι πολύ ταχαίως και να ακούμε όλα τα επιχειρήματα του τομέα που δεν θέλει να κάνει αλλαγές. Υπάρχουν στοιχεία των ΠΡΙΠΣ που πρέπει να αξιολογηθούν αν εφαρμόσει κυρίως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την νομοθεσία τη σχετική για τα PRIPS, συμπεριλαμβάνοντας κριτήρια κοινωνικά και περιβαλλοντικά. Αλλά ξέρω ότι επ' αυτών περιμένει τη μεγάλη μεταρρύθμιση που είναι και η σωστή εφαρμογή της ταξινόμησης. Είδα στις τροπολογίες του συγγητού κάποιες ε, θέσεις που έχουν σαν στόχο να καταργήσουν το ρόλο της ΕΣΜΑ. Θα ήθελα Μία αξιολόγηση λοιπόν όσον αφορά την έννοια των προτάσεων αυτών. Άλλη παρατήρηση. Συνέπειες της διασυνοριακής δραστηριότητας. Στα πλαίσια της αγοράς κεφαλαίων όλοι κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση. Υπάρχουν όμως κάποια μέτρα διαφύλαξης. Όπως και ο Λένα Μασούρ το έθεσε το θέμα. Αν η έλλειψη φυσικής έδρας συνεπάγεται έλλειψη φορολόγησης, τότε αυτό είναι πρόβλημα και είδαμε στον τομέα των ασφαλίσεων κάτι προσπαθήσαμε να διορθώσουμε, αλλά δεν είναι εύκολο. Ότι ασφαλίσεις είδαμε, λέω, ότι η δραστηριότητα διασυνοριακής διανομής οδηγεί σε καταστροφικές συνέπειες διότι υπάρχουν επιχειρήσεις γραμματοκιβωτίου, εικονικές, που εγκαθίστανται σε μια χώρα και διανέμουν το προϊόν τους, το χρηματοστικό προϊόν τους, άλλη χώρα, αρνούμενες πλήρες το πλαίσιο προστασίας του καταναλωτού που υπάρχει σε αυτή τη χώρα. Προτείνω αυτό να το δείτε από κοντά και να προσέξετε να λάβετε υπόψη τα μαθήματα αυτό που συνέβη στον τομέα των ασφαλίσεων. Είναι ο πρώτος τομέας όπου είχαμε διασυνοριακή διανομή προϊόντων και που ήταν και πιο ενεργή διανομή προϊόντων σε αυτό το τομέα. Σας ευχαριστούμε, Περβάνς. Τώρα έχουμε τον συνάδελφο Χάις στην διαδικασία του KHDI. Χάις, εδώ είμαι κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να συγχαρώ τον Βόλφ και θα ήθελα να κάνω κάποιες ε, παρατηρήσεις. Ε, συμφωνώ με τους ε, συναδέλφους ότι το θέμα ακριβώ αφορά το πώς θα γίνει καλύτερη η κεφάλαια αγορά, η ιστορική κεφάλαια αγορά. Και βεβαίω έχει δίκιο υπερβάνω, πρέπει να αντλήσουμε κάποια διδάγματα στην πλευρά <coughs> των ασφαλιών, μια ευρύτερη και πιο διευρυμένη αγορά είναι κάτι το οποίο όλοι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να επιτύχουμε στο πλαίσιο της Ένωσης ε, Κεφαλαίου Αγορών και βέβαια να μειωθούν οι διαφορές μεταξύ κρατών μελών. Έτσι μπορεί να γίνει αυτό. Θα ήθελα τώρα εγώ να συμφωνήσω με τον εισηγητή μας ε, του ΕΛΚΑ, τον Αλέν Λαμασούρ, τις παρατηρήσεις ε, που έκανε για το θέμα των Πρίψ και του ΚΙΔ. Ξέρω πως είπε στην αρχή αυτό το οποίο είπε η συνάδελφος, αν μπορούσαμε δηλαδή να δούμε αυτό το ζήτημα στο πλαίσιο του φακέλου. Αν δούμε τον στόχο της πληροφόρησης ε, των επενδυτών και των σχετικών ε, προσπέκτους, στόχος είναι να μην είναι υπερβολικά πολύπλοκα, αλλά εάν έχουμε δύο δυνητικά, διαφορετικά προσπέκτους, ε, δεν νομίζω ότι μας βοηθάει αυτό και δεν είναι και προς το συμφέρον των ε, μικροεπενδυτών. Οπότε ίσως είναι μια ευκαιρία να ξαναδούμε αυτό το ζήτημα. και βεβαίως ακριβώς ε, είχα απευθυνθεί στην Κομισιόν και το επεσήμανα αυτό ότι θα υπάρξει αυτή η διαφορά από το 2020 και μετά. Οπότε θέλω να ακούσω και την άποψη της Κομισιόν. Έχουν εδώ πέρα σημαντικό ρόλο να παίξουν οι αρχές, ε, αν έχουν δηλαδή αναγνωρίσει το πρόβλημα της ε, ασυνέπειας μεταξύ ε, δύο διαφορετικών προσπέκτους. Πρέπει να το έχουμε υπόψη αυτό. Έχουμε σημαντική εμπειρία και οι συγητές και οι σκιώδεις συγητές θα μπορούσαμε ακριβώς να λύσουμε αυτό το πρόβλημα διακομματικά και νομίζω αξίζει τον κόπο. Σας ευχαριστώ, Μπράιαν. Ποιος θέλει... Ε, λοιπόν, όπως ε, πρότεινε η Περβάνς ε, και Μπράιαν, να δώσω τον λόγο στον τμήματάρχη της Κομισιόν, τον κύριο Σβεν Γκέντνερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Αν επιτρέπετε, θα ξεκινήσω λέγοντα μερικά λόγια για τη δυσυνοριακή διανομή και μετά θα μιλήσω και για τα PRIPS, εφόσον πολλέ ερωτήσει σχετικέ ακούστηκαν. Με τα χαρά βλέπουμε το σχέδιο εκθέσεω. Είμαστε ικανοποιημένοι για το άκρο επικοδομητικό πνεύμα που επέδειξαν όλοι. Συμφωνούμε, είναι σημαντικό χαρτοφυλάκι αυτό, πρέπει να προωθηθεί με τη συμμετοχή όλων. Θα ήταν υπέροχο αν μπορούσαμε να ολοκληρώσουμε το θέμα της διανομής της διασυνοριακή σε αυτή τη θητεία. Θα κάνει τη διαφορά για την κατάσταση όσον αφορά τη διασυνοριακή κατανομή των πόρων, των ταμείων, συγγνώμη. Ε, τούτου λεχθέντος, έχουμε δύο θέματα που πρέπει να θέσουμε. Και με το κείμενο του Συμβουλίου και έκανε αλλαγέ στην πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρώτα απ' όλα, την, το pre-marketing, μας αρέσει η ιδέα της αρχικής διάθεσης στην αγορά, της πρώτης διάθεσης στην αγορά, το pre-marketing. Το προτείναμε σε αρχική πρωτοβουλία, αλλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Μην ανοίξουμε την πόρτα για παράκαμψη του καθεστώτος διαβατηρίου και μην δημιουργήσουμε ένα σύστημα που μπορεί να είναι πιο αδιαφανές από αυτό που έχουμε. Αυτό που θέλουμε είναι καλύτερα λειτουργούσα αγορά, αλλά και διαφανή αγορά, αγορά που μπορούμε να βλέπουμε πώς εξελίσσεται και να δούμε μαθήματα για το μέλλον. Υποστηρίζουμε αυτή την ε, ιδέα να υπάρχει μια περίοδος δηλαδή μετά το pre-marketing όπου εκεί σε αυτή την περίοδο δεν μπορείς να κάνεις τίποτα άλλο παρά marketing, διάθεση στην αγορά ή τίποτα. Τι μας προβληματίζει, ότι το παρόν κείμενο δεν έχει πρόβλεψη ούτω ώστε αυτό να ισχύει. Δεν υπάρχει υπο... πρόβλεψη για υποβολή πληροφοριών, διαφάνεια. Ο εποπτικός φορέας δεν μπορεί να καταλάβει ποιες είναι εξελίξεις. Το είπαμε αυτό και στο Συμβούλιο και πιστεύουμε ότι θα ήταν απλό και εύκολο και όχι δαπανηρό να προβλέπεται απέτηση. Δηλαδή ότι επιτακτικής περίοδου οι πάροχοι των ε, χρημάτων του, ε, του Ταμείου να δίνουν στον εποπτικό φορέα πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητε πριν από τη διάστηση στην αγορά, pre-marketing. Δεν θα σχετίζεται με τέλη, με κόστος αυτή η διαδικασία. Θα ήταν κάτι λογικό σαν να θέτει όριο ταχύτητα. Άρα όμω, αν έχει όριο ταχύτητα, πρέπει να βάζει και μια κάμερα, ώστε άμα παραβιάζει κανεί το όριο ταχύτητα, να μπορεί να επιβάσει κυρώσει. Κάτι άλλο. Για την πάυση κοινοποίηση. Η προσέγγιση του εισηγητού θα είναι δυνατότητα διαχειριστή του ταμείου να δραστηριοποιηθεί στην αγορά της χώρας ε, που, που εδρεύει. Πρέπει να προσέχουμε όμως ε, αν απομένει σημαντικό ποσό και επένδυση εκεί, προσπαθεί να περιορίσει τις αντίθετες συνέπειες για προστασία του καταναλωτού για να συνεχίζονται ε, υποχρεώσεις για ε, κοινοποίηση και να εξακολουθούν ισχύουν οι αρχές της φιλοξενούσας χώρας. Υπάρχει αντίφαση. Πρέπει να δίνουμε τη δυνατότητα να σταματάει η κοινοποίηση σε κάποιες περιστάσεις και να υπάρχει όφελο από αυτό να μην υπάρχει συμπροματική κοινοποίηση, συμπροματικό κόστο, αλλά πιστεύουμε ένθερμα ότι αυτό θα πρέπει να είναι εφικτό μόνο υπό κάποιε περιστάσει, υπό όρου, δηλαδή μόνο όταν υπάρχει περιορισμένο αριθμό επενδυτών που έχει απομείνει στη χώρα. Τι φιλοξενούσαν. Υπάρχει δυνατότητα να φύγει κανεί από, από την αγορά, να δώσει κίνητρα στου συμμετέχοντε στην αγορά, να μπουν στην, να, στους, σε κάποιου να μπουν στην αγορά, αλλά και επενδυτέ να ξέρουν ότι αν υπάρχει σημαντική βάση επενδυτών σε μια χώρα, δεν θα πρέπει να είναι πολύ εύκολο ο πάροχος να σταματήσει την κοινοποίηση. Πιστεύουμε θα ήταν καλό να έχουμε ε, όρια που έχουν νόημα. Ο ορισμός ενός ορίου ποτέ δεν είναι ακριβής επιστήμη. Συμφωνούμε από αυτού με τον εισηγητή. Όμως αυτό δεν πρέπει να μας σταματάει να προσπαθούμε να βρούμε κάτι, κάτι που βοηθάει για να δίνει κίνητρα όσον αφορά την παροχή και που προστατεύει ταυτόχρονα και τους ε, επενδυτές. Πάμε τώρα στο TRIPS. Βέβαια θέλουμε να εξασφαλίσουμε συγκρισιμότητα. Αυτή ήταν η αρχική μας προσέγγιση και στόχος, όλοι συμφωνούν. Από πλευράς των εποπτικών αρχών, τι διαπιστώσαμε, ότι είναι πρόθυμες να εξετάσουν στοχευμένες αλλαγές στο επίπεδο 2, στα πλαίσια του PRIPS, ούτως ώστε το PRIPS να εφαρμόσετε πιο εύκολα, να εφαρμόσετε και για τα μία usage. Ξέρουμε ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα για το usage κυρίως αλλά μας είπαν οι υποπτικές αρχές ευρωπαϊκές ότι μπορεί αυτό να διορθωθεί αρκετά γρήγορα, ούτω ώστε μέχρι το τέλος του επόμενου έτους θα μπορούσαμε να εφαρμόσουμε ένα έγγραφο και μόνο για όλα τα προϊόντα που εμπίπτουν στο PRIPS. Κατά την άποψή μα θα ήταν και το ιδεώδες αποτέλεσμα, τότε θα έχουμε συγκρισιμότητα, κάτι που επιθυμούν όλοι, διαφάνεια που όλοι επιθυμούμε, αλλά θα φροντίσουμε κάλυψη διαφόρων ζητημάτων που καταλαβαίνουμε ότι θα μπορούσαν να δημιουργήσουν επιπλοκές για τα ταμεία usage. Θέλουμε να ακολουθήσουμε αυτή την προσέγγιση που προτείνουν και οι ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές. Περιορισμένες στοχευμένες αλλαγές στο επίπεδο 2 και μέχρι το τέλος του επόμενου έτους ένα έγγραφο που θα μπορεί να ισχύει για όλη την αγορά και θα οδηγεί στο βέλτιστο αποτέλεσμα και για τους ε, επενδυτές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Γκέντνερ για να κλείσει. Το λόγο έχει ξανά ο εισηγητής Βολφ Κλίνς, αλλά ζητάει και υπερβάς το λόγο. Παρακαλώ. Ναι, όχι. Απλώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν απάντησε σε αυτό που ρώτησα εγώ για την προθεσμία ε, εφαρμογής. Κανονικά στο PRIPS, αν δεν απατώμε, είναι ανοιχτή η διαδικασία για το προσπέκτους, για το έγγραφο βασικών πληροφοριών και σε επίπεδο 2 πώς το κάνετε αυτό. Έχετε καμιά εικόνα για το χρονοδιάγραμμα και πώς θα το ορίσετε. Στο πρίψ υπάρχει καταληκτική ημερομηνία για τη μετάβαση από το ένα σύστημα στο άλλο. Υπάρχει. <coughs> Κύριε Κίρνερ, θέλετε να απαντήσετε. Οι άλλοι συνάδελφοι, έχετε συμπροματική διευκρινιστική ερώτηση μετά από όσα ακούσατε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όχι, ο κύριος Γκέντνερ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ για την ερώτηση που δίνει την ευκαιρία να διευκρινίσω κάτι. Καταρχάς, βεβαίως, το πρέπει θα τεθεί σε ε, ισχύ αργότερα από ό,τι έχει προβλεφθεί. Γι' αυτό δεν χρειάζεται πλήρη αξιολόγηση αυτή τη στιγμή το usage στο ΣΕΚΑ ε, λίγη του χρόνου. Έχουμε δύο παράλληλα έγγραφα που δεν είναι το ιδεώδες. Θα μπορούσαμε, για να είμαι ειλικρινής, να το κάνουμε, αλλά δεν θα ήταν το ιδεώδες αποτέλεσμα. Αν καταφέρουμε να προσαρμόσουμε το επίπεδο 2 για να μπορεί να λειτουργεί και για τα, τους οργανισμούς ως ΕΚΑ και κάνουμε και, και πολύ στοχευμένες αλλαγές για να μπορούν να χρησιμοποιήσουν και οι ΟΣΕΚΑ το προσπέκτους του Πρίπς ε, έχει καλός. Θα συζητήσουμε με όλους τους ενεχομένους και τους ενδιαφορομένους και χαιρόμαστε και για την πρωτοβουλία του εισηγητού να βρεθεί ένας τρόπος να προχωρήσουμε. Ευχαριστούμε κύριε κύριε Ο Βόλφ Κλίντς ε, για να κλείσει. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ τους συναδέλφους, ειλικρινά για τα όσα είπαν και πολύτιμες ήταν οι προτάσεις τους. Σίγουρα θα τις ε, μεταφράσουν και σε τροπολογίες. Βεβαίω, και προφανώς υπάρχουν κάποια σημεία που μπορεί να διαφωνούμε στην θεώρησή μας. Αλλά από όσα άκουσα μάλλον θα καταλήξουμε σε συνένεση για την προστασία των επενδυτών. Σβέν. Και βέβαια με ενδιαφέρει πολύ. Το είπα και προηγουμένως στις εποπτικές αρχές. Και φυσικά θα το αναφέρω. Σε καμία περίπτωση δεν θα αφήσουμε σε χειρότερη μοίρα τους επενδυτέ από ό,τι είναι σήμερα. Ίσα το αντίθετο θέλουμε. Βελτίωση. Προς τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ευχαριστώ πολύ ε, για τα όσα είπατε. Για, τους, για τα πρέψη έχουμε την ίδια στόχευση πιστεύω. Και αν καταφέρουμε να τα λύσουμε τόσο το καλύτερο. Ε, ας αξιοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία. Ε, πάντως το χρονοδιάγραμμα είναι αρκετά φιλόδοξο. Ε, τροπολογίες μέχρι τις 22 Οκτωβρίου, τις περιμένω με χαρά και έχουμε τη φιλοδοξία 19 και 20 Νοεμβρίου να ψηφίσουμε εδώ στην Επιτροπή ΕΚΟΝ έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι πολύ πριν τα τέλη του έτους και να μπορέσει να διαμορφώσει άποψη στο Κοινοβούλιο για να πάμε στις συνομιλίες και τις διαπραγματεύσεις του τριμερούς διαλόγου. Για να το κλείσουμε το θέμα μέχρι τέλη Φεβρουαρίου και πιστεύω ότι μπορεί να είναι φιλόδοξο το χρονοδιάγραμμα πλην ε, ρεαλιστικό όμως. Και χαίρομαι για τις συνομιλίες που θα έχω τι επόμενες μέρες με τους σκιώδει συγητές. Ευχαριστώ πολύ Βόλφ, ο Πρόεδρος. Θυμίζω, προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών 22 Οκτωβρίου. Στι 19 Νοεμβρίου θα ψηφιστούν εδώ, θα συζητηθούν και θα ψηφιστούν έτσι ώστε να πάει στη δεύτερη ολομέλεια του Νοεμβρίου το θέμα και να το ψηφίσουμε εκεί. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενο θέμα στη μέρη σε διάταξη. Το σημείο 9. Θέσπιση του προγράμματος φυσκάλης για τη συνεργασία στον τομέα της φορολογίας. Η συγκητής εδώ είναι ο κύριος Σβέν Γκίγκολτ, που έχει και το λόγο για 5 λεπτά, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, χαίρομαι που δεν με κατατάξατε στην ε, Γκουε με αυτή την ε, φορά. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε μία έκθεση που νομίζω τελικά μπορεί να τύχει ευρεία ε, συνένεση. Η Κομισιόν πρότεινε το πρόγραμμα Φίσκαλης να παραταθεί και έτσι να υπάρξει μια επιπλέον χρηματοδότηση κατά 82 εκατομμύρια ευρώ για να δείξουμε ακριβώς την έμφαση που αποδίδουμε στην ενίσχυση της συνεργασίας των φορολογικών αρχών των κρατών μελών. Γνωρίζετε ότι 70% των χρημάτων πάει σε τεχνολογία πληροφορικής για να διευκολυνθεί η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών. Ουσιαστικά θα υπάρξει μια συνεργασία για το θέμα της φοροδιαφυγής, φοροαποφυγής και καταπολέμησης του του χρήματος. Δεν νομίζω να διαφωνούμε πολύ εδώ πέρα. Η Κομισιόν έχει υποβάλει μια σωστή πρόταση και νομίζω ουσιαστικά συμφωνούν και τα κράτη-μέλη. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν κάποια σημεία στα οποία θεωρώ ότι θα πρέπει να επιμείνουμε σε κάποιες βελτιώσεις και αλλαγές και να μπούμε σε συζητήσεις με τα κράτη-μέλη. Δεν θα κάνουμε τώρα την παρουσίαση των αλλαγών που προτείνει το Κοινοβούλιο Απλά θα πρέπει να έχουμε δικαίωμα πλήρης, ε, πλήρους συναπόφασης και στην δευτερογενή νομοθεσία και να μην έχουμε κάποιες πράξεις κατά εξουσιοδότηση αγαπητοί συνάδελφοι. Επιπλέον, είναι σημαντικό στις ετήσιες ε, εκθέσεις ε, για το φυσκάλις να μάθουμε κάποια πράγματα. Δηλαδή το τι υπάρχει εκεί ως ευρήματα. Ε, γνωρίζετε ότι υπάρχουν και κάποιες κοινέ ε, επισκέψεις, η λεγόμενη κοινή έλεγχη. Και βεβαίως ε, τα ευρήματα δεν τα πληροφορείται η κοινή γνώμη και το Κοινοβούλιο, ενώ θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο για την νομοθετική διαδικασία. Γι' αυτό πρότεινα στην έκθεσή μου να διαμορφωθεί εδώ πέρα ένα πλαίσιο περισσότερης διαφάνειας ε, όσον αφορά τις αιτήσεις εκθέσεις. Επιπλέον, ε, στο θέμα των ε, ανταλλαγών πληροφοριών υπάρχουν εντωμεταξύ κάποιες διεθνείς προδιαγραφές Οπότε θα έπρεπε ακριβώς ε, οι χώρες οι οποίες ε, δεν έχουν προχωρήσει εδώ να βοηθηθούν ε, για να μπορούν να λαμβάνουν μέρος στην διεθνή αυτή δραστηριότητα. Επίσης θα ήθελα να τονίσω ότι κατά την άποψή μου θα ήταν λογικό το Κοινοβούλιο να καθορίσει κάποιες προτεραιότητες για συγκεκριμένους τομείς. Αυτό μπορεί να γίνει σε ένα παράρτημα, αλλά είναι επίσης αποφασιστικό να φροντίσουμε να υπάρχουν αρκετά κονδύλια για τις δραστηριότητες που όντως φέρνουν λεφτά. Οι κοινοί έλεγχοι, παραδείγματος χάρη, έχουν νόημα, έχουν ε, άμεση επίδραση στα έσοδα. Άρα θα έπρεπε να είναι ανάλογα πρώτη προτεραιότητα. Θεωρώ ότι είμαστε σε ένα τομέα μάλλον τεχνικών συζητήσεων και αναμένω το τι έχουν να πούν οι συνάδελφοι. Μια να δω. Α, ε, τι έχουν να πούν για το θέμα και ελπίζω να καταλήξουμε σύντομα σε έναν συμβιβασμό γιατί νομίζω ότι είμαστε οι πρώτοι που ασχολούμαστε με αυτό το θέμα το δεν είναι τόσο επίμαχο καλό θα ήταν λοιπόν η ΕΚΟΝ να καταφέρει να ολοκληρώσει πρώτη αυτά τα θέματα ευχαριστώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ συνάδελφος Φέρμπερ δεν είναι εδώ αυτήν την στιγμή. Α, είναι ο κύριος Σοβάμπ, μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ που μου δίνετε τον λόγο. Ο κύριος Στόλογιαν ε, κολλιέται σήμερα και μου ζήτησε να σχολιάσω την έκθεση του κυρίου Γκίγκολτ ως εξής κύριος Χαίρετε που μπορώ να τον αντικαταστήσω και μου είπε και στο Λογιάννη το πρόγραμμα Φισκάλη απο... ήταν αποτελεσματικό στο τρέχον ε, δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020 και σε αυτό συμφωνεί με τον ΣΒΕΝ. Ε, είναι το μόνο ευρωπαϊκό πρόγραμμα που εστιάζεται επειδή βασικών στόχων να αναπτύξει και να διατηρήσει τι πληροφορίε τεχνική, πληροφορική για την αλλαγή πληροφοριών και στη μεταξύ των φορολογικών αρχών των κρατών μελών. Να υποστηριχθεί η δημιουργία δυνατότητα διοικητική και ανθρωπίνων δυνατοτήτων και δεξιοτήτων και να υπάρχει και ανταλλαγή απόψεων άμεση και ερωτήσει των πρακτικών μεταξύ επαγγελματιών από τι αρχέ φυσκάλη, άλλα θεσμικά όργανα και εμπειρογνώμου για τα φορολογικά, ώστε να καταπολεμηθεί η φορολογική απάτη, κοινό στόχο όλων μα, η φοροδιαφυγή και η φοροαποφυγή. Τι ο τρόπο θεωρούμε σαν ΕΛΚ ότι το φυσκάλη θα πρέπει να συνεχίσει στο νέο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027 και καλωσορίζουμε την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη σχετική προσέγγιση. Μετά πιστεύουμε ότι ο ο κ. τον ευχαριστούμε για το σχέδιο εκθέσεώς τους, ε, μπορούμε να το υποστηρίξουμε στι τροπολογίε που υποβάλλει και από την έποψη που βλέπουμε εμεί τα πράγματα, οι περισσότερε τροπολογίε μπορούν να στηριχθούν από το ΕΛΚ. Όμω υπάρχει δυνατότητα οι συνάδελφοι να εκφράσουν προτάσει, να προτείνουν τροπολογίε όσον αφορά το σχέδιο κανονισμού και όσον αφορά το σχέδιο κειμένου, σχέδιο εκθέσεω του συγκητού. Τρίτον, είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε και να επεξεργαστούμε τι αναγκαίε συμβιβαστικέ συμπεριλαμβανομένων άλλων πολιτικών ομάδων σχετικά με αρκετέ τροπολογίε, όπω 17 που αναφέρεται στο άρθρο 7 παραγραφο 2 2α. Εδώ θα θέλαμε να δούμε καλύτερη διατύπωση για να εγκαθίσει σαφέ ότι η δημιουργία ποιοτικού μητρώου για τους δικαιούχου ιδιοκτήτες εταιριών αποτελεί ευθύνη του κράτου μέλους. Η τροπολογία 19 το ίδιο που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 ε, δεν βλέπουμε το λόγο για τον οποίο δεν μπορούμε να δεχτούμε εξωτερικούς εμπειρογνώμονες όπως εκπροσώπους διεθνών και άλλων σχετικών οργανισμών δεν συμφωνούν με την τροπολογία να αποκλειστούν από τη συμμετοχή τους σε δράσεις που διοργανώνονται στα πλαίσια του προγράμματος. Τέλος, τροπολογία 35 που αναφέρει στο παραδειγμα 2, σημείο 2α, δίκτυοι που προτείνει ο συγγετής περί εισοδημάτων που συλλέγονται στην προσπάθεια καταπολεμήσεων φοροδιαφυγής, φοροαποφυγής για να δουν πόσο αποτελεσματικό είναι το πρόγραμμα. Αυτό θα δημιουργούσε κίνητρα να αναφέρονται μεγάλοι αριθμοί που δεν έχουν ε, σχέση με την πραγματικότητα και δεν πρέπει να είναι αυτό το στόχο των τροπολογιών και ο σκιώδη ηγητή θα ήθελε να δει μια τροπολογία που θα βελτιώνεται, θα βελτιώνει την κατάσταση. Αυτά είναι τα σχόλια του συναδέλφου Στόλο που δεν μπορεί να είναι εδώ. Ευχαριστώ την προσοχή σα. Ευχαριστώ, Αντρέα, από του Σοσιαλιστέ και Δημοκράτε. Κανονικά, ο Ουικ Μπαγιέ, τον οποίο εκπροσωπεί η κυρία Περβάν Βερέ. Βερές. Ευχαριστώ. Εγώ τώρα βρίσκομαι σε περίεργη κατάσταση, γιατί ο κύριος Ζουικ Μπαγιέ μου έδωσε κάποια σημεία να διαβάσω στα αγγλικά για να το αντικαταστήσω. Λοιπόν, ζητάει συγγνώμη διότι δεν μπόρεσε να είναι παρόν, όμως καλωσορίζει το έργο του Σβέν Γκίγκολτ που έκανε πάνω σε αυτή την έκθεση. Ε, διεξοδική προσπάθεια που καταβάλει, θα υποβάλουμε κάποιες τροπολογίες. Κυρίζει τη φορολόγηση φυσικών προσώπων και εταιριών. Το φυσκάλις πρέπει να βάλει προτεραιότητες προτεραιότητα έχει η εφαρμογή των διαθετήσεων επιμερισμού διάδοση των πληροφοριών σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ενώσεω από τον DAC 3, 4, 5, 6 και για την οδηγία για διοικητική συνεργασία μεταξύ εφοριών πρέπει να εφαρμόζουν οι αρχές ασφαλή λογισμικό και εφοριακή αρχή πρέπει να είναι εκπαιδευμένοι να χρησιμοποιεί το ειδικό λογισμικό, κάτι που χρειάζεται πόρους ειδικού για να επιδιωχθεί ο στόχος συλλογής πληροφοριών για δυσκολίες που δημιουργήθηκαν από την εφαρμογή της συνεργασίας των εφοριών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ενώσης, συλλογή πληροφοριών χρειάζεται θα μπορούσε να υπάρχει μια μόνιμη, μικρή μόνιμη αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες που θα συγκεντρώνει σε κεντρικό σημείο τις πληροφορίες από όλα τα κράτη-μέλη. Επίσης, θα προσπαθήσουμε να διευκρινίσουμε το κομμάτι, το ρόλο που παίζει το πρόγραμμα Φισκάλης, η επιτροπή του προγράμματο Φισκάλης και προσβλέπουμε στη συζήτηση από αυτού που γίνεται περαιτέρω σημαντική στα πλαίσια που χρειάζεται συνεργασία για την καταπολέμηση ξεπλήματο χρήματος και θα είναι σημαντικό κομμάτι της επικείμενης μεταρρύθμισης όπως ο φόρος για τις ψηφιακές υπηρεσίες. Ευχαριστώ πολύ Περβάς. Ρόπερτ Ζήλε κανονικά από το ECR, τον οποίο εκπροσωπεί ο Άσλι Φόξ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο δικός μας σκιώδης ηγητής, κύριος Ζήλε, ζητεί συγγνώμη για την απουσία του σήμερα. Ε, είναι ακόμα στη Ρήγα, ε, και, ε, γιατί έγιναν εκλογές εκεί το Σάββατο. Ε, καλωσορίζουμε την έκθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ευχαριστούμε τον κύριο Γκίγκολ για τις προσπάθειες του να βελτιώσει το κείμενο. Το ECR συμφωνεί ότι είναι σημαντικός ε, ο θεμητός ανταγωνισμός στην εσωτερική αγορά. Επίσης, η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής και της φορολογικής απάτης είναι υψίστης σημασίας. Ιδιαίτερα γιατί είναι σημαντικά έσοδα που χάνονται από τους κρατικούς προπολογισμού. Υποστηρίζουμε τον εισηγητή στι προσπάθειες αυτές και Εκτιμούμε το γεγονό ότι ο κύριο Γκίγκολτ λέει ξεκάθαρα ότι το Μένο Βασίλειο θα μπορέσει να ενταχθεί στο πρόγραμμα αυτό μετά την αποχώρησή του από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε περίπτωση που το επιλέξει. Από την άλλη δεν συμφωνούμε με τον εισηγητή ότι λιγότερο ανεπτυγμένε χώρε θα πρέπει να έχουν μεγαλύτερη προτεραιότητα ειδική μεταχείριση. Η πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ένταξη και τι συνδεδεμένε χώρε φαίνεται πιο ισόρροπη. Φρονεί το ECR ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει κατάλογο προτεραιοτήτων, θεμάτων προτεραιοτήτων, γιατί ακόμα και αν δεν είναι εξαντλητικό. θα περιόριζε το πεδίο εφαρμογής και θα ήταν ιδιαίτερα ε, ε, έτσι, καθοδηγητικός. Είναι καλή αρχή και αφετηρία η έκθεση Γκίγκολ και προσβλέπουμε στην επικοδομητική συνεργασία μαζί του. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ, Άσλι. Από τους φιλελευθέρους δεν υπάρχει κανείς. Οπότε, Γκουε, ε, ο Μάρτιν Σίρδεβαν, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Είναι γνωστό ότι εμείς οι αριστεροί έχουμε γενικά κριτική στο σχέδιο για το PDP αυτό δεν έχει να κάνει κυρίως με το φυσκάλι Σβέν, αλλά τις περικοπές ε, στα διαρθρωτικά ταμεία και τα περιφερειακά και η μεταφορά πιστώσεων στη στρατιωτική συνεργασία. Σε αντίθεση με όλα αυτά, εμεί επενούμε την έκθεση του Σφεν για το φυσκάλι, γιατί θεωρούμε πάρα πολύ σημαντική την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής. Δηλαδή, εμεί δεν υποστηρίζουμε την πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά την πρόταση του εισηγητού, γιατί τη θεωρούμε καλύτερη δεν ξέρω πώς χειρίζεσαι τον έπαινο Σφεν, επειδή δεν έχουμε μπει ακόμα στην προεκλογική εκστρατεία. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει και, μέσα στην εκστρατεία τα πει Μάρτιν, δεν πειράζει να με πενείτε όποτε θέλετε. Ε, μάλιστα, αμοιβαία τα αισθήματα. Οι ε, δικές μας τροπολογίες έχουν να κάνουν με τη μεγαλύτερη διαφάνεια ε, συμφωνούμε με αυτά που προτείνει και για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Γενικά είμαστε πάρα πολύ θετικοί και θα παρακολουθήσουμε την έκθεση αυτή. Η ΕΝΕΦ κανονικά η Μπάρμπαρα Κάπελ, η οποία επίσης απουσιάζει. Η FTD είναι κανείς εδώ. Όχι. Τότε θα δώσω αμέσως το λόγο στον εισηγητή μας, τον κύριο Σβέν Γκίγκολτ. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ για όλα αυτά τα σχόλια. Θα ήθελα να κάνω μόνο κάποιες ε, σύντομες παρατηρήσεις. Πρώτα απ' όλα, δεν πρότεινα, και ίσως υπάρχει εδώ μια παρεξήγηση, να μην προσκαλούμε πλέον εξωτερικούς, δηλαδή η τροπολογία 19 διακρίνει μεταξύ συναντήσεων των εκπροσώπων του κοινού και τη δυνατότητα μετά να προσκαλέσουμε όλους τους άλλους. Γιατί έτσι νομίζω θα λειτουργούν ε, κανονικά οι ευρωπαϊκές αρχές. Έχουμε δηλαδή ευρωπαϊκούς φορείς ε, που αποτελούνται από εκπροσώπους του Δήμου και μετά μπορούμε να προσκαλέσουμε και κάποιους εξωτερικούς εμπειρογνώμονες ανάλογα με τις ανάγκες. Ίσως πρέπει να το διευκρινίσω, αλλά ε, διαβεβαιώ τον κύριο Στόλογιαν ότι αυτό δεν ήταν ποτέ η πρόθεσή μου. Να αποκλείσω δηλαδή όλους τους εξωτερικούς συμμετέχοντες. Μετά, όσον αφορά τα έσοδα και εκεί η έκθεση όπως ε, την έχω συντάξει μπορεί να βελτιωθεί. Δεν ήταν ποτέ η πρόθεσή μου γενικός ε, όλη η ανάκτηση χρημάτων στην καταπολέμηση φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής να χρησιμοποιείται ως δίκτυς, αλλά συγκεκριμένα τα έσοδα που δημιουργούνται μέσω των δραστηριοτήτων του προγράμματος. Μόνο η κοινή έλεγχη δηλαδή. Και μπορεί να το ξεκαθαρίσει αυτό η τροπολογία ε, για την πιθανή αυτή κατάχρηση που αναφέρει ο κύριος Στόλογιαν για να αποφευχθεί. Από αυτό αναμένω τις ε, προτάσεις του Ουγγ για την θεσμική πτυχή και είμαι οπωσδήποτε ανοιχτός ε, στην ιδέα του να έχουμε οπωσδήποτε μια ισχυρότερη θεσμική πλαισίωση και αναμένω να δω πώς θα το παρουσιάσει. Ευχαριστώ Μάρτιν για την στήριξη ε, και όπου δεν συμφωνώ αν και βεβαίως σημειώνω το ότι γενικότερα είναι κάπως πιο ανοιχτός ο κύριος Ζήλε του ECR και μας στηρίζει είναι ότι δεν μπορούμε ότι θα έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε τα όσα έχουμε για να βοηθήσουμε και τις φορολογικές διοικήσεις στις φτωχότερες χώρες. Δεν ξέρω γιατί θέλετε να διαγραφεί αυτό. Νομίζω ότι είναι προστιθέμενη αξία για αυτούς που το χρειάζονται περισσότερο. Και τέλος, για τα θέματα προτεραιότητας. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε και αυτό είναι κάτι το οποίο είχα πει στο σχέδιο έκθεσης πως ε, δεν πρέπει για έναν οριστικό κατάλογο αλλά δείχνει ότι το κοινοβούλιο αυτό μετά από πολλά χρόνια δουλειάς ε, στις ε, επιτροπές μας έχουμε καταλήξει κάπου όσον αφορά τα βασικά προβλήματα στη συνεργασία μεταξύ φορολογικών αρχών και λογικό είναι να θέσουμε και κάποιες προτεραιότητες ε, για αυτά τα 7 χρόνια για να αξιολογήσουμε και την εφαρμογή του προγράμματος. Αλλά θα ήθελα να τονίσω ότι δεν έχουν στόχο αυτά να είναι περιγραφικά και να λέμε ότι μόνο με αυτά πρέπει να ασχοληθεί το φυσκάλις. Πρέπει να είναι κάποια πολιτική κατεύθυνση και θεωρώ ότι οπωσδήποτε οι πολίτες αφού πληρώνουν για το πρόγραμμα νομίζω ότι δικαιούνται να θέσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάποιες προτεραιότητες. Οπότε ε, είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε πάρα πολλές ε, τροπολογίες και υπό αυτή την έννοια ελπίζω να έχουμε την ευρύτερη δυνατή πλειοψηφία. Για κάτι το οποίο αξίζει νομίζω. Ευχαριστώ πολύ Σβέν κανονικά. Α, προθεσμή υποβολή τροπολογιών. 17 Οκτωβρίου. Συζήτηση τροπολογιών. 19. Ψηφοφορία 27 Νοεμβρίου στην ΕΚΟΝ. Συνάδελφοι, κανονικά θα ξεκινούσαμε το σημείο 10 της μέσης διαταξίας. Συνορική σύγκληση, συγχωνεύσεις κλπ. Στις 6 και 4. Βλέποντας τον κατάλογο σκιωδών, μόνο ο Ραμόν Τρεμόζα αναμένεται. Είναι ενδεικτικό το χρονοδιάγραμμα. Προτείνω να ξεκινήσουμε τώρα λοιπόν. Αν δεν έχετε πρόβλημα βέβαια. Ο πρώην πρόεδρος, η πρώην πρόεδρος, η Περβάνς Περές, συμφώνησε να αναλάβει την προεδρία Ας ξεκινήσετε με αυτό το σημείο. Πιο λογικό αυτό, παρά να ξεκινήσω και να αναλάβετε εσείς μετά. Και ίσως να καταφτάσει και ο Ραμόν μέχρι τότε. Um, λοιπόν, προχωρούμε στην εξέταση 10 και θα δώσω το λόγο στον Όλε Λούτβικσον για να μας μιλήσει για τις διασυνοριακές μετατροπές συγχωνεύσεις και διαιρέσεις και τις ναι, αντίστοιχες τροπολογίες. Ευχαριστώ πολύ. Ξεκινώντας θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους σκιώδεις ε, εισηγητές για τις συζητήσεις που υπήρξαν άκρως επικοδομητικές και πράγματι είχαμε πολλές υποβληθήσεις τροπολογίες και θα πρέπει να τις εξετάσουμε. Υπάρχουν πολλές τροπολογίες πολύ ποιοτικέ. Είναι προφανές επίσης ότι υπάρχει κάποια απόλωση σχετικά με αυτό το θέμα συνδέεται κυρίως η πόλωση με τους ε, όρους, με τις συνθήκες ε, όσον αφορά τη διασυνοριακή δραστηριότητα, αφορά επίσης και τον ορισμό των διαφόρων τεχνητών ε, μέτρων. Θα πρέπει να υπάρχει επαρκής ορισμός του τεχνητού διαχωρισμού, θα πρέπει να, να καθορίσουμε τι είναι αυτό από πλευράς φορολογικής θα πρέπει να αποφύγουμε το ότι τα κράτη-μέλη δεν θα ερμηνεύσουν τον ορισμό αυτό με έναν τρόπο ασυνεπή, με έλλειψη συνοχής. Δεν θα πρέπει λοιπόν αυτού του είδους οι κινήσεις ε, να είναι τεχνητού χαρακτήρα και θα πρέπει να υπάρχει συσχετισμός πραγματικός με την χώρα που φιλοξενεί τις ε, εταιρείε. Θα πρέπει να υπάρχει ασφάλεια δικαίου και να αποφύγουμε κάθε κατάχρηση της ελευθερίας ε, εγκατάστασης. Υπήρξε μια σειρά απόψεων ε, που εξεφράστη από τους συναδέλφους επ' αυτού την ελευθερία της εγκατάστασης και των τεχνητών αυτών συγχωνεύσεων, ε, διαχωρισμών κλπ. Η άποψή μου να προσπαθήσουμε να συμφωνήσουμε μεταξύ μας. Θεωρώ, εν πάση περιπτώσει, ότι υπάρχει συμφωνία όσον αφορά το διασυνοριακό χαρακτήρα αυτών των κινήσεων. Είναι σημαντικό ε, να λάβουμε υπόψη ορισμούς που είναι σαφείς και θα πρέπει βέβαια να είναι και εναρμονισμένοι οι κανόνες για τις διασυνοριακές ε, αυτές κινήσεις και επιχειρήσεις. Θα πρέπει να ε, τοποθετηθούμε και επί των ελέγχων που θα διενεργούνται. Πρέπει να διενεργείται από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα έλεγχος ή από κάποια αρμόδια αρχή. Είναι σημαντικό επίσης η έκθεση που υποβάλλουν οι εταιρείε να συντάσσεται ε, με τέτοιο τρόπο που να υπάρχει δυνατότητα σύγκρισης μεταξύ εκθέσεων των κρατών μελών, να υπάρχει συγκρισιμότητα ε, και θα πρέπει να καταλήξουμε και στην ε, κατάλληλη πρόταση νομοθετικού περιεχομένου. Θα προσπαθήσω να επικεντρωθώ επί των σημείων που άπτονται της αρμοδιότητας της Επιτροπής μας. Είναι αυτό που είπα και την προηγούμενη φορά κατά τη διάρκεια της παρουσιάσεως του θέματο. Το άρθρο 86 είναι ένα άρθρο ιδιαίτερα σημαντικό και ξέρω ότι υπάρχουν πολλές τροπολογίες που αφορούν το άρθρο 86. Αυτό το άρθρο αφορά θέματα σημαντικότατα, αλλά πιστεύω ότι είναι σημαντικότατο να μην λησμονούμε ποια είναι η δική μας αρμοδιότητα θα πρέπει να παραμείνουμε στις αρμοδιότητες της Επιτροπής της Οικονομικής και γι' αυτό κάποιες τροπολογίες κατά την άποψή μου δεν μπορεί να είναι αποδεκτές. Είναι σημαντικότατο λοιπόν να επιμείνουμε σε αυτό το κείμενο επί του πραγματικά διασυνοριακού χαρακτήρα αυτών των κινήσεων. Είναι σημαντικό να συζητήσουμε μεταξύ μας το θέμα και να δούμε πού θα καταλήξουμε από κοινού ε, και ποια θα είναι η θέση της ε, που θα ακολουθήσουμε συμπεριλαμβανομένων και των διασυνοριακών στοιχείων. Αυτά και σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και περιμένω να ακούσω την άποψη των σκιωδών εισηγητών των άλλων ομάδων. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ από το ΕΛΚ. Ο Ανδρέας Σφάμπ. Ευχαριστώ. Έτσι νομίζω το λένε στα Σουηδικά. Κύρια Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Λούτβιχστον, ε, με τον οποίο είχα την ευκαιρία να συναντηθώ πολλές φορές. Την προηγούμενη εβδομάδα συναντηθήκαμε οι σκιώδεις συζητές για την έκθεση. Για εμένα και για την ομάδα του ΕΛΚ ε, μεγάλη σημασία έχουν τα εξή ε, σημεία όπως φαίνεται άλλωστε και από τις τροπολογίες. Πρώτα απ' όλα οι προϋποθέσεις για τις διασυνοριακές μετατροπές και συγχωνεύσεις. Θα ήθελα να ξεκαθαρίσω αφενός πως ε, και εγώ θα ήθελα να πω ότι είναι σημαντική η ψευδής ε, τέτοια πρακτική για στόχους ε, φόρου αποφυγής. Εξάλλου, ήδη ο Ευρωπαίος νομοθέτης έχει νομοθετήσει μία οδηγία. Βεβαίως, το φορολογικό δίκαιο δεν επαρκεί για ε, τα ζητήματα του εταιρικού δικαίου μας λέτε, κάτι το οποίο δεν μου έχει εξηγηθεί επαρκώς και είμαι κάπως επιφυλακτικός. Δεύτερον, όμως, ε, το βασικό πρόβλημα βρίσκεται ακριβώς στο άρθρο 86 γάμα το οποίο λέει ότι οι φορολογικές πτυχές θα πρέπει να συνδέονται με την δυνατότητα μη έγκρισης. Γιατί εδώ πέρα βλέπουμε δύο διαφορετικά ζητήματα γιατί ε, θα παραβιαστεί νομίζω με τρόπο που δεν επιτρέπεται η, η ελευθερία της εγκατάστασης ε, των εταιριών που προβλέπεται στην συνθήκη και στην απόφαση Πολμπούτ νομίζω το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει κρίνει ότι είτε μας αρέσει είτε όχι μπορούν να επιλέξουν ελεύθερα έδρα ή εταιρείε για οποιονδήποτε λόγο. Τρίτον, υπάρχει εδώ πέρα ένας όρος ο οποίος περιέχεται στην πρόταση της ε, Κομισιόν, ο οποίο δημιουργεί κάποια νομική ανασφάλεια. Υπάρχει μια προσπάθεια, αλλά ο ορισμός ε, αναφέρεται πάλι σε άλλους ασαφείς ε, όρους, οι οποίοι νομίζω αντιβαίνουν ξεκάθαρα στην απόφαση του δικαστηρίου την οποία μόλις ανέφερα και δεν μπορεί να στηρίξει ομάδα μας. Το δεύτερο κομμάτι εδώ πέρα λέει ότι οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν πληγεί από την κρίση δεν θα πρέπει να αποκλειστούν από την διαδικασία αυτή αναδιάρθρωσης ή συγχώνευσης για να μπορέσουν να βγουν από την κρίση. Και χαίρομαι για το ότι το δέχτηκε στις συμβατικές προτάσεις ο εισηγητής επιπλέον θα πρέπει να πω πως έχουμε μεγάλη ανησυχία για τις ε, τροπολογίες που επεκτείνουν κατά πολύ το πεδίο εφαρμογή και περιορίζουν την ελευθερία εγκατάστασης. Για εμένα κάποιες από αυτές τις εξαιρέσεις δεν είναι αντιληπτές, όπως του χάρη το να αποκλείεται κατηγορηματικά η μετατροπή εάν είχε λάβει επιδοτήσει στο παρελθόν η επιχείρηση. Εδώ πέρα μιλάμε για θέσεις εργασίας, για επιχειρήσεις και οι θέσεις αυτές εργασίας θα πρέπει ακριβώς όταν επιλέγεται μια τέτοια νομική κατασκευή να διατηρηθούν και να μην ε, διακινδυνεύουν από τέτοια νομικά εμπόδια. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε την πραγματική εφαρμοσιμότητα όλων αυτών των διατάξεων για να μπορούν να εκπληρώνουν και τον επιθυμητό στόχο. Θα πρέπει δηλαδή οι διατάξεις αυτές να μην έχουν μόνο νομική βεβαιότητα, αλλά να είναι και εφαρμόσιμες στην πράξη από τις επιχειρήσεις. Αυτό ακριβώς ε, είναι κάτι το οποίο πρέπει να δούμε σε διάφορες ε, τροπολογίες, ε, γιατί δεν ισχύει για πολλές από αυτές και ακριβώς δεν αξίζει το επιπλέον άχθος το οποίο υπερβαίνει και την πρόταση της ε, Κομισιόν το οποίο θα επομιστούν οι επιχειρήσεις και εκεί πέρα ακριβώς θα αποτύχει αυτή η πρόταση και θα χρησιμοποιήσουν λιγότερο την ελευθερία εγκατάστασης οι επιχειρήσεις δηλαδή θα περιοριστεί η εσωτερική αγορά. Λοιπόν, θα πρέπει να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους ε, τα κράτη-μέλη ειδικά όσον αφορά την εφαρμογή της φορολογικής νομοθεσίας για να μην υπάρχει δυνατότητα φόρο αποφυγής και θα πρέπει να ε, τα δει αυτά και ο εθνικός νομοθέτης να διασφαλίσει δηλαδή ότι υπάρχουν τα απαραίτητα εργαλεία στην φορολογική πρακτική και να μην υπάρχει ένας ανταγωνισμός μεταξύ των κρατών μελών και να δίνεται έτσι η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να χρησιμοποιούν την εσωτερική αγορά χωρίς να κάνουν κάποια φορολογικά κόλπα. Ευχαριστώ. Από τους φιλελευθέρους. Ο κύριος Τρεμόσα. Κατέφτασε. Έχει αμέσως το λόγο. Αλλά προηγουμένως το ECR γιατί είναι μεγαλύτερη ομάδα. Είναι εδώ κάποιος από το ECR. Δεν τον εκπροσωπεί κανένας άλλος. Ο κύριος Τρεμόσα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω τον συγγητή Όλε Λούτβιξον για το έργο του. Λέει στα αγγλικά ο κύριος Τρεμόσα. Ορισμένοι συμβιβασμοί συζητήθηκαν την περασμένη εβδομάδα, όπως η συμβαστική πρόταση F που συνδέεται με την H. Η ομάδα μου διαφωνεί για την σύγκληση και ποιος θα, το εξετάζει, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους ή ανεξάρτητος εμπειρογνώμων. Εμείς διαφωνούμε σε αυτό το σημείο. Σε ό,τι αφορά τον ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα, συμφωνούμε με τη σημερινή συμβαστική πρόταση H. Θα πρέπει να είναι ανεξάρτητος ο εμπειρογνώμονα από την εταιρεία σύγκλησης και να μην υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ ε, των ενεχομένων. Σε ό,τι αφορά τον συμβασμό I, η εταιρεία που κάνει τη μετατροπή. Ε, μετατροπή, conversion, όχι σύγκληση. Το ε, αντίστοιχο πιστοποιητικό θα πρέπει να έρθει μετά από ε, ειδική αίτηση. Σε ό,τι αφορά τη συμβαστική πρόταση γάμα, οι προϋποθέσεις για τις διασυνοριακές συνεργασίες δεν είναι ξεκάθαρες για την ομάδα μας. Εμείς θα θέλαμε να ε, γίνει μια διάκριση ανάμεσα στην φοροαποφυγή και στη φοροδιαφυγή. Τα ξανά είπαμε αυτά την περασμένη εβδομάδα. Και θέλουμε να διαγραφεί το σημείο ΙΑΙΑ που είχε να κάνει με τη συνένεση που θα πρέπει να δώσουν οι εκπρόσωποι των εργαζομένων. Στην ε, συμβιβαστική day ζητούμε το JJ και το JK να διαγραφούν που κάνουν τις μετατροπές ιδιαίτερα άκαμπτες Επίσης, ε, το σημείο BA, μεταξύ άλλων, έχει να κάνει με τις βασικές πληροφορίες για το τζίρο των εταιριών και ε, τον ισολογισμό τους τελευταία πενταετία. Συμβαστική ή e για την ενημέρωση εργοδοτών και εργαζομένων. Συμφωνούμε με τα όσα λέει ο εισηγητής. Δεν χρειάζεται τα pension funds να ενημερώνονται. Και ε, J, K, L, M και N μας βρίσκουν σύμφωνοι. Αύριο θα συζητήσουμε τις νέες ε, συμβαστικές και θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πολύ. Ραντεβού αύριο. Δεν Γκίγκολτ από τους Πρασίνους. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. I just like to, follow Πάνω στα βασικά θέματα που αναφέρθηκαν να πω και εγώ κάποια πράγματα σημαντικό αυτή η έκθεση να μπει στο σωστό πλαίσιο. Θυμάμαι και πολύ καλά μάλιστα που στα πλαίσια των συζητήσεων της διαβόητης εκθέσεως Μπόλκενστάιν οδηγίας Βολκενστάιν και μετά διάφορες αποφάσεις του ΔΕΚ διαμορφώθηκε μια μεγάλη αμφιβολία κυρίως στην κοινωνία των πολιτών, των συνδικάτων, και στον επιχειρηματικό κόσμο δημιουργήθηκαν αμφιβολίε κατά πόσο είναι καλή πρακτική εταιρείε της κοινή αγοράς να προσπαθούν να επιλέξουν το ρυθμιστικό περιβάλλον και να υπάρχει ανταγωνισμός ρυθμιστικών περιβαλλόντων. Δημιουργήθηκε αναταραχή στην κοινωνία των πολιτών και τελικά ιτήθηκε το βασικό κομμάτι της οδηγίας Μπολκενστάιν σε αυτό το τομέα έχουμε κάτι πολύ παρεμφερές. Και γι' αυτό αυτή η οδηγία μπορεί να είναι νέο πεδίο μάχης για παρομοίου τύπου δημόσια συζήτηση. Οι εταιρείε θα έπρεπε να έχουν τη θέση, τη δυνατότητα μέσω ε, εξαγορών, συγχωνεύσεων να αλλάξουν το ρυθμιστικό περιβάλλον και να το κάνουν αυτό σκόπιμα ούτως ώστε να πετύχουν σημαντικά ωφέλη έναντι ανταγωνιστών. Αν δείτε τις διαφορές που υπάρχουν όσο αφορά την νομοθεσία και τους κανόνες, κυρίως για τα φορολογικά και τη συμμετοχή των εργαζομένων, αν όπως υπάρχουν ενδείξεις ότι αυξανωμένως συμβαίνει αυτό, αν οι εταιρείε χρησιμοποιώντας συγχώνευση και ε, αναδιαρθρώσεις αποφεύγουν ισχυρότερα, ισχυρότερο περιβάλλον ε, νομοθετικό για να μετακινηθούν προς ένα ασθενέστερο, μπορεί να, λες, να αρέσει σε προασπιστή ε, της ελεύθερης αγοράς να θεωρεί ότι υπάρχει ισχυρός νομοθετικός ανταγωνισμός. Αλλά αυτό ε, δημιουργεί προβλήματα όσον αφορά την κοινή αγορά για μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού. Πρέπει να βρούμε λύσεις για τα πραγματικά προβλήματα, χωρίς να αμφισβητούμε τη δέσμευση για συμμόρφωση με την κοινή αγορά, αλλά για να προστατεύσουμε ε, μια γενικότερη ε, υποχρέωση και δέσμευση έναντι της κοινή αγοράς. Όπως τα βλέπω εγώ τα πράγματα. Πρέπει να είναι ισχυρός ε, ο ορισμός για τεχνητές διευθετήσεις. Και αυτό σχετίζεται με οικονομική ουσία. Έτσι αποφεύγουμε αυτές οι αναδιατάξεις να γίνονται βασικά για να επιτευχθούν οι αλλαγές στον κανονισμό. Πιστεύουμε μετά, και αυτό είναι και νομικό θέμα, ο Ανδρέας Σφάμπ το έθεσε όσον αφορά το άρθρο 86C και παρεμφερεί άρθρα αν υπάρχει περιθώριο για κάποιους ελέγχους χωρίς να αντιβαίνουμε τις αποφάσεις του ΔΕΚ ό,τι προτείνουμε εμείς πρέπει να είναι νόμιμο. Διαφορετικά είναι άχρηστο. Δεν πρέπει να δώσουμε συμβολική μάχη εδώ πάνω σε μια γνωμοδότηση που δεν έχει νόημα. Αυτά τα θέματα είναι πάρα πολύ σοβαρά για συμβολικές μάχες. Είναι, πολύ, είναι πολύ εύκολο να γίνει αυτό. Να το πλαισιώσουμε έναν τρόπο που θα αποτελέσει πεδίο συμβολικής μάχης. Πρέπει να δούμε τι περιθώριο νομικό έχει αφήσει για να κινηθούμε εμείς το ΔΕΚ και να χρησιμοποιήσουμε ε, το χώρο αυτό για να πετύχουμε το μέγιστο δυνατόν. Έτσι θα είναι πιθανότερο η φοροαποφυγή και η φοροδιαφυγή να χρησιμοποιούνται μέσω συγχωνεύσεων και γενικών αναδιατάξεων των επιχειρήσεων. Να μην διευκολύνεται αυτό. Και να αποφεύγουν και τους κανόνες ε, ε, καθορι... ε, αυτοκαθορισμού των επιχειρήσεων. Αυτό που δεν μπορούμε να κάνουμε είναι να αλλάξουμε τη συνθήκη. Όταν χρειάζεται να αλλάξουμε τη συνθήκη για να πετύχουμε τους στόχους, ε, τότε βγαίνουμε εκτός πεδίου. Μπορούμε να έχουμε αποκλίνουσες απόψεις, αλλά αυτός δεν είναι ο στόχος μας. Δεν έχει νόημα να χρησιμοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία ε, για να κάνουμε αυτό το πράγμα. Εκεί που δεν συμφωνώ με τον Αντρέα Σφάμπ είναι εδώ. Να πούμε ότι όσον αφορά τους φόρους, ψηφίσαμε το ΑΤΑ 1, ΑΤΑ 2 και τα πάντα είναι καλά. Ξέρουμε ότι αυτά δεν λύνουν τα προβλήματα. Διότι δεν έχουμε εναρμονισμένα, εναρμονισμένα ποσοστά φορολόγηση. και έχουμε επιθετικά καθεστώτα, συντελεστές φορολόγηση. επιθετικά καθεστώτα σε διάφορα κράτη-μέλη, ε, τα μέτρα. Και να μιλήσουμε τώρα για τον κύριο Σόιμπλε. Προσπάθησε επί μακρόν ο κύριο Σόιμπλε να πετύχει αυστηρότερους κανόνες όσον αφορά τα θέματα ε, ε της ε, Και χώρες από τη Γαλλία, τη Γερμανία είχαν κίνητρο να συγχωνευτούν και να δημιουργήσουν ε, να, να ενταχθούν σε καθεστώτα με πολύ αυστηρούς κανόνες περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Λοιπόν, το άτα 1 και το άτα 2 δεν αρκούν. Άρα, όπως είπε και ο συγητής και άλλοι, θα έπρεπε αυτά να τα καλύψουμε, αυτές τις τυχές. Αλλά όπως λέγατε, πρέπει να σεβαστούμε το νομικό σεφικτόν. Τέλος, στο πνεύμα το συμβιβαστικό μπορούμε να αποδεχτούμε οι μικροεπιχειρήσεις και οι μικρές επιχειρήσεις και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις να εξαιρεθούν αυτό το πεδίο εφαρμογή. Θα θέλαμε να ήμασταν φιλόδεξοι για την επίλυση των πραγματικών προβλημάτων που ενδεχομένως αφορούν ε, μεγάλο αριθμό πολιτών, την τοπική αυτοδιοίκηση, τα κράτη-μέλη που χάνουν είτε δικαιώματα συμμετοχής στις εταιρείε είτε φορολογικό εισόδημα. Συγγνώμη που μακρηγόρησα κάπως, αλλά νομίζω ότι είναι σημαντική αυτή η συζήτηση. Ε, που, από την ομάδα της Γοέ ο κύριος Μάρτιν Σίρντεβαν. Ε, ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Σε προηγούμενη συζήτηση έχω ξαναπεί για το θέμα αυτό ότι η αριστερά έχει ως κέντρο βάρους της τα εξή δύο και είναι πολιτικά τα ζητήματα αυτά. Πρώτον, τα ε, συμφέροντα των εργαζομένων να προστατεύονται και δεύτερον, να ε, αποκλείονται οι πρακτικές φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής. Γι' αυτό εκφράσαμε και κάποια κριτική και στην πρόταση οδηγίας Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπάρχουν κάποια σημεία που δεν είναι αρκετά σαφή η διατύπωση και χωράει και βελτίωση. Και έχει γίνει μεγάλη βελτίωση στη γνωμοδότηση και ευχαριστούμε τον κύριο Λουτβίξον, <coughs> αλλά υπάρχουν ακόμα μια σειρά από τροπολογίες που κάναμε και θέλω να επικεντρωθώ σε αυτές. Το έχουμε συζητήσει και με τον εισηγητή και με τους άλλους συναδέλφους και ψάχνουμε συμβιβασμούς. Πρώτον, για μας έχει σημασία ε, ορισμός για τις τεχνητές, ε, τα κατασκευάσματα αυτά. Να υπάρχουν κριτήρια που να ορίζουν την πραγματική οικονομική δραστηριότητα για να μην έχουμε φοροδιαφυγή και να προστατεύονται τα συμφέροντα των εργαζομένων, ανδρών και γυναικών και να επιβάλλονται. Δεύτερο, πάρα πολύ κομβικό για μας είναι η συναπόφαση, η συμμετοχή στις αποφάσεις των εργαζομένων. Έχουμε τροπολογίες που ζητούμε ε, νέα διαπραγμάτευση όταν ξεπεραστούν κάποιες οριακές τιμές που υπάρχουν στα κράτη και ζητούμε και ε, με μετενέργεια της προστασίας των εργαζομένων. Ιδιαίτερα σε περίπτωση συγχωνεύσεων και διαιρέσεων στην πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, υπάρχουν παραθυράκια και χωράνε παρερμηνίες και στρεφλές εφαρμογές. Και το τρίτο έχει να κάνει με ενίσχυση της θέσης των εμπειρογνωμόνων ή της αρμόδιας αρχής για τον έλεγχο, κατά πόσο η μετεγκατάσταση ή διαίρεση χρησιμοποιείται για καταχρήσεις και ελαφροχειρίες. Ελπίζουμε να είναι επικοδομητική η συζήτηση και να καταλήξουμε σε συμβιβασμούς. Είμαι πολύ αισιόδοξο. Παραμένουμε ε, σε επικοδομητικό πνεύμα συνεργασίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, η Πρόεδρος. Δεν έχουμε άλλες ομάδες παρούσες που να θέλουν το λόγο. Όχι. Άλλοι συνάδελφοι. Μα σκιώδεις όχι. Θα ξαναδώσω το λόγο στον εισηγητή μας, Όλε Λούντβικσον. Τόσο μικροφόνο δυστυχώς. I can understand that you understand Swedish. Ε, καταλαβαίνω, καταλαβαίνετε σουηδικά, δεν είναι πρόβλημα, καταλαβαίνετε σουηδικά. Να ξεκινήσω από την αρχή. Θα ήθελα ξεκινώντα να ευχαριστήσω όλου του συναδέλφου που πήραν το λόγο. όπω έλεγα προηγουμένω, αναμφισβήτητα υπάρχουν αποκλίνουσες απόψει, απόψει που υπάρχουν για διάφορα ζητήματα. Και είναι το θέμα κυρίω των όρων, των συνθήκων που σχετίζονται με αυτά, αυτές τις τεχνικές μεταρρυθμίσεις όσον αφορά το τι γίνεται σε δυσυνορικό επίπεδο αυτή είναι η πρόκληση που θα έχουμε εν συνεχεία. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε επί ενός σημείου. Θέλουμε να αποφύγουμε κάθε κατάχρηση. Θέλουμε να αποφύγουμε τη δημιουργία περισσότερων ε, εταιριών ε, εικονικών γραμματοκιβωτίου. Θέλουμε μεγαλύτερη ασφάλεια για όλους. Το ερώτημα που δημιουργείται είναι το εξής. Πώς να τα καταφέρουμε. Πώς θα καταφέρουμε να το πετύχουμε. Λάβαμε πάρα πολλέ τροπολογίε. Είναι προφανέ ότι πρέπει να συνεχίσουμε τι συζητήσει μεταξύ μα προσπαθώντα να βρούμε συμβιβαστικέ ε, λύσει. Ολοκληρώνοντα, θέλω να πω ότι θα είμαι πολύ ευτυχή να συναντηθώ με του σκιώδει εισηγητέ ήδη από αύριο να τα πούμε, διότι αύριο γίνεται η συνεδρίαση των σκιωδών εισηγητών. Σίγουρα θα διεξαχθούν άκρως επικοδομητικές συζητήσεις οι οποίες θα μας επιτρέψουν να καταλήξουμε σε μια καλή ψηφοφορία στην Επιτροπή. Ελπίζω να είμαστε όλοι ευέλικτοι. Εν πάση περιπτώσει πιστεύω ότι είναι σημαντικότατο να συνεργαστούμε αποτελεσματικά για να βρούμε μια αποτελεσματική επίσης λύση. Ε, αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι να βρούμε τι λύσει που είναι επαρκεί και υλοποιήσιμε. Ιδού, για μια ακόμη φορά ευχαριστώ όλου και ελπίζω θα καταλήξουμε σε καλή συνεργασία από αύριο για να βρούμε μια καλή λύση. Σα ευχαριστώ όλους. Τέλεια. Θα πρέπει να δουλέψετε καλά και σκληρά, αλλιώ δεν θα προλάβουμε να ψηφίσουμε στι 18 Οκτώβρη. Γιατί έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για να λάβουν υπόψη στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων το θέμα μας. Λοιπόν, η Γιούρη θα ψηφίσει στις 20 Νοεμβρίου, την αρμόδια επί της ουσίας. Ερχόμαστε λοιπόν τώρα στο επόμενο θέμα, το τελευταίο για σήμερα, το σημείο 11. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι γνωμοδότηση, επί της ουσίας είναι αρμόδια η Επιτροπή Προϋπολογισμών. Με εισηγητή εκεί τον κύριο Λεβαντόφσκι. Στη δική μας Επιτροπή συντάκτης γνωμοδότηση είναι ο Ραμόν Χάουρεγγι. Του δίνω μέσω στο λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στα γαλλικά και στα ισπανικά. Πάρα πολύ σύντομα θέλω να πω τα συνεργαστήκαμε με τους σκιώδεις των διαφόρων πολιτικών ομάδων με στόχο να συντάξουμε αυτή τη γνωμοδότηση, όπως είπατε, από την ΕΚΟΝ προς την Επιτροπή Προεπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας για την έκθεση αυτή. Ποιο είναι το σημαντικότερο για, την, για μένα, για την Επιτροπή μας η ΕΚΟΝ θα πρέπει να διαβεβάσει στην Επιτροπή Προεπολογισμών την ανάγκη να είμαστε πιο φιλόδοξοι στην πρόταση που εξετάζουν το Συμβούλιο και η Επιτροπή. Από εκεί πρέπει να ξεκινήσω. Πιστεύω ότι είναι κοινή αντίληψη εδώ στην ΕΚΟΝ. Αυτό. Φιλοδοξούν Συμβούλιο και Επιτροπή να βάλουν στους ιδίους πόρους τρία μικρά φορολογικά έσοδα αυτό είναι πολύ χαμηλή ως φιλοδοξία. Σε αυτό καταλήξαμε. Γιατί όπως γνωρίζετε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκέφτεται και εξετάζει μαζί με το Συμβούλιο μόνο τη δυνατότητα να ενταχθούν ως ήδη οι κάποια μικρά ποσοστά της ε, κοινή ε, ενοποιημένης φορολογικής βάσης για τις επιχειρήσεις, το CCCTB, όταν τεθεί σε ισχύ και φοβούμε πάρα πολύ γιατί χρειάζεται ομοφωνία για αυτό το θέμα. Οπότε θα πάρει χρόνο. Μετά προτείνει ένα μικρό κλάσμα των εσόδων από τους σπόρους που έχουμε από την εμπορία εκπομπορήπων και επίσης κάτι λίγα από τα πλαστικά μη ανακυκλούμενα. Μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξυγχρονίζει τώρα τους ιδίους πόρους σε σχέση με τους ισχύοντες, αλλά έχω την αίσθηση ότι θα έχουμε ένα χρηματοδοτικό σύστημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με πολύ λίγους ιδίους πόρους. Θα συνεχίσουμε να το έχουμε αυτό και είναι αντίθετο με την ιδέα που έχουμε και εκφράζουμε όλες οι πολιτικές ομάδες κάθε φορά στο PDP ή στον ετήσιο προπολογισμό της Ένωσης. Για τον λόγο αυτό οι διάφορες πολιτικές ομάδες έχουν κάνει πολλές τροπολογίες για να ενταχθούν νέοι φόροι. Ο κύριος Παπαδημούλης, ας πούμε, εξ ονόματος της ΓΚΟΕ και άλλοι εκπρόσωποι των Πρασίνων κλπ. Και φυσικά και η δική μας ομάδα, σοσιαλιστές και δημοκράτες, κάναμε μια σειρά από προτάσεις. Ε, συμβιβαστική πρόταση στην οποία καταλήξαμε ποια είναι. Να βάλουμε τέσσερις φόρους με τους οποίους συμφωνούμε όλοι. Και είναι σημαντικό επίτευγμα αυτό κατά την άποψή μου. Σας προτείνω λοιπόν το συμβιβασμό αυτό, με την επιφύλαξη βέβαια κάθε πολιτική ομάδα να ψηφίσει και τις δικές της τροπολογίες ως συμπροματικές της συμβιβαστική. Συμβαστική α λοιπόν περιλαμβάνει τα εξής. Ήδη οι πόροι θα πρέπει να είναι φόρος επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών που το έχουμε συζητήσει, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας, επίσης τα πρόστιμα του δικαστηρίου και ένας μηχανισμός προσαρμογής στην ε, εισαγωγή προϊόντων που ε, στην παραγωγή τους εκπέμπεται πολύ διοξίδιο του άνθρακα. Και ένα τέταρτο έχει να κάνει με τα έσοδα και τα κέρδη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ε, από το ευρώ. Αυτό συνδέεται με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και τη σταθερότητα. Και ε, όλα αυτά δεν χρειάζονται αλλαγή των συνθήκων, είναι με κείμενες συνθήκες. Διαπραγματευόμαστε τώρα για να φέρουμε αύριο ένα συνενετικό κείμενο γύρω από αυτό το συμβασμό που σας ε, προτείνω. Αυτά είναι τα σημαντικότερα. Υπάρχουν και άλλες τροπολογίες, Πρόεδρε, που έχουν να κάνουν με την ανάγκη στο να αναφέρονται οι οδηγίες, τα συμπεράσματα της ομάδας υψηλού επίπεδου, του πρώην Επιτρόπου Μόντι, θυμάστε, ε, ε, αυτό μας οδήγησε και στη σημερινή έκθεση. Επίσης, να ζητήσουμε το Κοινοβούλιο να έχει ένα πιο σημαντικό ρόλο. Αυτό μπορεί να θεωρηθεί και τελειτουργικό, το ζητάμε πεφάγια, Για το Συμβούλιο μπορεί να χρησιμοποιήσει τις λεγόμενες ρήτρες πασαρέλας για να μην εξαρτάται από την ομοφωνία και μετά να καταργήσουμε τις εθνικές διορθώσεις με την ευκαιρία του Brexit. Δηλαδή αυτή τη στιγμή το Ηνωμένο Βασίλειο να τερματιστούν οι διάφορες διορθώσεις και επιστροφές και επιταγές που δινόντουσαν για να επιστραφούν στο Ηνωμένο Βασίλειο τα χρήματα που ζητούσαν. Όλα αυτά δεν θα γίνουν απότομα και βία, αλλά παρόλα αυτά θα πρέπει να στείλουμε το μήνυμα ότι τώρα που φεύγει το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να τερματιστούν αυτά στα πλαίσια του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Αυτά, Πρόεδρε, αυτές είναι οι τροπολογίες και ελπίζω αύριο να συμφωνήσουμε με τους σκιώδες και να ψηφίσουμε στο αυριανό ψήφισμα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, Πολύ καλά. Η ψηφοφορία όμω είναι αύριο. Και διαπραγμα... ακόμα συμβαστικέ. Εκτό μικροφώνου η απάντηση. Θα μεταμορφώσουμε τη συνεδρίαση σε ένα είδο διαπραγματεύσεων. Αυτή είναι η λύση, ε. Και έτσι θα υπάρχει και πλήρης διαφάνεια. Για το ΕΛΚ ο Αλέων Λαμασούρ. Να το πω εκ των προμένων ότι είναι αρκετά αποφασισμένο ε, για κάποιες συμβαστικές. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ναι, εργαζόμαστε σε πραγματικό χρόνο. Είναι έξοχη δουλειά που γίνεται. Νομίζω ότι τα συμπεράσματα που σας προτείνουμε αύριο θα σας ικανοποιήσουν. Σε αυτό το πνεύμα εργαζόμαστε και βεβαίως θα ικανοποιήσουν και την πλειοψηφία των συναδέλφων, μη τι όλους. Δεν χρειάζεται να επενθυμίζω, το έκανε ο Ραμόν, πόσο σημαντικό είναι το θέμα. Η βασική επιτροπή είναι η Επιτροπή Προπολογισμών που έχει επιληφθεί. Έξι επιτροπές μεταξύ των οποίων και η δική μας η ΕΚΟΝ έχουν επιφορτιστεί με το να γνωμοδοτήσουν. Η ΕΚΟΝ ενδιαφέρεται για δύο λόγους. Από τη μία πλευρά, από τη στιγμή όπου ετοιμαζόμαστε τα επόμενα χρόνια και πρέπει να αντικατοπτρίζεται αυτό στο επόμενο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Να μεταφέρουμε ευθύνε, νέε ευθύνε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό θα πρέπει να βοηθήσει τα κράτη-μέλη να μειώσουν κάποιε από τι εθνικέ του δαπάνε. Αν γίνει μεταφορά φόρτου, θα γίνει μεταφορά δαπανών και ίσω και μεταφορά φόρων. Από την άλλη πλευρά είναι προφανέ ότι όσον αφορά τους νέους ιδίους πόρους, η Επιτροπή ΕΚΟΝ είναι αρμόδια όσον αφορά τα θέματα τα φορολογικά και είναι σημαντική η άποψή της. Όπως είπε και ο Ραμόν, να πω και εγώ ότι το Brexit θα έχει σαν αποτέλεσμα μείωση των πόρων του κοινοτικού προπολογισμού, διότι παρά την πολιτική της επιστροφής του rebate είναι καθαρός συνεισφορέας στον προπολογισμό του ΕΒ. θα πρέπει να βρούμε τη δυνατότητα αντιστάθμισης και πέραν αυτού λάβαμε υπόψη ότι πέρα από το Ηνωμένο Βασίλειο είχαμε άλλα πέντε κράτη-μέλη της Ενώσεως που έχουν επιστροφές, rebates. Κάποια από τα rebates υπολογίστηκαν βάσει του βρετανικού rebate, κάποια άλλα είναι συγκρίσιμα με το βρετανικό rebate. Και αυτό εξηγεί και ότι χρειαζόμαστε κάποιο χρόνο για να καταφέρουμε να πετύχουμε αποδεκτό συμβιβασμό αποδεκτό από όλους όσον αφορά το θέμα αυτό. Οι διαφορές είναι λιγότερο μεταξύ πολιτικών ομάδων από ότι είναι η εθνική καταγωγή των μελών της ε, Επιτροπής Οικονομικών Νομισματικών Θεμάτων. Καταλήξαμε σε κάποιους συμβιβασμούς, τουλάχιστον φορά το ΕΛΚ, που θεωρούμε ότι είναι ικανοποιητικέ. Υπάρχει ένα σημείο επί του οποίου θα προτείνουμε κατά τη διάρκεια της βραδιάς ένα κείμενο, τελικό κείμενο, επί ενός ε, θέματος που είναι η χρηματοδότηση δημοσιονομικής δυνατότητας για χρηματοδότηση πολιτικών ή των ιδίων πόρων της Ευρωζώνης. Ε, προσανατολιζόμαστε προς ένα κείμενο που θα αντιστοιχεί στο ευκταίο από εσά. Εξάλλου, αυτό συνάδει και με τη βούληση του ΕΛΚ οι προτάσεις που θα κάνουμε στην Οικονομική και Νομισματική Επιτροπή να εντάσσεται στα πλαίσια των ισιουσών συνθήκων και να μην προϋποθέτει τροποποίηση των συνθήκων. Όσον αφορά τα rebates, μετά από μακρά συζήτηση, προσανατολιζόμεθα προς πιο ευέλικτη λύση από ότι η άκρος άκαμπτη που είχα προτείνει μετά το high level group, δηλαδή ότι οι Βρετανοί δεν είναι εκεί. Αύριο βγάζουμε όλα τα rebates, κάποιοι συνάδελφοι ε, μέσω στοιχείων είπαν ότι θα ήταν θεματικές συνέπειες αυτού όσον αφορά την αύξηση των εθνικών συνεισφορών κάποιων χωρών. Γνωρίζοντας ότι εν λόγω χώρες δεν είναι πιο σημαντικές από άλλες. Όλος ο κόσμος είναι ισότιμος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά εν γέννη αυθόρμητα δεν έχουν την τάση να αυξήσουν όλες οι χώρες τη συνεισφορά στον εθνικό προϋπολογισμό. Οπότε πρέπει να μας διαπνεύσει ο ρεαλισμός και έτσι να αποδεχτούμε ένα σύστημα σταδιακό όπως αυτό που είχε προτείνει η ίδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτά με την επιφύλαξη κάποιων άλλων σημείων που είναι δευτερευούση σημασίας νομίζω ότι θα μπορέσουμε αύριο, όπως είπε και η θα μπορούσαμε να καταλήξουμε σε αρκετά ευρεία συνένεση πάνω σε αυτό το σημαντικό θέμα. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Από τους φιλελευθέρους. Λίβε. Αγαπητή κυρία Πρόεδρε, κύριε Σίγητα και αγαπητοί συναδελφοί, σας ευχαριστώ για την συνεργασία στο θέμα αυτό. Συνολικά συμφωνώ πως η Ένωση μας χρειάζεται περισσότερους ίδιους πόρους για να εξαρτάται λιγότερο από τις συνεισφορές των κρατών μελών. Μαζί έχουμε καταλήξει σε κάποιους συμβιβασμούς ε, που ελπίζω ότι θα βαρούν ευρεία στήριξη. Αν και δεν μπορούμε να εξαναγκάσουμε τα κράτη-μέλη να υιοθετήσουν την κοινή φορολογική βάση των επιχειρήσεων, σε μια νομοθετική πρόταση όπως αυτή θα ήθελα και πάλι να τονίσω ότι θα πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο. Επιπλέον δράτω με τις ευκαιρίες να ξεκαθαρίσω τέσσερις τροπολογίες μου που θεωρώ πολύ σημαντικές ε, και στις οποίες θα ήθελα την στήριξη σας. Είναι οι 87, 89, 90 και 92. Οι τροπολογίες αυτές δεν αυξάνουν τον προϋπολογισμό και διασφαλίσουν ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Απλά αφήνουν ανοιχτή την επιλογή ο προϋπολογισμός να είναι 100% από ίδιους πόρους ε, στην περίπτωση στην οποία οι πόροι που έχουμε αναφέρει δημιουργούν πολύ ψηλό εισόδημα. Οποιοδήποτε επιπρόσθετο ευρώ σε ίδιους πόρους θα αφαιρείται από την εθνική συνεισφορά. Αλλά δεν έχει νόημα να βάλουμε κάποιο όριο σε αυτό. Ελπίζω να στηρίξετε αυτή την ιδέα και να ψηφίσετε τις τροπολογίες 87, 89, 90 και 92. Ευχαριστώ. Μικρόφωνο η Πρόεδρος. Ε, βλέπω κανένα από τους πρασίνους. Από την Ενωτική Αριστερά, κ. Παπαδημούλης, παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή, τον κύριο Ραμόν Χαουρέγγι. Νομίζω ότι έχει κάνει μια σημαντική θετική δουλειά. Ε, είμαι ικανοποιημένο και για το επίπεδο συνεργασίας ανάμεσα στους κοιόδης εισηγητές. Ε, βλέπω αρκετές από τις τροπολογίες που κατέθεσα εκ μέρους πολιτικής μου ομάδας να έχουν γίνει δεκτές στην ουσία τους, όχι κατά λέξη, ε, στο, στα συμβιβαστικά κείμενα που ε, έχουν ετοιμαστεί. Με αυτό το πνεύμα θα συνεχίσουμε και σε ό,τι απομένει ακόμη. Ο στόχος είναι να εγκρίνουμε μια γνωμοδότηση με την ευρύτερη δυνατή συνένεση, η οποία όμως να είναι φιλόδοξη, να οθεί προς την κατεύθυνση που το Ευρωκοινοβούλιο εδώ και χρόνια πιέζει και επιδιώκει και να μην ε, πηγαίνει με το business as usual. Ο λόγος είναι προφανής. Μετά το Brexit, προκειμένου να μην έχουμε μεγάλες μειώσεις του κοινοτικού προϋπολογισμού, χρειάζεται επιτέλους να προχωρήσουμε στην υιοθέτηση της αύξησης των ιδίων πόρων με την υλοποίηση κάποιων προτάσεων που εδώ και χρόνια το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, έχει βάλει στο τραπέζι, όπως ο φόρος επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, έσοδα από τις εκπομπές του διοξιδίου του άνθρακος που βοηθούν και τα έσοδα του κοινοτικού προϋπολογισμού αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος, κέρδη από τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας διότι είναι έσοδα που παράγει η λειτουργία του ευρώ και του κοινού και άρα πρέπει να τροφοδοτούν τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Ε, να αξιοποιήσουμε την εργαλειοθήκη με άλλα λόγια των προτάσεων Μόντι ε, για την ανάγκη να ξανασκεφτούμε πιο φιλόδοξα το θέμα ε, των ε, ιδίων πόρων. Πιστεύω επίσης ότι θα πρέπει να επανεξετάσουμε αυτή την ανορθογραφία του rebate η οποία είναι μια κληρονομιά ε, μπαλώματος θεσμικού από την εποχή της Μάργαρετ Thatcher και η οποία δεν είναι ε, ότι το καλύτερο. Καταλαβαίνω τις δυσκολίες τις οποίες αναφέρθηκε και ο κύριος Λαμασούρ. Πρέπει να πάμε ενδεχομένως βήμα-βήμα και με ένα ε, συμβιβαστικό πνεύμα, αλλά ο στόχος είναι να εξαλείψουμε τελικά ως τελικό στόχο αυτές τις ανορθογραφίες για να υπάρχει ένα δίκαιο και διαφανές ε, σύστημα. Πιστεύω επίσης ότι ε, έχει αξία όχι μόνο οι ίδιοι οι πόροι να φτάσουν στο 25% του συνολικού ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, αλλά να δούμε και τις προτεραιότητες και για το πού θα πρέπει να κατευθυνθούν αυτοί οι πόροι. Νομίζω δηλαδή ότι στη συζήτηση που εκφεύγει δηλαδη οτι στη συζητηση που εκφευγει αυτή της γνωμοδότησης και που αφορά το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, πρέπει να δούμε πώς αυτοί οι πόροι θα αποδειχθούν χρήσιμοι ε, και αποδοτικοί για την ενίσχυση πολιτικών συνοχής, τη θωράκιση της απασχόλησης, την ενίσχυση των επενδύσεων, μια στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης, τη μείωση των ανισοτήτων κοινωνικών και περιφερειακών, διότι ε, μόνο έτσι μπορεί η Ευρώπη να γίνει καλύτερη ε, για τους ε, πολίτες. Ένα τελευταίο θέμα που ήθελα να τονίσω είναι η ανάγκη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διεκδικήσει πιο δυναμικά το θεσμικό ρόλο του, να μην ανέχεται πρακτικές που το παρακάμπτουν στο όνομα της ευελιξίας. Είναι μια πρακτική στην οποία μας έχουν συνηθίσει αρκετές φορές στο Συμβούλιο, που είναι ο κυρίως υπεύθυνο, αλλά καμιά φορά με την συμμετοχή και της Κομισιόν. Νομίζω ότι το Ευρωκοινοβούλιο και ιδιαίτερα λίγους μήνες πρώτων ευρωεκλογών πρέπει να απαιτήσει να έχει ουσιαστικό ρόλο στην ε, ε, πολιτική που τελικά θα αποφασιστεί για το θέμα των ιδίων πόρων. Σας ευχαριστώ. Ε, η πρόεδρος. Άλλος. Άλλη πολιτική ομάδα. Όχι. Άλλοι συνάδελφοι. Μεμονωμένοι ούτε να ξαναδώσω το λόγο στον εισηγητή. Είναι <laughs> ευτυχής ο εισηγητή και περιμένει τους τελικούς συμβιβασμού. Αν ήμουν συντάκτη νομοδότη, απαντούσα στον κύριο Παπαδημούλη ότι στι πολλέ τροπολογίε, ε, πολλέ έχουν συμπεριληφθεί στι συμβαστικέ και πολλέ βρίσκουν σύμφωνο τον εισηγητή. Αλλά εγώ δεν είμαι εισηγητρία για να τα πω αυτά. Ε, ε, κύριος Χάουρεγγι, ε, δεν έχω να προσθέσω τίποτα. Θα προσπαθήσουμε αύριο να ενημερώσουμε τις ομάδες για την τελική μας πρόταση. Τώρα είμαστε στο στάδιο της σύνταξης των τελικών κειμένων. Ζητώ συγγνώμη από όλους, αλλά οι ομάδες μας έφεραν σήμερα το απόγευμα τις προτάσεις τους. Γι' αυτό καθυστερήσαμε λίγο και σας ζητώ συγγνώμη απόψε ή αύριο το πρωί θα έχετε την ενημέρωση και θα ψηφίσουμε το απόγευμα έτσι καλώς. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Μάλιστα. Καλή επιτυχία και καλή δουλειά στις ομάδες διαπραγμάτευσης. Δεν ξέρω αν έχετε πολλές ώρες ή λιγότερο από μία ώρα. Τελειώσαμε. Ευχαριστούμε και τους διερμηνείς. Ραντεβού αύριο το πρωί στις 9 η ώρα.